Iniziamo. Ξεκινήσουμε παρακαλώ. Καλησπέρα σα. Α ξεκινήσουμε τι συνεδρίε τη Επιτροπή. Έχουμε πολύ πλούσια ημερησία διάταξη. Προχωρήσουμε λοιπόν γρήγορα. Σημείο 1. Έγκριση τη ημερησία διάταξη η ανταλλαγή απόψεων με τον Επίτροπο Τζόλος για τις συνέπειες ε, για τη Γεωργία την πρόταση της Κομισιόν για τις δημοσιονομικές προοπτικές είχε προβλεφθεί για τις 4 σήμερα το απόγευμα αλλά ο Επίτροπος μας ανακοίνωσε ότι θα έρθει εδώ στις 4.30 Γι' αυτό σας προτείνω αμέσως μετά το σημείο 4 να δούμε το επόμενο σημείο για να μπορέσουμε να μιλήσουμε, να συνομιλήσουμε με την Επίτροπο στο τέλος. Αν δεν υπάρχουν άλλες παρατηρήσεις εγκρίνεται η ημερησία διάταξη έγκριση των πρακτικών. Αν δεν υπήρχουν, υπάρχουν παρατηρήσεις πριν από το τέλος της συνεδρίασης, θα θεωρήσουμε ότι θα έχουν εγκριθεί και τα πρακτικά. Παρακαλώ. There's Γιατί δεν υπάρχει διερμηνία. Facciamo le verifiche. Για να επαληθεύσουμε. Funziona. Λειτουργεί το σύστημα. Υπάρχει διερμηνία στα γερμανικά, μάλιστα, πολύ ωραία. γαλλικά. Funziona. Prova ancora. Λοιπόν, λειτουργεί το σύστημα. It's number three Germany now. Λοιπόν, τα γερμανικά βγαίνουν στο κανάλι 3 τώρα. Εντάξει. Εντάξει. Possiamo proseguire? Μπορούμε να συνεχίσουμε. Germany doesn't work. No, they switch, they switch the channel. Provo a parlare per vedere se viene tradotto. Λοιπόν, εγώ θα μιλήσω για να δω αν υπάρχει διερμηνία. Είστε έτοιμοι για να πάτε για διακοπές. Πολύ ωραία. Τώρα εδώ κάνουμε κάποιες ασκήσεις διερμηνίας, λέει ο πρόεδρος λειτουργεί η διερμηνία στα γερμανικά. Πολύ ωραία. Ας προχωρήσουμε. Σας ευχαριστώ και συγγνώμη για το μικρό πρόβλημα. Λοιπόν, έλεγα για το σημείο 2, πρακτικά, αν δεν υπάρχουν παρατηρήσεις, θεωρούμε ότι εγκρίνονται. Και τώρα, προσοχή, γιατί θα σας δώσω ορισμένες πληροφορίες. Ήθελα να επισημάνω ότι η προθεσμία για την ε, κατάθεση των τροπολογιών στο σχέδιο προπολογισμού Κομισιών είναι 20 ε, Ιουλίου 2011 το μεσημέρι. Η Γραμματεία θα στείλει στα mail ένα ενημερωτικό σημείωμα για τη διαδικασία και τι τεχνικέ λεπτομέρειε. Λοιπόν, τροπολογίε για το σχέδιο προπολογισμού τη Κομισιόν 20 Ιουλίου στι 12 το μεσημέρι. Και τώρα επικαιροποίηση, ενημέρωση για τον τριμερή διάλογο. Να σας ενημερώσω ότι για τους δύο τριμερείς διαλόγου που έλαβαν χώρα για το θέμα της ευθυγράμμισης της αγροτικής ανάπτυξης και των άμεσων ε, ενισχύσεων 24 Μαΐου και 22 Ιουνίου με το Συμβουλίο υπό την Ουγγρική Προεδρία και την Κομισιόν. Ακόμη, και αν δεν έχουμε καταλήξει σε τελική συμφωνία, ε, έχουμε σημειώσει πρόοδο και στους δύο φακέλους. Στην πρόοδο για την αγροτική ανάπτυξη ε, εξετάστηκαν όλα τα σημεία και καταλήξαμε σε συμφωνία για τα λιγότερο ευαίσθητα σημεία. Όλα τα γλωσσικά θέματα διευκρινίστηκαν με τη βοήθεια των νομικών σε τεχνικές συνεδριάσεις σε διοικητικό επίπεδο. Και στα δύο θέματα υπάρχουν θέματα οριζόντιας φύσεως ε, που θα είναι σημαντικά και για τις υπόλοιπες εκθέσεις για την ευθυγράμμιση όπως το χάρη το θέμα των ελέγχων και των κυρώσεων. Στην περίπτωση αυτή το Συμβούλιο προχωρά με πλήρης τροποποίηση ενώ η Κομισιόν προτείνει κατεξουσιοδότηση πράξης. Το Συμβούλιο εν μέρη εντάσσει εφαρμοστικούς κανονισμούς, εκτελεστικούς κανονισμούς ε, της Κομισιόν στη βασική πράξη και για τα λοιπά προτείνει εκτελεστικές πράξεις. Ε, για μας ε, δεν είναι κατάλληλη αυτή η προσέγγιση για δύο λόγους. Καταρχήν, στην περίπτωση που χρειαστεί να γίνουν, να γίνουν τροποποιήσεις, μια ολόκληρη τακτική νομοθετική διαδικασία θα πρέπει να ξεκινήσει και αυτό σημαίνει φυσικά ότι θα έχουμε γραφειοκρατικό άχθος για θέματα ισονοσημασίας συνήθως. Δεύτερον, το Κοινοβούλιο θα αποκλειόταν από οποιοδήποτε έλεγχο στην τροποποίηση της νομοθεσίας. Σας υπενθυμίζω ότι έχει δικαίωμα βέτο το Κοινοβούλιο μόνο για τις κατεξουσιοδότηση πράξεις και όχι για τις εκτελεστικές πράξεις. Έτσι λοιπόν, κάθε φορά που το Συμβούλιο προτείνει το πέρασμα ε, σε εκτελεστική πράξη από κατεξουσιοδότηση πράξη, σημαίνει ότι το Κοινοβούλιο αποκλείεται ολοκληρωτικά. Ας το έχουμε αυτό κατά νου. Το Συμβούλιο μέχρι τώρα δεν έχει αλλάξει την προσέγγιση του, αλλά ελπίζουμε ότι η ομάδα των διαπραγματευτών του θα έχει εντολή για να προχωρήσει στο πρόβλημα αυτό. Θα να σημειώσει κάποια πρόοδο στις επόμενε συνεδριάσεις. Ε, συζητήσαμε για το θέμα αυτό με την Πολωνική Προεδρία και ελπίζουμε να σημειωθεί πρόοδος. Ένα άλλο οριζόντιο θέμα είναι η πρόταση του Συμβουλίου να χρησιμοποιηθεί το άρθρο 5 παράγραφος 4 του κανονισμού για τις εκτελεστικές πράξεις, σύμφωνα με το οποίο η Κομισιόν δεν μπορεί να δράσει αν ε, η αρμόδια επιτροπή δεν γνωμοδοτήσει. Στην περίπτωση αυτή δεν συμφωνούμε με το Συμβούλιο, γιατί αυτό θα σήμαινε ότι εισάγεται εξαίρεση στις δύο οργανικές ε, συμφωνίες σε ό,τι αφορά το φάκελο των άμεσων ενισχύσεων, το πιο σημαντικό θέμα για το Κοινοβουλίο είναι το άρθρο 11 για την εφαρμογή της ε, δημοσιονομικής πειθαρχίας. Εδώ είχαμε κάθετες θέσεις σε αυτή την Επιτροπή, υπενθυμίζω την εμπλοκή μας στη διαδικασία, καθώς ε, έχουμε και τις νέες νομοθετικές ονοδιότητες και σε ό,τι αφορά και τον προϋπολογισμό. Το Κοινοβούλιο λοιπόν έχει αποκλειστική αρμοδιότητα ή τουλάχιστον σημαντικό ρόλο. Η θετική πλευρά είναι ότι η Κομισιόν που αρχικά ήταν κατά της θέσης του Κοινοβουλίου μας δήλωσε ότι είναι ανοιχτή τώρα στα δικά μας επιχειρήματα και θα παρουσιάσει πιθανότατα τις επόμενες εβδομάδες μία πρόταση για το θέμα αυτό. Και τέλος, σύμφωνα με τη γενική προσέγγιση του Κοινοβουλίου, προσπαθήσαμε να επρασπίσουμε τη χρήση όπου είναι δυνατόν των κατεξουσιοδότηση πράξεων, στην περίπτωση όπου θα μπορούσαν να απειλούνται τα δικαιώματα των αγροτών. Δηλαδή, όταν πρόκειται για δικαιώματα των αγροτών, δεν μπορούμε παρά να προβλέψουμε κατεξουσιοδότηση πράξης, όπου η εμπλοκή του Κοινοβουλίου είναι πλήρης και όχι εκτελεστικές πράξεις που επαναλαμβάνω αποκλείουν το Κοινοβούλιο. Σε ό,τι αφορά τώρα τη χρήση των κατεξουσιώτηση πράξεων για τροποποίηση των παραρτημάτων, η Κομισιόν δέχτηκε τα επιχειρήματα της δικής μας νομικής υπηρεσίας. Έτσι λοιπόν, για το σημείο αυτό, εγώ σας καλώ, συνάδελφοι, όχι μόνο για αυτά τα θέματα των ε, εκτελεστικών ε, πράξεων, αλλά και για ε, τους επόμενους φακέλους που θα έρθουν στο μέλλον, να ε, βάζετε στις τροπολογίες που παρουσιάζετε θέματα ουσίας που αφορούν το έργο της ε, δικής μας Επιτροπής. Φυσικά ο κάθε βουλευτής έχει την ελευθερία να προτείνει οποιαδήποτε τροπολογία, όμως εγώ σας καλώ οι τροπολογίες προτείνετε να αφορούν ακριβώς τα θέματα στα οποία αναφέρθηκαν πριν, δηλαδή κατεξουσιοδότηση πράξης και εκτελεστικές πράξεις, γιατί στην περίπτωση αυτή η δουλειά που κάνουμε κυρίως στους τρεις πρώτους φακέλους αγροτική ανάπτυξη, άμεσης ενισχύσεις ε, και ενιακόα. Προσπαθούμε να υπερασπίσουμε εκεί τα δικαιώματα του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου και τις αρμοδιότητές του και να διατηρήσουμε όσο το δυνατόν περισσότερο τις ε, πράξεις κατά εξουσιοδότηση παρά να έχουμε εκτελεστικές πράξεις. Έτσι λοιπόν Τροπολογία από την πλευρά των συναδέλφων Πολλέ φορέ ε, φαίνεται να υπαγορεύονται από το Συμβούλιο, από τι εθνικέ αντιπροσωπείε. Κάτι τέτοιο αποδυναμώνει προφανώ ε, τη θέση που προσπαθούμε εμεί να παρουσιάσουμε και να προωθήσουμε κατά τη διάρκεια των τριμερών διαλόγων. Και ελπίζουμε ότι την Πολωνική Προεδρία θα συνεχίσουμε τον τριμερή διάλογο με την Πολωνική Προεδρία για μια ενδεχόμενη συνολική συμφωνία. Λοιπόν, αν υπάρχουν συνάδελφοι που θέλουν το λόγο για τα θέματα αυτά, παρακαλώ, παρακαλώ, Τζόρτζ, έχεις το λόγο. Yeah, be very brief Θα είμαι πάρα πολύ σύντομος, Πρόεδρε, να συμφωνήσω με αυτά τα οποία είπατε για τη συζήτηση μεταξύ ημών και του Συμβουλίου για πράξεις κατευσιοδότηση και τα σχετικά μέτρα. Είναι μια συζήτηση οριζόντια για όλες τις διαπραγματεύσεις που εξελίσσονται αυτή τη στιγμή. Και ε, ίσως ε, αύριο να αναγκαστούμε να ψηφίσουμε τροπολογίες που είναι η θέση του Συμβουλίου και όχι του Κοινοβουλίου. Ελπίζω λοιπόν να μπορέσουμε να μην είμαστε σε αυτή τη θέση αύριο ε, ή δυνατόν και η Επιτροπή Γεωργίας υποστηρίζει τις απόψεις που έχουν ήδη εκφραστεί για τις ε, διαδικασίες ε, αγροτικής ανάπτυξης και της κοινή οργάνωσης αγοράς, πώς εμείς θα πρέπει δηλαδή να έχουμε ως τον εδώ μεγαλύτερο λόγο στις ε, μελλοντικέ αποφάσεις για τα πάρα πολύ σημαντικά αυτά μέτρα για τους ψηφοφόρους μας που μας ψήφισαν ακριβώς για να υπερασπιστούμε τα συμφέροντά τους δεν έχει νόημα να αλλάξει ο κανόνα και να λέμε δεν ξέρει τι γίνεται το κοινοβούλιο. Πρέπει να δώσουμε αυτόν τον αγώνα σήμερα και του ερχόμενου μήνε και ελπίζω η Επιτροπή να σα ε, στηρίξει, εσά που είστε εισηγητή και του άλλου ε, εισηγητέ σε άλλε εκθέσει. Ευχαριστώ. Ε, Ευχαριστώ, George. Λοιπόν, ακριβώ αυτό είναι ο λόγο που όφησε όλου ε, του συντονιστέ ε, των ομάδων να εμπιστευτούν στον πρόεδρο τι πρώτε τρει εκθέσει. Γιατί σε ό,τι αφορά αυτά τα οριζόντια θέματα, πρέπει να ακολουθήσουμε μία ενιαία κατεύθυνση. Πρέπει να υπάρχει συνέπεια έναντι στα υπόλοιπα όργανα. Έτσι λοιπόν, εγώ ελπίζω να προχωρήσουμε καλά στις εργασίες μας και αν δεν υπάρχουν άλλες παρεμβάσεις, περάσουμε στο σημείο 4, υγεία των μέλισσών και προκλήσεις για το μελισσοκομικό τομέα. Εισηγητής ε, Τσάμπα Σάντορ Ταμπάτζη και ας περάσουμε στην εξέταση αυτή τη σημαντική γνωμοδότηση πρωτοβουλία για την υγεία των μελισσών και τι προκλήσει για τη γεωργία. Όπω ξέρετε, το μεγαλύτερο ε, μέρος των καλλιεργιών χρειάζονται τα έντομα για την επικονίαση και η επικονίαση γίνεται μέσω ε, της υποστήριξης αυτών των πολύ σημαντικών εντόμων των μελισσών ε, λόγω της διάδοσης των νόσων και των πρασίδων και, της, και των κλιματικών αλλαγών μειώνονται οι επικές των μελισσών στην Ευρώπη. Ο εισηγητής μας προτείνει δράση σε ευρωπαϊκό επίπεδο για να αντιμετωπιστούν οι ανησυχίες και τα προβλήματα των μελισσοκόμων στα περισσότερα τι μελη Θα δώσω λοιπόν τώρα το λόγο στον Μισημητή και νομίζω ότι είναι εδώ και ο πρόσωπος της Κομισιόν παρόν, ο Διευθυντής Μπερνόρη από τη ΓΑΜΑ ΔΕΛΤΑ ΣΑΝΚΟ και Νιούμαν από τη ΓΑΜΑ ΔΕΛΤΑ Άγκρη. Παρακαλώ, κύριε Σιγητά, έχετε το λόγο. Ευχαριστώ κύριε Πρόεδρε. Ήδη θέσατε τους βασικούς άξονες αυτού του προβλήματος. Το Νοέμβριο το Ευρωπαϊκό Κοινοβούλιο ενέκρινε ένα ψήφισμα και το Δεκέμβριο η Ευρωπαϊκή Επιτροπή υπέβαλε ένα διεξοδικό κείμενο. Ε, λάβαμε και την ανακοίνωση του Συμβουλίου και τώρα συντάξαμε ένα ψήφισμα που ουσιαστικά αντιδράσει όλα αυτά τα έγγραφα και υποβάλλει και κάποιες προτάσεις συγκεκριμένες προτάσεις για να καταπολεμήσουμε την κρίση στον μελισσοκομικό κλάδο. Ο μελισσοκομικός κλάδος, όπως είπε και ο πρόεδρος, δεν περιορίζεται στην παραγωγή μελιού μόνο. Απασχολεί περίπου 600.000 άτομα στην Ευρώπη η μελισσοκομεία και επίσης διαδραματίζει σημαντικό ρόλο στην επικονίαση. Οι μέλισσες χάρη στην επικονίαση ε, βοηθούν στον πολλαπλασιασμό 84% των φυτικών ειδών και 60% της παραγωγής τροφίμων εξαρτάται από αυτή την επικονίαση των μελισσών. Θα πρέπει και αυτό να το έχουμε υπόψη όταν ασχολούμαστε με την μελισσοκομεία. Θα πρέπει να υποστηρίξουμε αυτόν τον κλάδο, γιατί όπως σας είπα παίζει σημαντικό ρόλο και στα περιβαλλοντικά ζητήματα. Ξεπερνώντας την απλή παραγωγή μελιού. Πολλοί είναι οι λόγοι της τρέχουσας κρίσης. Κύριε Πρόεδρε, αναφερθήκατε σε πολλούς παθογονούς παράγοντες. Είπατε ότι Η μιλισοκομεία είναι ο λιγότερο ε, επαγγελματικό κλάδο τη κτηνοτροφίας ε, και το 90% των μιλισοκόμων σχεδόν είναι ερασιτέχνες. Επίσης, ε, υπάρχει πρόβλημα με τη χρήση φυτοφαρμάκων, με κάποιους φυτογενομικούς μηχανισμούς. Mm. Θα πρέπει να δούμε να προωθήσουμε μάλλον την έρευνα σε νέα προϊόντα για να καταπολεμήσουμε τα διάφορα παράσιτα και να επενδύσουμε και στην δημιουργία νέων φαρμάκων. Δυστυχώς οι μεγάλες φαρμακοβιομηχανίες δεν ενδιαφέρονται να επενδύσουν στην έρευνα φαρμάκων για τη μελισσοκομεία γιατί δεν είναι αποδοτικές επενδύσεις εκεί. Αν δεν υποστηρίξουμε κοινοτικά κονδύλια αυτό το κλάδο, δεν θα μπορέσει από μόνος του ο μελισσοκομικός κλάδος να επιλύσει το πρόβλημα. Η κυρία Λούλινγκ και ο κύριος Νίκολσον είπαν ότι πάει μία εικοσαετία που ασχολούμαστε με το θέμα αυτό και ακόμη δεν το έχουμε ρυθμίσει. Και το γεγονό ότι έχει μείνει ανεπίλητο αυτό το πρόβλημα οφείλεται στο ότι δεν αφιερώνουμε επαρκεί πόρου ε, στην έρευνα. Δεν υπάρχει αρκετή ε, παραγωγή, ανάπτυξη των προϊόντων που χρειαζόμαστε γιατί για τις ανθρώπινες νόσους έχουμε συνέχεια νέα αντιβιωτικά και φάρμακα, αλλά δεν ισχύει το ίδιο και για τις νόσους των μελισσών. Γι' αυτό η κατάσταση παραμένει αμετάβλητη. Σε ό,τι αφορά τη βαροϊκή ακαρίαση, πρόκειται για μία νόσο που οφείλεται σε ένα ακαριό που δημιουργεί πολλά προβλήματα, αλλά δυστυχώς δεν υπάρχει φάρμακο κατάλληλο για την αντιμετώπιση αυτής της ε, βαροϊκής ακαρίασης. Έχουν εντοπιστεί 11 δραστικές ουσίες, αλλά δεν έχουμε βρει ένα κατάλληλο φάρμακο. Στα πλαίσια του ερευνητικού προγράμματος πλαισίου θα μπορούσαμε να χρηματοδοτήσουμε την έρευνα για φάρμακα για την καταπολέμηση αυτής της νόσου, γιατί δεν κινδυνεύει μόνο η λησοκομεία αλλά και η κτηνοτροφία υπέβαλ, και η γεωργία. Υπέβαλα 30 περίπου προτάσεις. Χρειαζόμαστε καλύτερο monitoring, καλύτερη παρακολούθηση που δεν υπάρχει αυτή τη στιγμή στην Ευρώπη. Φυσικά οι μέλησες ε, δεν καταλαβαίνουν σύνορα, εθνικά σύνορα, γι' αυτό χρειαζόμαστε ένα καταξοχήν ε, υπερεθνικό, πανευρωπαϊκό σύστημα και φυσικά ένα συντονισμό μεταξύ των κρατών μελών. Είναι πολύ θετικό που αναφέρθηκε το θέμα των σημείων αναφοράς ε, γιατί χρειαζόμαστε εκτός από τα εργαστήρια που κάνουν διαγνώσεις και εργαστήρια που θα κάνουν έρευνες επιτόπου. Και επίσης θα πρέπει να χρησιμοποιήσουμε τα προγράμματα όπως COST, COLOS, BDOC και STEP. Αυτά έδωσαν καρπούς και θα πρέπει να τα αξιοποιήσουμε. Ε, τα διάφορα αισθήματα ελέγχου των καλλιεργιών είναι πολύ σημαντικά. Αυτή τη στιγμή δεν έχουμε αρκετά στοιχεία σαφή και συγκρίσιμα στην Ευρώπη για να δούμε ποια είναι ακριβώς η εικόνα της υγείας των μελισσών. Η ανταλλαγή πληροφοριών μεταξύ των εθνικών εργαστηρίων δεν είναι επαρκής. Όπως σας είπα, το 90% των μελισσοκόμων είναι ουσιαστικά ερασιτέχνες. Είναι ο λιγότερο επαγγελματοποιημένος κλάδος της κτηνοτροφίας η μελισσοκομεία. Και μάλιστα για να γίνει κανείς μελισσοκόμος δεν χρειάζεται καν ειδική κατάρτιση. Θα πρέπει όμως να προβλέψουμε κάποιο είδους πιστοποίηση που ισχύει για τους αλείς, για άλλα επαγγέλματα και γι' αυτό χρειάζεται χρημα... χρηματική υποστήριξη της Ευρωπαϊκής Ένωσης να χρηματοδοτήσουμε την κατάρτιση των μελισσοκόμων. Ούτε και οι κτηνίατροι δεν γνωρίζουν συγκεκριμένα τα ειδικά προβλήματα της υγείας των μελισσών. Χρειαζόμαστε λοιπόν φάρμακα, κτηνιατρικά προϊόντα και κονδύλια για να γίνει πιο ελαστικό το σύστημα και να αναπτυχθεί περαιτέρω. Επίσης κάποια κτηνιατρικά προϊόντα φυτικής προέλευσης χρησιμοποιούνται μεν, αλλά τίθενται σε εμπορία με πολύ αργούς ρυθμούς. Θα πρέπει να προωθήσουμε τέτοια φυτικά φάρμακα και να επιταχύνουμε τους ελέγχους και να είμαστε και πιο επικοδομητικοί για το μελισσοκομικό κλάδο προασπίζοντας καλύτερα και την πνευματική ιδιοκτησία για τα προϊόντα αυτά. Γιατί σήμερα, αν κάποιος ερευνητής ή ένα ερευνητικό κέντρο εφεύρει ένα νέο προϊόν, δεν, προστατεύεται παρκώς, δεν προστατεύονται παρκώς τα πνευματικά δικαιώματά του για το προϊόν αυτό. Αν θέλουμε λοιπόν ένα εξυγχρονισμένο γεωργικό κλάδο, θα πρέπει να επενδύσουμε και στη μελισσοκομεία. Ε, δώρος γίνεται για την επιρροή των φυτοφαρμάκων στην υγεία των ε, μελισσών. Βέβαια, η γεωργία χρησιμοποιεί φυτοφάρμακα, αλλά τουλάχιστον θα πρέπει να περιορίσουμε την ποσότητά τους. Τα φυτοφάρμακα ε, μας υποχρεώνουν ε, σε συγκεκριμένη μελέτη για την επιρροή τους ε, στην υγεία των μελισσών. Δηλαδή, θα πρέπει να βρούμε ποιε είναι οι δραστικές ουσίε που περιέχονται στα φυτοφάρμακα αυτά και πώς αυτές επηρεάζουν την υγεία των μελισσών. Γιατί θα μπορούσαμε κάλλιστα να αντικαταστήσουμε ορισμένε δραστικές ουσίε από άλλε που είναι λιγότερο επιβλαβείς για τις μέλισσες. Ενώ θα είναι εξίσου αποτελεσματικές ό,τι αφορά τη φυτογενομική του δράση. Πολύ λόγο. γίνεται και για την ε, υποχρέωση των γεωργών να ενημερώνουν τους ε, ε, μελισσοκόμους που βρίσκονται στην περιοχή τους για την χρήση κάποιων προϊόντων πριν ε, χρησιμοποιηθούν ένα αέρι ψεκασμοί, για παράδειγμα, κατά των, ζυζάνι, κατά των παρασίτων ή κουνουπιών. Αυτή τη στιγμή, επαναλαμβάνω, δεν υπάρχει καμία επιστημονική έρευνα και για τα αποτελέσματα των γενετικώ τροποποιημένων οργανισμών στην υγεία των ε, μελισσών. Δεν υπάρχουν ούτε θετικέ μελέτε, ούτε θε... μελέτε με θετικά αποτελέσματα, ούτε με αρνητικά. Και από αυτή την άποψη χρειαζόμαστε κάποιε αντικειμενικέ επιστημονικέ μελέτε για να δούμε αν υπάρχει κάποιο σχετισμό μεταξύ των ε, γενετικώ τροποποιημένων οργανισμών και των επιπτώσεων που έχουν στην υγεία των μελισσών. Σε ό,τι αφορά την επισητιστική ασφάλεια, πολύ συχνά εισάγουμε προϊόντα από τρίτες χώρες. Γίνονται έλεγχοι, αλλά δεν είναι αρκετοί. Θα μπορούσαμε ε, για ορισμένες περιπτώσεις ακόμη και να απαγορεύσουμε τις ορισμένες εισαγωγές. Βέβαια, με μια ολοσχερή απαγόρευση, μάλλον θα ενισχύσουμε το λαθρεμπόριο. Η οδηγία έχει κάποια καλά στοιχεία, αλλά ο ρυθμός εφαρμογής της είναι πολύ αργός παράμετροι ποιότητας του μελιού θα πρέπει να διευκρινιστούν περαιτέρω. Γιατί υπάρχει κάποια σάφια στο σημείο αυτό. Και στο σημείο 25 προτείνω διάφορα στοιχεία, δεν θα σας τα διαβάσω, αλλά ζητώ καλύτερη διευκρίνηση ορισμένων διατάξεων για να μπορούμε να εκτιμούμε καλύτερα την ποιότητα του μελιού και να καταπολεμήσουμε την ανώθευση του ή την αλλίωση του μελιού σε ό,τι αφορά την ε, χώρα προέλευσης. Εξετάζουμε στα πλαίσια της ε, σήμανσης των προϊόντων αν ε, πρέπει να είναι υποχρεωτική η της χώρας προέλευσης. Στην οδηγία για το μέλι γίνεται διάκριση μεταξύ τριών κατηγοριών. Το μέλι Ευρωπαϊκής Ένωσης, μείγμα μελιού ευρωπαϊκού και εξοκοινοτικού μελιού και τρίτη κατηγορία είναι μέλη εκτό Ευρωπαϊκή Ευρωπαϊκής Ένωσης. Αυτό όμω είναι πολύ γενικό, θα πρέπει να αναφέρουμε ρητά τη χώρα προέλευση, συγκεκριμένη χώρα προέλευση του προϊόντο. Στην αναθεώρηση της οδηγίας για τη σήμανση των τροφίμων θέλουμε να διαβρύνουμε την υποχρέωση μιας χώρας προέλευσης ε, σε πολλά προϊόντα και ένα από αυτά είναι και το μέλι. Γι' αυτό όμως θα πρέπει να αναθεωρήσουμε και την οδηγία για το μέλι. Θα θέλαμε η Ευρωπαϊκή Επιτροπή στην πρόταση αναθεώρηση που θα υποβάλει να λάβει υπόψη και αυτό το στοιχείο. Σε ό,τι αφορά την πολιτική ποιότητας, ένα από τα σημαντικά σημεία είναι το θέμα των ε, γεωγραφικών ενδείξεων, προστατευμένων γεωγραφικών ενδείξεων ή προστατευμένων ε, ε, αναφορών προέλευσης. Δεν χρησιμοποιούνται πάντα αυτές οι διατάξεις. Η Γαλλία και άλλες χώρες χρησιμοποιούν αυτές τις ονομασίες προέλευσης για να προστατεύσουν διάφορα προϊόντα, αλλά για το μέλι μόνο σε 14 μέλια από όλη την Ευρωπαϊκή Ένωση χρησιμοποιείται η ονομασία προέλευσης. Θα πρέπει λοιπόν να προσφύγουμε περισσότερο στη χρήση της ονομασίας προέλευσης για να προασπίσουμε την ποιότητα του μελιού. Ας μην ξεχνούμε και την ανάπτυξη της υπαίθρου εδώ. Για παράδειγμα, θα μπορούσαμε να ε, δώσουμε έμφαση σε συγκεκριμένες καλλιέργειες, καλλιέργειες ψυχαθών ή περισσότερη άμυψη σπορά, γενικώ καλλιέργειες που είναι φιλικές προς τις μέλισσες. Σε ό,τι αφορά τις ενώσεις μελισσοκόμων, δυστυχώς είναι ελάχιστες. Καλό θα ήταν λοιπόν να ενισχύσουμε και το δικό τους ρόλο. Και τέλος, να πω ότι αυτή τη στιγμή και ο τομέας ζάχαρης στην Ευρωπαϊκή Ένωση αντιμετωπίζει κρίση εξαιτής αύξησης της τιμής ε, της ζάχαρης. Και αυτό επηρεάζει και τη μελισσοκομεία. Γι' αυτό θα ήθελα να σας ζητήσω να υποστηρίξετε την πρότασή μου που ζητά Η ζάχαρη που χρησιμοποιείται από τους μελισσοκόμους για τον εμπλουτισμό του μελιού να εμπίπτει στην κατηγορία της βιομηχανικής ζάχαρης για να ε, είναι πιο φθηνή. Σημαντικά θέματα είναι η έρευνα, η υγεία, τα φάρμακα, η περιορισμένη χρήση φυτοφαρμάκων, επιστημιστική ασφάλεια πρέπει να γίνει μια συνδυασμένη εξέταση όλων αυτών των παραγόντων και με μέτρα συγκεκριμένα για τη μελισσοκομία. Όλα αυτά θα πρέπει φυσικά να γίνουν σε συνεργασία με τα κράτη-μέλη. Και φυσικά και οι ενός μελισσοκόμων θα πρέπει να συμμετέχουν στην όλη διαδικασία. Μόνο με συνεργασία όλων των ενδιαφερομένων θα καταφέρουμε να λύσουμε το πρόβλημα, έως θα περάσει άλλη μια εικοσαετία και θα βρισκόμαστε στο ίδιο σημείο γιατί όπως είπε η κυρία Λούλινγκ, εδώ και 20 χρόνια όλα το ίδια ακούμε και δεν έχει γίνει τίποτα σημαντικό. Νομίζω ότι αυτή τη φορά μπορούμε να επιλύσουμε το πρόβλημα άπαξ και διαπαντός. Μάλιστα, σας ευχαριστούμε πολύ. Κύριε Ταμπάτση, πριν ε, να δώσουμε το λόγο στους συναδέλφους ε, που το ζήτησαν, ε, θα ήθελα να καλωσορίσω συνάδελφο Λαβία Μισήλια, που είναι ε, φιλανδικό μέλος ε, του Ελεγκτικού Συνεδρίου. Νέβες, ευχαριστώ Πρόεδρε. Θα ήθελα καταρχήν ε, να συγχαρώ τον συνάδελφο, τον κύριο Συγητή, για την εξαιρετική παρουσίαση. Πραγματικά ιδιαίτερα εξαντλητικά προσέγγισε όλα τα θέματα που θίγουν την υγεία των μελισσών καθώς το θέμα αυτό είναι ζωτική σημασία για τη γεωργία και πρέπει να συνειδητοποιούμε το μεγάλο αντίκτυπο που ε, έχει ε, το θέμα αυτό της προστασίας της υγείας ε, των μελισσών λόγω της επικανίωσης. Είναι πάρα πολύ σημαντικό αυτό το ζήτημα για μας. Γι' αυτό λοιπόν εγώ εδώ στην εισαγωγή μου θα ήθελα να αναφερθώ σε τρεις πτυχές ε, που θεωρώ ότι είναι ιδιαίτερα σημαντικές. Καταρχήν, αυτό το θέμα απαιτεί μια εθνική προσέγγιση, η οποία υπάρχει μεν, αλλά χρειάζεται και μια ευρωπαϊκή προσέγγιση. Και στο πλαίσιο αυτό, εγώ θα έλεγα επίσης ότι απαιτούνται να υπάρχουν επικαιροποιημένες μελέτες ε, σχετικά με τον αντίκτυπο που μπορεί να ε, έχει υγεία των, των μελισσών και των επικέντρων μελισσών σε μια συγκεκριμένη περιοχή. Εμεί χρειαζόμαστε αυτά τα νούμερα, αυτά τα αριθμητικά στοιχεία, πραγματική αξιολόγηση του θετικού αντικτύπου για να μπορέσουμε να διεκδικήσουμε τα όσα είναι απαραίτητα για να εγγυηθούμε την ανάπτυξη του τομέα αυτό. Δεύτερη πτυχή. Είναι αλήθεια ότι περισσότεροι μελισσοκόμοι ε, εργάζονται σε μερική απασχόληση ε, στη μελισσοκομεία. Εγώ άκουσα το ότι είναι ερασιτέχνες. Ε, δεν είναι ερασιτέχνες, απλώς εργάζονται με μερική απασχόληση σε αυτό το τομέα, αλλά πράγματι λαμβάνουν κατάρτιση και μαθήματα και παρακολουθούνται στη δραστηριότητά τους. Αυτή η πτυχή είναι πάρα πολύ σημαντική, κυρίως όταν ε, η ΚΑΠ κάνει λόγο για τον ενεργό γεωργό. Αυτός ο μελισσοκόμος, ο οποίος ε, ε, απασχολείται μερικώς, είναι ενεργός αγρότης. Είναι ενεργός μελισσοκόμος, έτσι λοιπόν θα πρέπει εδώ να λάβουμε υπόψη τις ιδιαιτερότητες. Και τρίτη και τελευταία πτυχή που θα ήθελα εδώ να τονίσω έχει να κάνει συγκεκριμένα με τις ονομασίες προέλευση, την πιστοποίηση, την, την επισήμανση. Ε, είναι δυνατόν να υπάρχουν μείγματα με μέλη που προέρχονται από την Ασία. Αυτή είναι πολύ συνήθες, ιδιαίτερα συνήθες πρακτική. Αν εμεί στην Ευρώπη και σε διάφορες περιφέρειες ανάλογα με το τύπο του μελιού που παρουσιάζεται θέλουμε να έχουμε προσθεμένη αξία για ορισμένες ποικιλίε μελιού, δεν θα μπορέσουμε προσπαθήσουμε να το κατορθώσουμε όσο επιτρέπονται αυτά τα μείγματα, τα οποία ε, στη συνέχεια δεν αντικατοπτρίζονται και ορθά στην επισήμανση. Έτσι λοιπόν θα ήθελα και πάλι να ευχαριστήσω τον συζητητή. Σας ευχαριστώ που θα λάβετε υπόψη την ενίσχυση αυτών των πτυχών, να τονίσετε περισσότερο αυτές τις πτυχές, γιατί νομίζω ότι ε, με αυτόν τον τρόπο μπορώ να συνεισφέρω στην εξαιρετική εκθεσή σας. Σας ευχαριστώ. Ευχαριστούμε την κυρία Πατρεωνέδες. Γκαρσία παρακαλώ. Ευχαριστώ. Θα ήθελα να ευχαριστήσω την Ευρωπαϊκή Επιτροπή, τον εισηγητή, την κυρία Πατράου και όλους όσους ασχολούνται με το πολύ σημαντικό και ενδιαφέρον αυτό θέμα, πως είναι η μιλισσοκομεία για το μέλλον της Ευρωπαϊκής Γεωργίας. Θα ήθελα να υπογραμμίσω αυτό που είναι το πιο σημαντικό κατά τη γνώμη μου, να προσδιορίσουμε με ακρίβεια τους λόγους νησιμότητας των μελισσών πέραν των προκαταλήψεων, των δυσιδαιμονιών, των παλιών μας απόψεων, το πιο σημαντικό είναι και ξέρουμε πόσο μία προκατάληψη ή μία δυσιδαιμονία μπορεί να περιπλέξει την ε, ανέβρεση σωστής λύσης. Είχαμε την εμπειρία με το κολοβακτηρίδιο. Θα πρέπει να αποφύγουμε λοιπόν τέτοιε προκαταλήψει και να υποστηρίξουμε την Ευρωπαϊκή Επιτροπή στην προσπάθεια ενίσχυση των μέτρων επαγρύπνηση στα διάφορα κράτη-μέλη. Γιατί τα κράτη-μέλη είναι σε τελική ανάλυση ε, υπεύθυνα και θα πρέπει να δείξουν αυτή την ε, υπευθυνότητα στην προσπάθεια επίλυσης του προβλήματο. Βέβαια, η Ευρωπαϊκή Επιτροπή θα παίξει ένα συντονιστικό ρόλο. Ε, το θέμα των φυτοφαρμάκων είναι επίση σημαντικό. Στην Ισπανία υπάρχουν ήδη ε, σημαντικές μελέτες που δεν συνδέουν την θνησιμότητα των μελισσών με τη χρήση των φυτοφαρμάκων. Άρα δε, ίσως δεν είναι αυτή η αιτία. Οπότε τα διάφορα βιοκτώνα και τα φυτοφάρμακα δεν κυκλοφορούν στην Ευρωπαϊκή Ένωση χωρίς προηγούμενη μελέτη επιπτώσεων. Οπότε από τη στιγμή που δεν υπάρχει απόδειξη ότι σχετίζεται η θρησιμότητα των μελισσών με τα φυτοφάρμακα, γιατί να επιμένουμε. Τώρα άλλο το θέμα των γενετικώς τροποποιημένων οργανισμών. Η Ευρωπαϊκή Επιτροπή ήδη έκανε μελέτε για του γενετικώ τροποποιημένου οργανισμού και μέχρι στιγμή σε καμία περίπτωση, και το υπογραμμίζω αυτό, σε καμία περίπτωση δεν αποδείχθηκε κάποια σχέση, κάποια επίπτωση των γενετικώ τροποποιημένων οργανισμών στον πληθυσμό τη απικία των μελισσών. Και αυτό είναι παράλογο να συνεχίζουμε και να επιμένουμε ε, σε θέματα που έχουν λυθεί. Ούτε υπήρξε καμία προειδοποίηση ή κανένα επιστηστικό συναγερμό σε σχέση με του γενετικώ τροποποιημένου οργανισμού. Γιατί να επιμένουμε ότι υπάρχει κίνδυνο. Φαίνεται ότι αποκτούμε κάποιε ιδεολειψίε και επιμένουμε να αποδείξουμε κάτι όταν ήδη βλέπουμε ότι οι επιστημονικέ μελέτε δεν το αποδεικνύουν. ελπίζω να συνεχίσουμε την συνεργασία γιατί ο στόχος μας είναι κοινό, είναι να σταματήσει αυτή η καταστροφή ενός πολύ σημαντικού εργαλείου όπως είναι η μελισσοκομεία και η συμβολή των μελισσών στην Ευρωπαϊκή Γεωργία. Ευχαριστώ. Ευχαριστούμε κύριε Γκαρσία. Συνάδελφος Ρέιμες για το Πινόσκινγκ. Ευχαριστώ και εγώ θα ήθελα να ευχαριστήσω τον συγητή για την δουλειά του. Ήταν πάρα πολύ ενδιαφέρον να διαβάζει κανείς αυτή την έκθεση. Λίγα πράγματα λείπουν. Αυτό το οποίο είναι σημαντικό για εμένα είναι πως όταν μιλάμε για παρακολούθηση να έχουμε ενιαίες ευρωπαϊκές προδιαγραφές γιατί βλέπουμε πως όταν κάνει ο καθένας τη δική του παρακολούθηση σε κάθε χώρα δεν είναι συγκρίσιμα τα στοιχεία και αν ε, το πρόβλημα είναι σε ευρωπαϊκό επίπεδο και πρέπει να το καταπολεμήσουμε σε ευρωπαϊκό επίπεδο, πρέπει να μπορούμε να έχουμε τα ίδια δεδομένα και σημαντικό είναι να υπάρχει μια συνολική στρατηγική. Και νομίζω πως ε, θα πρέπει να υπάρξει μια καταγραφή των ε, μελισσοκόμων, γιατί δεν ξέρουμε μέχρι σήμερα πραγματικά πόσοι είναι οι μελισσοκόμοι και πόσες είναι οι κυψέλες, τα μελίσια και Νομίζω φτάνουν ε, λίγες πηγές ε, μόλυνσης σε αυτές τις πολύ μικρές επιχειρήσεις για να βρεθούν νοκάουτ ε, ορισμένες επιχειρήσεις και περιοχές. Οπότε θα πρέπει να ενημερώνονται οι αγρότες λέτε από τους μελισσοκόμους βεβαίως για να, πριν χρησιμοποιήσουν κάποια ε, φάρμακα. Οπότε πράγματι βεβαίως αυτό σημαίνει πως θα πρέπει να υπάρχει αμοιβαία ενημέρωση και από πλευράς των ε, γεωργών. Για να μην, υπάρχουν, ε, για να μην υπάρχει οργή και επιθετικότητα όπως έχει εμφανιστεί σε ορισμένες τέτοιες περιπτώσεις. Νομίζω με τα σύγχρονα μέσα που υπάρχουν και από τις ε, δύο πλευρές και θα έχουμε στην ε, διάθεσή μας, εάν ε, επενδύσουμε περισσότερο στην έρευνα και έχουμε βεβαίως και νέες εξελίξεις στα φάρμακα, να έχουμε κάποια πρόοδο. Ευχαριστώ. Σας ευχαριστώ. Μάρτιν Όσλινγκ έχει τώρα τον λόγο. Ναι πρώτα απ' όλα να συγχαρώ τον εισηγητή για την έκθεσή του αν ε, ανέφερε κάποια πράγματα. Δεν θέλω τώρα να διαφωνήσω με την κυρία Γκαρσία, δεν μου είναι ευχαριστώ, αλλά το ότι έχουμε πρόβλημα σε πολλά σημεία με τα ζυζανιοκτώνα ε, δεν μπορεί να το διαψεύσει κανείς. Στη Γερμανία είχαμε πέρσι ε, ένα περιστατικό που επηρέασε πολλά μελίσια γιατί χρησιμοποιήθηκε στο ένα φυτοφάρμακο, ένα μέσο φυτοπροστασίας. Και υπάρχει νομίζω ανάγκη εδώ πέρα να δράσουμε και πρέπει να τα πούμε αυτά τα πράγματα ανοιχτά. Δηλαδή να παριστάνουμε ότι είναι όλα εντάξει και δεν υπάρχει καμία ανάγκη δράσης είναι λάθος. Βεβαίω, το λένε οι μιλισσοκόμοι. Η βαροϊκή ακαρίαση παραμένει το μεγαλύτερο πρόβλημα, αλλά υπάρχουν ε, πάρα πολλά πράγματα που συνεισφέρουν ε, ε, στο να επιτείνεται αυτή η δύσκολη κατάσταση μέσω των φυτο... μέσων φυτοπροστασίας. Επίσης, παρά το ότι αμφισβητείται, εγώ θεωρώ πως πρέπει να ερευνήσουμε το ζήτημα των γενετικά τροποιημένων οργανισμών και εκεί πέρα υπάρχουν διαφορετικές έρευνες. Τώρα μην ισχυριστώ πως ε, έχουν ερευνηθεί τα πάντα όσον αφορά του γενετικότητα τροποποιημένους οργανισμούς και δεν υπάρχει πρόβλημα, κάθε άλλο. Ίσως να υπάρχουν σε έρευνες στην Ισπανία, εγώ πάω πάντως προς την άλλη κατεύθυνση. Για τα αντιβιωτικά που αναφέρθηκαν και αυτό είναι ένα πρόβλημα, ειδικά όσον αφορά την προστασία των καταναλωτών πράγματι, αλλά νομίζω πως ε, ένα πράγμα είναι επίσης σημαντικό να αναφερθεί. Έχουμε πολλούς μελισσοκόμους που είναι, κάνουν αυτή τη δουλειά ως χόμπι και τους δυσκολεύουμε και δεν υπάρχει, ξέρετε, μια επόμενη γενιά για να έρθει σε αυτή τη δουλειά. Είναι δύσκολη δουλειά και δεν τους την κάνουμε ευκολότερη. Και θα ήθελα να επενδύσουμε στο να προωθήσουμε μια νέα γενιά και πανευρωπαϊκά σε όλα τα κράτη-μέλη για να έχουμε και καλύτερη κατάρτιση των μελισσοκόμων. Το τελευταίο αναφέρθηκε ο τομέας της ε, νέας γεωργικής πολιτικής και συγκεκριμένα η προώθηση της βιοπικιλότητας είναι βασικό αυτό για την ε, κοινή γεωργική πολιτική. Έχουμε μεγάλη απώλεια της ε, βιοπικιλότητας και αυτό βεβαίως ε, δεν είναι μόνο θέμα των... για να βρίσκουν τροφή οι μέλισσες Τώρα, όπως είπαν και οι προλύσαντε, είναι πάρα πολύ σημαντικό να ενισχύσουμε χρηματικά την έρευνα και τον συντονισμό. Γιατί γίνει, υπάρχει πάρα πολύ έρευνα, αλλά δεν χρησιμοποιούνται τα αποτελέσματα. Οι μελισσοκόμοι λοιπόν αναμένουν ε, στην Ευρώπη να κάνουμε κάτι για τον κλάδο τους. Eichhout και μετά Ευχαριστώ κύριε Πρόεδρε, ευχαριστώ και τον εισηγητή, ε, τον κύριο Ταμπαϊντή, για το θέμα των μελισσών, γιατί είναι κρίσιμο και νομίζω πως το αντικατοπτρίζει αυτό ε, η έκθεση. Για όσους λένε πως πρέπει να βασιζόμαστε στην επιστήμη, νομίζω πως είναι σαφές ε, το από πού ξεκινάει ο κύριος Ταμπαϊντή. Αλλά εάν δεν είναι αντικειμενική η επιστήμη, ή αν υπάρχουν κάποια εμπόδια ε, για να βρούμε τα δεδομένα, τότε είναι σαφές ε, πως πρέπει να βασιζόμαστε στην ε, επιστήμη και να έχουμε πρόσβαση, πρόσβαση σε όλα τα δεδομένα που υπάρχουν. Οπότε, καλά τα λέει ο εισηγητής. Ένα θέμα που νομίζω ακόμα δεν αναφέρεται επαρκώς στην έκθεση είναι το ζήτημα του ότι η γεωργία γίνεται όλο και περισσότερο μονοκαλλιέργεια. Και είναι ζήτημα για τις μέλισσες. Να δώσω ένα παράδειγμα στη ΣΥΠΑ, και δεν έχουμε φτάσει βεβαίως ακόμα σε αυτή τη θέση, είναι ένα καλό παράδειγμα για το που οδεύουμε. Π.χ. στην παραγωγή των αμυγδάλων, η πολιτεία, στην πολιτεία της Καλιφόρνιας, όπου παράγονται, ξέρετε, 80% των αμυγδάλων, ε, ξέρετε πως πηγαίνουν εκεί πέρα, μεταφέρουν τις μέλισσες ε, για ένα μήνα για την επικονίαση. Και επί ένα μήνα βεβαίως στρέφονται με το ίδιο λουλούδι, με τον ίδιο ανθό. Οπότε και αυτή η γεωργία δημιουργεί προβλήματα για τις μέλισσες. Οπότε ε, ξέρουμε πως υπάρχει πρόβλημα με τη βαροϊκή ακαρίαση, υπάρχει πρόβλημα με τα ζυζανιοκτώνα, με τους μελισσοκόμους, αλλά και οι μέλισσες, και οι μέλισσες πρέπει να έχουν ε, μια διατροφή ε, ποικιλόμορφη και υπάρχει βεβαίως το ζήτημα της ποράς ε, και πράγματι θα πρέπει να το τονίσουμε αυτό και για τις μέλισσες. Πρέπει να το αναφέρουμε αυτό. Αναφέρεται στις ψηφιματικές δηλώσεις νομίζω αλλά πρέπει να αναφέρετε και πιο πολύ στην έκθεση. Κατά λοιπά καλωσορίζουμε νομίζω αυτή την έκθεση γιατί πρέπει να έχουμε όλα τα δεδομένα, να γίνει περισσότερη έρευνα, να έχουμε γνώση για να μπορέσουμε να αντιμετωπίσουμε τους διάφορους παράγοντες που είναι όπως είπα και η μονοκαλλιέργεια και όλα αυτά τα ζητήματα. Και να δώσουμε λίγο λιγότερο βάρος επίσης ε, στα φάρμακα γιατί τελικά αν έχουμε καλύτερη γνώση και περισσότερη ποικιλία στη γεωργία τότε θα χρειαζόμαστε νομίζω λιγότερα φάρμακα για να μην φτάνουμε στο σύμπτωμα, μπορούμε να αντιμετωπίσουμε την πηγή του προβλήματος. Ευχαριστούμε λοιπόν τον κύριο Ταμπαϊντή και ε, υποστηρίζουμε την έκθεση τόσο για αυτή τη στιγμή. Ωραία, σας ευχαριστώ, ο κύριος Μπουβέ. Και εγώ θα ήθελα να ευχαριστήσω τον εισηγητή μας, τον κύριο Ταμπάτζη, είναι αλήθεια ότι έχουμε πρόβλημα σήμερα με την θνησιμότητα μελισσών στη μελισσοκομεία. Φτάνει μερικές φορές το 70% και το 80% σε ορισμένες περιοχές. Και όντως, μέχρι σήμερα είχαμε κάποιες επιστημονικές μελέτες και η τελευταία που δημοσιεύτηκε τον τελευταίο μήνα από ένα ειδικευμένο περιοδικό που ασχολείται με αυτό το θέμα επισήμανε ένα νέο φαινόμενο που θα πρέπει να μας απασχολήσει και να μας προβληματίσει και γι' αυτό και να συνεχίσουμε την προσπάθειά μας. Το γεγονός ότι σήμερα δεν είναι μόνο ένα χημικό προϊόν, ε, προϊόν που μπορεί να δημιουργήσει η θνησιμότητα, δεν είναι κατά ανάγκη τα φάρμακα, οι χημικά προϊόντα που δημιουργούν, προκαλούν το θάνατο των ε, μελισσών. Αυτό που ανακαλύφθηκε είναι ότι κάποια παράσιτα, εντερικά παράσιτα της μέλισσας, όταν αναμειγνύονται με ελάχιστες ποσότητες, πυροελάχιστες ποσότητες προϊόντων και έγιναν ε, κάποιες ε, συγκρίσεις με το καλυψό της μπάγερ ή ένα άλλο φάρμακο, δείχνει ακόμη και με ελάχιστες ποσότητες ε, ε, πρόβλημα στις μέλισσες. Έχουμε αυτό το πρόβλημα δηλαδή που δημιουργείται, το νέο φαινόμενο, ε, την, τις παραδοσιακές, μέλισσες, ε, παραδοσιακές παθήσεις των ε, μελισσών με τη χρήση των νέων χημικών προϊόντων. Και ο συνδυασμός αυτών των δύο μερικές φορές έχει ολέθρια συνέπεια για την υγεία των μελισσών. Και αυτό θα πρέπει να μα προβληματίσει για την πιστοποίηση των προϊόντων, γιατί ίσω δημιουργήσει δύσκολε και καινοφανεί καταστάσει. Και εδώ θα πρέπει να δώσουμε την προσοχή μα, γιατί αυτό ο συνδυασμό, αυτό το κοκτέιλ είναι που δημιουργεί πρόβλημα ε, Και αυτό που ανακάλυψαν οι ερευνητέ τι τελευταίε εβδομάδε, αυτό το συνδυασμό κάποιων ε, ε, παρασίτων που έχουν ήδη μέληση όταν έρχονται σε επαφή με τα νέα χημικά προϊόντα, αυτό είναι που θα πρέπει να μα απασχολήσει και να μα φέρει σε νέα σκέψη. Ο κύριο Καπόλα Σάντο. Ευχαριστώ Πρόεδρε, αγαπητοί συνάδελφοι. Πολύ σύντομα θέλω να παρέμβω εγώ εξ ονόματο τη ομάδα των Σοσιαλιστών και Δημοκρατών να πω ότι ευχαριστούμε πάρα πολύ τον συγητή. Θέλουμε να τον συγχαρούμε για το έργο του, Καθώ ε, φαίνεται να διαχειρίζεται ένα θέμα το οποίο χαίρει συνένεση ε, και έτσι λοιπόν ε, δεν θα ήταν σωστό να μην τοποθετηθώ κι εγώ και να πω ότι αναγνωρίζουμε πλήρω αυτό το έργο και ελπίζω να τύχει, με, να τύχει έγκριση. Σε ευχαριστώ Λούί Να δώσω τώρα το λόγο στου εκπροσώπου τη Ευρωπαϊκή Επιτροπή, τον Διευθυντή

Επρόκειτο για ένα έγγραφο που απευθυνόταν και στο Συμβούλιο και στο Κοινοβούλιο, προκειμένου να προκληθεί συζήτηση επί του θέματος αυτού. Και εμείς, όπως και ο συγητής, θεωρούμε ότι είναι πάρα πολύ σημαντικό αυτό το θέμα και ήταν πάρα πολύ σημαντικό για μας ε, να έχουμε feedback από τα δύο αυτά όργανα. Η Ευρωπαϊκή Επιτροπή Ήδη έχει προβεί σε μια σειρά δράσεων, ανάληψη δράσεων, για να προσπαθήσει να βελτιώσει την κατάσταση σε ό,τι αφορά στην υγεία των μελισσών. Ήδη ένα τμήμα των δράσεων αυτών περιγράφονται στην ανακοίνωση και άλλες ήδη έχουν αναλυφθεί και θα πρέπει να ολοκληρωθούν. Άκουσαμε ικανοποίηση και από την πλευρά του συγητή και από τους εξαιτούμους και τους βουλευτές που τοποθετήθηκαν ότι οι δράσεις που αναλάβαμε απαντούν σε όσα ζητήθηκαν και ακούστηκαν σήμερα. Υπογραμμίστηκε συγκεκριμένα η σημασία μιας παρακολούθησης ε, της εθνισμότητας των πολισών με έναν εναρμονισμένο τρόπο και αυτό σημαίνει ότι θα πρέπει να γίνεται αυτή η παρακολούθηση με νέο τρόπο σε όλα τα κράτη-μέλη γιατί κάτι τέτοιο θα μας επιτρέψει να έχουμε βασικά δεδομένα επί των οποίων θα μπορέσουμε να εργαστούμε σοβαρά και με σταθερά, στερές βάσεις, σταθερά στοιχεία στερές βάσεις. Επίσης συμφωνούμε ότι δεν είναι εύκολο το καθήκον αυτό το έργο αυτό, γιατί ο κόσμος της μελισσοκομείας παρουσιάζει πολλές ιδιαιτερότητες, όπως υπογραμμίστηκε. Έχουμε πολλούς ε, μελισσοκόμους, ε, οι οποίοι ασχολούνται πιο ρωστακτικά και φυσικά αυτό περιπλέκει τα πράγματα όταν μιλάμε για παρακολούθηση και αποπτία. Έτσι λοιπόν, ε, με το Ευρωπαϊκό Εργαστήριο Αναφοράς για την Υγεία των Μελισσών, που συστήθηκε και λειτουργεί από την 1η Απριλίου. Εργαζόμαστε για να καταλήξουμε σε ένα πιλωτικό σχέδιο με τα κράτη-μέλη, προκειμένου να μπορέσουμε να καταλήξουμε σε μια, οργανισμένη, σε μια ε, ενιαία μέθοδο που θα μπορούσε να χρησιμοποιηθεί από όλα τα κράτη-μέλη. Θεωρούμε ότι αυτό είναι ένα πολύ σημαντικό βήμα, ένα πολύ σημαντικό σημείο αφετηρίας. Έχουν ξεκινήσει ήδη και άλλε ε, πρωτοβουλίες σε ό,τι αφορά την απλούστευση της νομοθεσία για τα κτηνιατρικά φάρμακα. Και εδώ η Κομισιόν θα συνεχίσει τι εργασίε ε, με τον πλέον αποτελεσματικό τρόπο. Μπορώ να σας πω ήδη ότι μετά τι καλοκαιρινές διακοπέ θα λάβει η χώρα μια συνεδρίαση με τα ενδιαφερόμενα μέρη, ακριβώς ε, για να συζητήσουμε τη νέα νομοθεσία για τον τομέα αυτό. Και Φυσικά θα λάβουμε υπόψη και όλα όσα ακούστηκαν σήμερα. Αυτά είναι τα σχόλιά μου. Μάλιστα, ευχαριστούμε κύριε Μπερνόριο. Κύριε Νούμερ, θέλετε το λόγο, παρακαλώ. Ναι, ευχαριστώ. Να υπενθυμίσω στην Επιτροπή πως ε, πέρσι το Σεπτέμβριο θετήσαμε το, τα προγράμματα μελισσοκομείας για τα κράτη-μέλη και καταφέραμε να έχουμε επιπλέον χρηματοδότηση, οπότε τα επόμενα τρία χρόνια θα έχουμε 32 εκατομμύρια για το 2011, 2012 και 2013 που θα διατεθούν στα κράτη-μέλη. Υπάρχει συγχρηματοδότηση, οπότε το 32 εκατομμύρια σημαίνει πως θα φτάσουν 64 ε, εκατομμύρια στον κλάδο και σε σύγκριση με το προηγούμενο πρόγραμμα μιλάμε για μια αύξηση κατά 25%. Νομίζω πως είναι αρκετά καλό βήμα προς τα εμπρός. Ε, ευχαριστώ. Μάλιστα. Πολύ ωραία. Σημειώθηκε πρόοδο τώρα. Το λόγο έχει ο κύριο Σταμπάτζη για να ε, εξαγάγει κάποια συμπεράσματα σε σχέση με τι ερωτήσει που έθεσαν οι συνάδελφοι. Παρακαλώ. Ευχαριστώ. Σε ό,τι αφορά στις ερωτήσει που τα έθεκαν, νομίζω ότι δεν δημιουργείται ιδιαίτερη πολεμική. Νομίζω ότι απλώ υπάρχουν κάποιες διαφοροποιήσει σε σχέση με το που πρέπει να δοθεί έμφαση. Κυρίω ε, σε ό,τι αναφέρεται την πραγματική αιτία της κατάσταση. κατάστασης. Να πούμε ότι κυρίως ε, οι νέες και άγνωστες ε, νόσοι ε, είναι αυτό που πρέπει να δούμε. Γιατί παίρνουμε το σχάρι για τη βαρολική κρίση δεν υπάρχει αποτελεσματικό φάρμακο. Τώρα, σε όσα είπε ο κύριος ε, Μποβέ συγκεκριμένα, αναφερθήκατε στις συνέργειες που τις έχω αναφέρει και εγώ στο κείμενό μου, δηλαδή αυτή την αναφορά ότι υπάρχουν μια σειρά ε, συνδυαζόμενων παραγόντων. Υπάρχει και μεγάλη συζήτηση εδώ μεταξύ των ε, κυρίων βουλευτών ε, για τα αποτελέσματα και τις επιπτώσεις των βιοκτώνων και των φυτοφαρμάκων. Εγώ θεωρώ ότι αυτό είναι δευτερογενής παράγοντας. Η κύρια αιτία είναι διαφορετική. Όμως, Βεβαίως, αν ε, δείτε τι λέω το σημείο 18 εκεί υπάρχει συγκεκριμένη αναφορά σε μια σειρά δραστικών ε, ουσιών και ε, φυτοφαρμάκων που θεωρώ ότι θα πρέπει να απαγορευτούν γιατί εδώ έχουμε αποτελέσματα μελετών και δείχνουν ότι ε, αυτά τα προϊόντα βλάπτουν ιδιαίτερα την υγεία των μελισσών. Όμω το θέμα αυτό για τα φυτοφάρμακα και το βιοκτών είναι ιδιαίτερα πολύπλοκο στη χώρα μου. Τη δεκαετία του 70 και του 80 χρησιμοποιούνταν ε, πάρα πολλά παρασιτοκτόνα και βιοκτόνα, δηλαδή στην κεντρική Ευρώπη γενικότερα. Και δεν ε, είδαμε άμεσα τις επιπτώσεις, δεν ε, είδαμε την καταστροφή όπως ε, αυτή που λαμβάνει χώρα σε όλη την Ευρώπη. Όπως είπε και ο Γιώργος Μπεβέ, υπάρχουν πολλοί παράγοντες και η μονοκαλλιέργεια. Επίσης είναι παράγοντες, δηλαδή υπάρχει επιρροή διάφορων παραγόντων. Όμως εγώ θα ζητούσα από την Κομισιόν πάρα πολύ σοβαρά να μελετήσει το κύριο θέμα κατά την άποψή μου, δηλαδή πώς μπορούμε να έχουμε ε, στην αγορά προϊόντα που να καταπολεμούν πραγματικά τους παθαγόνους παράγοντες, γιατί διαφορετικά δεν μπορούμε να αντιμετωπίσουμε το πρόβλημα αυτό. Και ένα άλλο κάπως πολεμικό θέμα, σε αυτό αναφέρθηκαν ε, συνάδελφοι Γκαρσία και Χάουσλινγκ για τους γενετικά τροποποιημένους οργανισμούς. δεν υπάρχουν επιστημονικές μελέτες που να μας υποδεικνύουν αν οι γάμματα φόμικρον ε, έχουν αρνητικές επιπτώσεις ή αν ε, δεν έχουν επιπτώσεις στην υγεία των μελισσών. Έτσι λοιπόν, ε, το επίσης η Κομισιόν ε, να προβεί στην ε, εκπόνηση μιας μελέτης για το θέμα αυτό, γιατί τώρα δεν υπάρχουν στοιχεία ούτε υπέρ ούτε κατά, δεν υπάρχει μελέτη ακόμη. Και βάσει προσωπικών επαφών με την Κομισιόν, το είπε και ο κύριος Εκχάουτ, θα ήταν ε, πολύ σημαντικό κάτι τέτοιο. Βέβαια δεν μπορούμε να παρεμβούμε στην επιστήμη. Πάντοτε βέβαια διακυβεύεται εδώ και υπάρχει και το θέμα της χρηματοδότησης. Κύριε Πρόεδρε, όταν συνομιλούμε με του Αμερικανού συναδέλφου, πάντοτε ανέκυπτε το θέμα αυτό, γιατί αυτοί πάντοτε αναφέρονται στην επιστήμη. οι επιστήμονε λένε αυτό, όμω τελικά ποιο χρηματοδοτεί την επιστήμη, ε, η Μοσάντο, η Αμερικανική κυβέρνηση ή η Ευρωπαϊκή Ένωση. Αυτά πρέπει να τα έχουμε κατά νου. Γιατί χρειάζεται χρηματοδότηση για να μελετήσουμε και τα βιοκτών αλλά και τους γενετικά τροπομένους οργανισμούς. Ό,τι αφορά τώρα το θέμα της, ε, των ονομασιών προέλευσης ε, και των γεωγραφικών ενδείξεων, ε, συμφωνώ που το, και χαίρομαι που το αναφέρατε αυτό, συμφωνώ με την κυρία Γκαρσία ότι δεν μπορούμε να θεωρήσουμε ότι είναι υπεύθυνα 100% τα φυτοφάρμακα, αλλά φυσικά έχουν και αρνητικέ επιπτώσεις. Αυτό δεν μπορούμε να το απορρίψουμε. Και ο Λίνος είπε κάτι πολύ σημαντικό. Χρειάζεται μια συνδυασμένη βάση δεδομένων, το είπε και γιατί αν ε, δεν μπορούμε να συγκρίνουμε τα στοιχεία, τότε δεν μπορούμε να αντιμετωπίσουμε τα προβλήματα του εν λόγω τομέα. Αν ε, δεν ξέρουμε πόσες κυψέλες υπάρχουν σε μια χώρα, από πού ξεκινάμε. Δηλαδή υπάρχουν χώρες για τις οποίες δεν υπάρχει κανένα στοιχείο. Και όλοι το γνωρίζουν. Δεν θα αναφέρω ονόματα εδώ, αλλά όλοι το γνωρίζουν το θέμα αυτό και είναι πολύ σημαντικό. Τώρα, αυτό το θέμα που εμφανίζεται και στην ε, έκθεσή μου έχει να κάνει με το θέμα της παρακολούθησης και εποπτείας. Πρέπει να γίνεται με έναν ομοιόμορφο τρόπο σε όλη την Ευρωπαϊκή Ένωση. Διαφορετικά δεν μπορούμε να αντιμετωπίσουμε το πρόβλημα. Κύριε Άσλινγκ, ε, κύριε Άσλινγκ, με συγχωρείτε, είπατε τι σκέφτεστε και σε ό,τι αφορά τα αντιβιωτικά. Νομίζω ότι είναι ένα θέμα που δεν έχει ρυθμιστεί το θέμα του μελιού και συζητείται πάρα πολύ το θέμα αυτό στην Ουγγαρία. Στην περίπτωση, παραδείγματο χάρη του κρέατο, ε, υπάρχουν και εκεί πάρα πολλά αντιβιωτικά, αλλά δεν υπάρχει ένα κοινό κανόνα. Η Γερμανία έχει ε, ένα κατώτατο όριο που επιτρέπει, αλλά αυτό διαφέρει σε κάθε χώρα και ίσω ε, κάποιε χώρε δεν μπορούν να θέσουν σε εμπορία την ίδια ποσότητα. Αυτό πρέπει να το λύσουμε. Σε ό,τι αφορά τώρα την αμύψη σπορά. Υπάρχει μια σχετική αναφορά στην εκθεσή μου, αλλά μπορούμε φυσικά να δώσουμε μεγαλύτερη έμφαση και να εξηγήσουμε τα θέματα αυτά στην έκθεση. Θέλω να ευχαριστήσω και την κυρία και την Κόπα Κοσέγκα και όλους όσους με βοήθησαν και όλους όσους συνέβαλαν στην εκπόνηση της έκθεσης αυτής, γιατί συνεργαστήκαμε και με πυρογνώμονες και επιστήμονες στον τομέα αυτό και ελπίζω να μπορέσουμε όλο ένα περισσότερο να διευκρινίζουμε τα στοιχεία και να μπορέσουμε να λάβουμε δράση. Η Κομισιόν και τα κρότη μελη θα πρέπει να στρωθούν στη δουλειά από τώρα και ελπίζω να μπορέσουμε να τα καταφέρουμε. Μάλιστα, σας ευχαριστώ πολύ. Σας ευχαριστώ και για την ποιότητα της εργασίας σας και για το πάθος σας. Λοιπόν, προθεσμία κατάθεσης τροπολογιών 30 Αυγούστου, 12 το μεσημέρι. Και τώρα, ας περάσουμε πολύ γρήγορα στο σημείο 6 της ημερησίας διάταξης. Ε, σας επενθυμίζω ότι στις 4.30 θα έρθει ο Επίτροπος Τσόλος. Επομένως, πρέπει να καταφέρουμε να το συζητήσουμε σε 20 λεπτά. Χάρτης πορείας για ε, μετάβαση σε μια ανταγωνιστική οικονομία χαμηλών ε, πέδων εκπομπών δεξιού του άνθρακα για το 2050. Μπίλιντα Γκλαντφέντερ είναι συντάκτρια της ομοδότησης. Πρόκειται για ε, μια γνωμοδότηση για την Επιτροπή Περιβάλλοντος. Είναι πάρα πολύ σημαντικό και λεπτό το θέμα αυτό. Πολλές φορές σε αυτή την Επιτροπή είπαμε ότι η Γεωργία αποτελεί βέβαια τμήμα του προβλήματος, αλλά και τμήμα της λύσης. Γι' αυτό θα δώσω τώρα το λόγο στην κυρία Κλατφέντερ για την παρουσίασή της και κατόπιν θα κάνουμε και μια σύντομη συζήτηση. Παρακαλώ. Ευχαριστώ κύριε Πρόεδρε. Σήμερα πρωτοστατούν οι Ούγγροι ομιλητέ και εγώ Ουγγρικά θα μιλήσω. Θα σας παρουσιάσω το σχέδιο γνωμοδότησής μου. Όπως ξέρετε η Ευρωπαϊκή Επιτροπή εκπώνησε μία ανακοίνωση με θέμα της ε, μεταρρύθμισης της ευρωπαϊκής βιομηχανίας, ώστε μέχρι το 2050 να μειώσουμε δραστικά κατά 80% τα, ε, τις εκπομπές αερίων θερμοκηπίου. Επίσης αναφέρει ένα άλλο πολύ σημαντικό θέμα εδώ για την υλοποίηση αυτού του στόχου, το ρόλο που θα πρέπει να αναλάβει η γεωργία για να συμβάλλει στην υλοποίηση αυτής της δραστικής περικοπής των ε, αερίων του θερμοκηπίου. Βέβαια, όπως λέει και η ανακοίνωση, η γεωργία αυτή τη στιγμή δεν μπορεί να αντικαταστήσει όλα τα ορυκτά καύσιμα από άλλες πηγές ενέργειας. Για παράδειγμα, για την παραγωγή λιπασμάτων καταναλώνεται μεγάλη ενέργεια, αλλά είναι απαραίτητο αυτό. δεν μπορούν να καταργήσουν τη χρήση καυσίμων, οπότε θα είναι μερική αυτή η, η περικοπή. Άλλωστε, η γεωργία δεν καταναλώνει μόνο ενέργεια, την παράγει, για παράδειγμα, παράγοντας βιοκαύσιμα ή βιομάζα, που είναι σημαντική πηγή ενέργειας πια στην Ευρωπαϊκή Ένωση και τα βιοκαύσιμα περιέχουν ένα τεράστιο δυναμικό για την ενεργειακή πολιτική της Ευρωπαϊκής Ένωσης. Ιδιαίτερα θα περάσουμε στα βιοκαύσιμα δεύτερης γενιάς. Άλλωστε, οι εκπομπές αερίων θερμοκηπίου θέλουμε να μειωθούν αισθητά αλλά θα πρέπει να αποφύγουμε κατά την υλοποίηση αυτού του στόχου κάποιες αντιφάσεις. Για παράδειγμα, δεν θα πρέπει να έχουμε στην Ευρωπαϊκή Ένωση υπέρογγες τιμές άνθρακα που δεν θα μπορέσουν να τις καταβάλουν οι ενδιαφερόμενοι, γιατί έτσι θα δημιουργηθεί στρέβλωση ανταγωνισμού και θα έρθουν σε δυσμενή θέση τα ευρωπαϊκά προϊόντα, μια και οι ευρωπαίοι παραγωγοί θα δυνατούν να καταβάλουν τις υψηλές τιμές. Μπορείτε να διαβάσετε το κείμενο της γνωμοδότησης, αν θέλετε πιο διεξοδική παρουσίαση. Να επισημάνω όμως κάτι που δεν αναφέρεται στο κείμενο και είναι χρήσιμο να συζητηθεί. Στο μέλλον θα συζητήσουμε την μεταρρύθμιση της κοινή γεωρικής πολιτικής. Και συμφωνώ με όσους πιστεύουν ότι θα πρέπει να, ε, να αφιερώσουμε περισσότερα κονδύλια και στην ανάπτυξη της υπαίθρου, αλλά και στην ε, γεωρική πολιτική, προκειμένου να βοηθήσουμε τους γεωργούς να συμβάλλουν στη μείωση των εκπομπών αερίων του θερμοκηπίου και να επενδύσουμε και σε ανανεώσιμες πηγές ενέργειας στην ύπεθρο, στις γεωρικές ζώνες. Βιομάζα, αιωλική ενέργεια, ηλιακή ενέργεια, γεωθερμική και ούτω καθεξής, ώστε στην επόμενη επταετία να δημιουργηθούν οι προϋποθέσεις με κατάλληλη χρηματοδότηση ανάπτυξη πέθρου για να δοθεί έμφαση σε ανανεώσιμες πηγές ενέργειας στην Ήπεθρο. Και να θέσουμε και κάποιους ελάχιστους στόχους στα κράτη-μέλη σε ό,τι αφορά τη χρηματοδότηση των ανανεώσιμων πηγών ενέργειας στην Ήπεθρο. Και αν ένα κράτος δεν υλοποιήσει αυτούς τους στόχους, σε ό,τι αφορά το ποσοστό χρήσης ανανεώσιμων πηγών ενέργειας, τότε να μην μπορεί να εκταμιεύσει τα διαθέσιμα κονδύλια. Επαναλαμβάνω, αν ένα κράτος μέλος δεν υλοποιεί τους στόχους για τις ανανεώσιμες πηγές ενέργειας να έχει περιορισμένη πρόσβαση σε κονδύλια και για άλλα θέματα. Δηλαδή να μην μπορεί να χρησιμοποιήσει τα κονδύλια για άλλα σημεία, άλλα, άλλους τομείς της γεωργικής πολιτικής. Να υποχρεωθεί το κράτος να υλοποιήσει τους στόχους και τις δεσμεύσεις που έχει αναλάβει για τις ανανεώσιμες πηγές ενέργειας στην Ήπεθρο. Ευχαριστούμε κύριε Γκλαντφέντερ. Θα ξεκινήσουμε τη συζήτηση τώρα. Θα έρθει και ο κύριος Τζόλος ε, μάλιστα είναι εδώ, Τζολάιν. Ε, ε. Ευχαριστώ κύριε Πρόεδρε, ευχαριστώ και τον κύριο Γκλαντφέντερ Μιλάω εξ ονόματος ε, μια συναδέλφου βεβαίως που παρακολουθεί αυτή την έκθεση να αναφέρω δύο-τρία πράγματα. Πρώτα απ' όλα είναι μια πάρα πολύ καλή αρχή αυτή η έκθεση αλλά μπορούμε να είμαστε πιο φιλόδοξοι για να εξηγήσουμε ε, καλύτερα το πώς ε, μπορεί να συνεισφέρει ο τομέας γεωργίας και αν δείτε την ανάλυση της ίδιας Επιτροπής ε, λέει πως μέχρι το 2050 μπορούν να μειωθούν οι εκπομπές ε, μέχρι 50% σε σχέση με τα επίπεδα του 1990. Επίσης πρέπει να πούμε ξεκάθαρα πως η Γεωργία έχει νομίζω πάρα πολύ καλό ιστορικό μείωση των εκπομπών μέχρι στιγμής, ε, κυρίως μέσω αποτελεσματικότητας της παραγωγής και άρα μπορούμε να τα πάμε πολύ καλύτερα στο μέλλον αρκεί να υπάρχουν κίνητρα και οπωσδήποτε θα καταθέσουμε κάποιες τέτοιες ε, τροπολογίες. Οπότε νομίζω πως μπορούμε να γίνουμε πιο φιλόδοξοι για το τι θέλουμε να πετύχουμε σε σχέση μάλιστα με, άλλες, ε, με άλλους κλάδους όπου έχουν μειωθεί με τον ίδιο τρόπο σημαντικά εκπομπές. Ευχαριστούμε George. Eichhout. Θα είμαι και εγώ σύντομο γιατί θα συμφωνήσω και εγώ με τον κύριο Λάιον. Ε, συμφωνούμε με την έκθεση ως μια βάση γιατί νομίζω πως ακόμα η κλιματική αλλαγή θεωρείται περισσότερο απειλή και όχι ευκαιρία και πρέπει να αλλάξουμε τον τόνο, τον πυρήνα της έκθεσης, γιατί αν δούμε τις προκλήσεις του μέλλοντος που είναι βεβαίως ε, παραγωγή τροφίμων, κλιματική αλλαγή, βιοπικιλότητα, η γεωργία βρίσκεται στο κέντρο και μπορεί να παίξει ένα πολύ σημαντικό ρόλο που να μπορεί να ανταποκριθεί από πλευράς κλίματος, να μειωθεί το εξωτερικό κόστος ε, μέσω των ε, διαφόρων παραγωγών παραγωγής και βεβαίως να είναι πιο βιώσιμη και νομίζω πως αυτή η αμοιβαία υποφελής κατάσταση μπορεί να είναι πιο σαφής και εμείς θα καταθέσουμε κάποιες τροπολογίες ε, για να περιγράψουμε αυτή την ευκαιρία. Εάν δείτε τον άνθρακα στο έδαφος που οδηγεί σε περισσότερη αντοχή στο κλίμα αλλά προσφέρει και καλύτερες δυνατότητες για υψηλότερη παραγωγή και μειώνει ταυτόχρονα την εξάρτηση από λοιπάσματα που εξαρτώνται από το πετρέλαιο κτλ. Εάν δούμε το πώς θα κλείσει ο κύκλος των τροφίμων, να επανασυνδεθεί ξανά η παραγωγή αρωτρέων καλλιεργειών ε, με την παραγωγή ζωικού κεφαλαίου, να μειωθούν δηλαδή αλυσίδες, η ε, κρίκη της τροφικής αλυσίδας. Όλα αυτά νομίζω, όλες αυτές οι ευκαιρίες θα πρέπει να αναφέρονται πολύ περισσότερο στην έκθεση για να καταστήσουμε σαφές πως το θέμα του κλίματος είναι κρίσιμο για τη γεωργία. Αλλά πρέπει να είμαστε τολμηροί και να το δούμε σε βασικό επίπεδο. Γιατί αν συνεχίσουν τα πράγματα ως συνήθως, τότε έχετε δίκιο κύριε Γκλάτφελντερ, πως θα επιτύχουμε μόνο κάποια μείωση. Αλλά αν το δούμε αλλιώς, και επανασυνδεθεί νομίζω η παραγωγή αρωτρέων και ζωικού κεφαλαίου μπορούμε να δούμε ε, τις αλλαγές που θα γίνουν για να είναι αμοιβαία υποφιλής η κατάσταση. Χάουσλινγκ, μία σύντομη συμπλήρωση πρέπει να είναι σαφές πως είμαστε υποχρεωμένοι και στη Γεωργία να έχουμε κλιματικούς στόχους. Γιατί είναι πολύ προσεκτικά διατυπωμένο το πρώτο σημείο. Μπορούμε να είμαστε πιο φιλόδοξοι εδώ πέρα μπορεί να συνεισφέρει περισσότερα γεωργία. Και κάτι άλλο θέλω να αναφέρω. Δεν θα πρέπει να μην αναφέρουμε ορισμένα πράγματα. Μιλάμε για μεγάλη παραγωγή σε χώρες ε, εκτός ε, Ευρώπης, μιλάμε για 30 εκατομμύρια εκταρίων που χρησιμοποιούνται για την παραγωγή ζωοτροφών εντός της ε, Ευρώπης. Αυτό συμβαίνει εντός της Ευρώπης και πρέπει να το πούμε και η βιοενέργεια πως μπορεί να είναι μια αμοιβαία επωφελής κατάσταση αλλά να είμαστε ειλικρινεί. δεν μιλάμε για την ε, δεύτερη γενιά καυσιμών πρέπει να γίνει ήδη αποτελεσματικότερη η πρώτη γενιά και να χρησιμοποιήσουμε υπολείμματα και όχι όπως γίνεται στη Γερμανία στη λάθος κατεύθυνση να έχουμε μεγάλες ε, μονοκαλλιέργειες καλαμποκιού και εκεί πέρα λοιπόν πρέπει να έχουμε αποτελεσματικότερη χρήση τη ενέργεια. Ευχαριστώ Μάρτιν Εράν Καρσία. Ευχαριστώ, Πρόεδρε. Θέλω να ευχαριστήσω τον κύριο Κλαντφάιτερ για το έργο του και να κάνω κάποιε παρατηρήσει, Όταν ε, λέμε ότι ο γεωργικό τομέα έχει κάποιο μικρότερη δυναμική από άλλου τομεί σε ό,τι αφορά τη μείωση των εκπομπών, ε, μπορώ να σα πω ότι ο γεωργικό τομέα είναι λιγότερο δυστυχώ από όλου του οικονομικού τομεί και είναι και πιο γενναιόδωρος ε, σε ό,τι αφορά το περιβαλλοντικό σκέλος ε, γιατί ουσιαστικά το διοξείδιο του άνθρακα μετατρέπεται σε οξυγόνο και αυτό είναι κάτι πολύ σημαντικό και δεν μπορούν να το κάνουν άλλοι οικονομικοί τομείς στην Ευρώπη. Ε, μέρα με ανησυχούν δύο σημεία της ε, έκθεσης Gladfeder ε, σημείο 6, όταν αναφέρεται στο ότι η πολιτική για τη διαβίωση των ζώων θα πρέπει να θέτει σε κοινό τους στόχους της οικονομίας χαμηλών επιπέδων των εκπομπών. Νομίζω ότι κάπως υπερβάλλουμε εδώ η ελεύθερη διακίνηση των αγαθών θα μπορούσε να υποστεί επιπτώσεις γιατί υπάρχουν σε όλα τα 27 κράτη-μέλη θέματα μεταφοράς αγαθών που θίγουν και το περιβάλλον και την κτηνοτροφία. Και κατόπιν λέτε ότι η Ευρωπαϊκή Ένωση αποκλειστικά χρωματοδοτεί ε, ε, προγράμματα ενεργειακής αποδοτικότητας. Μήπως ε, θα μπορούσαμε να θέσουμε φρένο, δηλαδή με αυτόν τον τρόπο, στην ε, ιδιωτική πρωτοβουλία εδώ. Ε, εγώ δεν θα ήθελα σε καμία περίπτωση αυτή η αποκλειστικότητα της Ευρωπαϊκής Ένωσης να θέσει φρένο στην ιδιωτική πρωτοβουλία, γιατί πιστεύω ότι η ιδιωτική πρωτοβουλία είναι πάρα πολύ σημαντική και στον τομέα γεωργίας και εκτινοτροφίας. Αυτά από μένα. Ευχαριστώ πολύ. Πολύ ωραία. Λουίς, έχεις το λόγο. Ευχαριστώ. Εγώ αντικαστώ την κυρία Κάριν Κάτεμπαχ που είναι η σκιώδη συγγήτρια εδώ και θα ήθελα να διαβάσω στον εισηγητή ότι εκτιμούμε ιδιαίτερα στη γνωμοδότηση που τη θεωρούμε ισορροπημένη και θα την ε, υπερψηφίσουμε αλλά θα ήθελα να επιστήσω την προσοχή σας σε 34 σημεία για τα οποία και θα καταθέσουμε τροπολογίες. Καταρχήν, στο σημείο 1 της γνωμοδότησης ο εισηγητής αναφέρει ότι το δυναμικό μείωση ε, εκπομπών στη Γεωργία είναι σχετικά μικρό. Κι όμως ξέρουμε τι προσπάθειες έχει κάνει η Γεωργία για να μειώσει τις εκπομπές σε πιο Πολύ περισσότερο προσπάθησαν η Γεωργία από οποιοδήποτε άλλο. Νομίζω ότι με την διατύπωση που υιοθετεί ο θα δίνει σφαλμένο μήνυμα στην κοινωνία. Γιατί ε, λέγοντας ότι είναι περιορισμένο το δυναμικό μείωσης, ε, δίνω ένα αρνητικό μήνυμα. Θα προτιμούσα να δώσουμε έμφαση σε μια πιο θετική διατύπωση. Σε ό,τι αφορά τις επενδύσεις, πολύ σωστά ο εισηγητής ζητά επενδύσεις σε πράσινη φιλοπεριβαλλοντική ενέργεια. Ναι, ε, να, λέμε πράσινη ενέργεια, αλλά που θα παράγεται με αηφόρες μεθόδους. Γιατί δεν αρκεί να λέμε πράσινη ε, ενέργεια, γιατί ακόμη και η πράσινη ενέργεια, όταν η μέθοδη παραγωγής δεν είναι κατάλληλη, μπορεί να είναι επιζήμια για το περιβάλλον. Επίσης μιλάει ο εισηγητής για επενδύσεις μόνο σε εγκαταστάσεις που παράγουν ενέργεια με ανανεώσιμες, από ανανεώσιμες πηγές. Εγώ θα έλεγα να μην είμαστε τόσο κατηγορηματικοί να πούμε αποκλειστικά, να πούμε κατά προτίμηση τέτοιες εγκαταστάσεις, όχι αποκλειστικά εγκαταστάσεις και να τονίσουμε και πάλι με μεθόδους ε, γεωργικές που μπορούν να προαγάγουν τη μείωση των εκπομπών. Πιστεύω ότι με τις μικρές αυτές διορθώσεις ε, θα βελτιώσουμε την ήδη πολύ καλή γνωμοδότηση του εισηγητού. Ευχαριστώ. Ευχαριστώ, Λουίς. Τώρα θα ζητήσω από τον εκπρόσωπο της ε, Κομισιόν, Βαν Χιλάν, από την ομάδα ΕΛΤΑ για την κλιματική αλλαγή, να πάρει το λόγο και κατόπιν θα δώσουμε το λόγο και πάλι στον εισηγητή. Παρακαλώ. Ευχαριστώ. Θέλω να ευχαριστήσω την Επιτροπή για τη συνεισφορά της ε, για αυτό το σχέδιο ψηφίσματος, ε, για μια οικονομία με χαμηλές εκπομπέ άνθρακα. Καλωσορίζουμε την πρόταση αυτή, αλλά θέλουμε να τονίσουμε ορισμένα στοιχεία που θεωρούμε ότι μπορούσαν να υπάρξουν βελτιώσει. Ορισμένοι από του ομιλητέ ήδη πρότειναν ότι η διατύπωση μπορεί να ερμηνευτεί ως περιορισμένο δυναμικό. Είναι αλήθεια στο έγγραφο μα λέμε ότι σε σύγκριση με άλλου τομεί, όπω ο ενεργειακό τομέα, ο γεωρικός τομέα, μπορεί να μειώσει λιγότερο μακροπρόθεσμα τις εκπομπέ ε, λόγω της αύξησης του πληθυσμού, που ξέρουμε, και τις επόμενες δεκαετίες. Παρ' όλα αυτά, έχουμε 42-49% έναν αριθμό για τις μειώσεις ε, και μπορεί να ξεχνάτε ότι ε, εξακολουθεί να υπάρχει αυτή η δυναμική εκεί έξω. Όπως είπε και η Κομισιόν ε, στο έγγραφο της ε, για τις δραστηριότητες σχετικές με το κλίμα μέχρι το 2020, ε, τέτοιες δραστηριότητες μπορούν να λάβουν χώρο και ναι, στο γεωργικό τομέα. Έτσι λοιπόν ο γεωργικός τομέας εξακολουθεί να μπορεί να συνεισφέρει στο μετριασμό της κλιματικής αλλαγής στην επόμενη δεκαετία. Υπάρχει και μια αναφορά στο ότι η γεωργία παρέχει βιοκαύσιμα και μπορεί να οδηγήσει οδηγήσει στι χαμηλότερε εκπομπέ στην οδική ένωση, αλλά αυτό θα πρέπει να γίνει και με ένα βιώσιμο τρόπο. Έτσι λοιπόν στην ανακοίνωση τονίζουμε ότι πρέπει να σκεφτούμε την χρήση των γεών με καθολικό τρόπο. Και ε, ένα σχόλιο για το ότι η γεωργία ε, έχει να κάνει με την διαρροή του άνθρακα και το αναφέρουμε και εμεί αυτό. Λέμε ότι υπάρχει ένα τέτοιο κίνδυνο διαρροή του άνθρακα, όμω η γεωργία δεν αποτελεί τμήμα της, του συστήματο εμπορία εκπομπών τη Ευρωπαϊκή Ένωση και με αυτά που αναφέρεται εδώ για τι τιμέ ε, μπορεί να παρερμηνευτεί γιατί κάτι τέτοιο δεν υπάρχει. Δηλαδή δεν υπάρχει τιμή του άνθρακα στο γεωργικό τομέα αυτή τη στιγμή. Ευχαριστώ πολύ. Ευχαριστούμε πολύ τον εκπρόσωπο της Κομισιόν. Παρακαλώ, εισηγητής έχει το λόγο για να κλείσει προθεσμία για την καταστροπολογία 14 Ιουλίου, 12 το μεσημέρι. Παρακαλώ. Ευχαριστώ κύριε Πρόεδρε. Πολύ σημαντικό αυτό το τελευταίο που είπατε, η διορία για την κατάθεση τροπολογιών και ελπίζω ότι όντως θα καταθέσουν τροπολογίες οι συνάδελφοι για την γνωμοδότηση. Μερικοί το προανήγγυλαν ήδη, μακάρι. Επίσης θα ήθελα να πω ότι μας περιορίζουν εδώ οι διατάξεις για, τις διαστάσεις, για το εύρος ε, της γνωμοδότησης. Είμαστε υποχρεωμένοι να παραμείνουμε σε συγκεκριμένη έκταση και γι' αυτό θα ήθελα να ζητήσω από τη γραμματεία να εξετάσει με ελαστικότητα αυτές τις διατάξεις και να μπορέσω να επιμικίνω κάπως τη γνωμοδότησή μου. Όπως είπαν κάποιοι συνάδελφοι, ορισμένες παρατηρήσεις είναι πολύ σημαντικές, αλλά πραγματικά δεν χωρούσαν στη γνωμοδότηση, γιατί δεν μπορούσα να είμαι πιο α, Με τις τροπολογίες σας, σας παρακαλώ να εμπλουτίσετε τη γνωμοδότηση για να περιλάβουμε και άλλα στοιχεία και λεπτομέρειες. Και μην ξεχνάτε την προθεσμία για την κατάθεση των τροπολογιών. Γιατί όσο περισσότερες τροπολογίες καταθέσουμε, τόσο πιο καλό θα είναι το αποτέλεσμα της γνωμοδότησης, γιατί θα είναι πιο ευρία η συνένεση. Ένα λεπτό διακοπή μόνο για να δώσουμε την ευκαιρία στον ε, Επίτροπο να έρθει και να καθίσει και μετά θα περάσουμε στη συζήτηση του σημείου 5.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 Iniziamo. Allora possiamo Μπορούμε να ξεκινήσουμε. Καταρχήν θέλω να καλωσορίσω τον Επίτροπο, τον κύριο Ντατσαντσόλο, ο οποίος θα μας παρουσιάσει τα σχόλιά του για τις ε, επιπτώσεις ε, της ε, πρότασης ε, για το πολιτέ δημοσιονομικό πλαίσιο που θετήθηκε προσφάτω. Ε, Όπω γνωρίζετε υπήρξαν πάρα πολλά σχόλια όταν ε, παρουσιάστηκε η δημοσιονομική πρόταση και Μάλιστα, εκφράστηκαν και πάρα πολλέ ανησυχίε. Φανταζόμαι θα συστεθούν και ορισμένε ερωτήσει γιατί ε, διαψεύτηκε εν μέρη το πάγωμα, ένα μερικό πάγωμα και θέλουμε εσείς ε, να μας ε, πείτε ε, πώς αιτιολογούνται αυτές οι περικοπές έναντι μιας τόσο φιλόδοξης μεταρρύθμισης που το Κοινοβούλιο και αυτή η Επιτροπή με τις εκθέσεις Lion και Des συνσέφερε και έδωσε και μία πρόθεση με ξεκάθαρη κοινοβουλευτική ψηφοφορία. Εμείς δεν θέλουμε περικοπή πόρων σε αυτή την πολιτική, γιατί αυτή η πολιτική όχι μόνο θα πρέπει να διασφαλίζει και να ανταποκρίνεται στα συμφέροντα των 10 εκατομμυρίων γεωργών στην Ευρώπη, αλλά και όλων των πολιτών των 550 εκατομμυρίων της Ευρωπαϊκής Ένωσης. Έτσι λοιπόν, θα δώσουμε το λόγο πρώτα στους ε, ε, συντονιστές αφού θα έχει τοποθετηθεί ο Επίτροπος. Έχουμε μια μισή ώρα χρόνο. Είναι πάρα πολύ σημαντικό το ζήτημα. Γι' αυτό θα δώσω απευθείας το λόγο στον Επίτροπο, στον κύριο Τσόλος. Παρακαλώ. Merci, euh, Monsieur Ευχαριστώ κύριε Πρόεδρε. Χαίρομαι για την εισαγωγή σα, γιατί διαπιστώνω ότι έχει μείνει αμύωτος ενθουσιασμό σας και φιλοδοξία σας ό,τι αφορά τον κοινοτικό προϋπολογισμό για την κοινή γεωρική πολιτική. Και ελπίζω το γεγονό ότι η φιλοδοξία του Κοινοβουλίου είναι μεγαλύτερη από τις επιτροπή ό,τι αφορά το γεωργικό προπολογισμό δεν μπορεί παρά να με χαροποιεί. Βέβαια τώρα το μπαλάκι βρίσκεται στο πεδίο του Συμβουλίου και ανάλογα με την έκβαση θα ενεργήσει και η Ευρωπαϊκή Επιτροπή. Και μάλιστα η Ειδική Επιτροπή ΣΟΥΡ με την έκθεσή της είχε ζητήσει από την Ευρωπαϊκή Επιτροπή ένα πάγωμα του γεωργικού προϋπολογισμού, του προϋπολογισμού για την ΚΑΠ το 2013. Και πάνω σε αυτή τη βάση οι υπηρεσίες προϋπολογισμού της Ευρωπαϊκής Επιτροπής εργάστηκαν και αυτή θα είναι η πρόταση για την κοινή γεωργική πολιτική. Ένα πάγωμα της ονομαστικής αξίας του προϋπολογισμού που δεν περιλαμβάνει τον πληθωρισμό για τον πρώτο και τον δεύτερο πυλώνα, αλλά θα επανέλθω πιο διεξοδικά ε, στα επιμέρους αυτά σημεία. Σε ό,τι αφορά το ονομαστικό πάγωμα ε, στο επίπεδο του 2013 με βάση την αξία του ευρώ του 2011, την ισοτιμία του ευρώ του 2011, ήταν για ευρώ και είναι το ποσό που περιέχει η ανακοίνωση της Ευρωπαϊκής Επιτροπής 371,7 δις ευρώ. Γιατί βλέπω ότι στον τύπο και σε όλες τις συζητήσεις ε, μιλούμε για, για ευρώ. Με την τρέχουσα αξία, γιατί αυτή χρησιμοποιείται, με την τρέχουσα αξία είναι 418,4 δις ευρώ. Αυτή είναι η βάση για το ονομαστικό πάγωμα ε, χωρίς τον πληθωρισμό για τον πρώτο και δεύτερο πυλώνα. Ο πληθωρισμός όμως ε, του πρώτου πυλώνα ε, προϋπέθεται μία διόρθωση 1% για την τρέχουσα περίοδο. Γι' αυτό και υπάρχει μία μείωση της αξίας του προπολογισμού της ΚΑΠ στο συνολικό προπολογισμό γιατί δεν λαμβάνεται υπόψη αυτό το 1% του πληθωρισμού. Και με το 1% χρηματοδοτήσαμε την σταδιακή ε, αύξηση χρηματοδότηση των νέων κρατών μελών μετά την ε, διεύρυνση δηλαδή. Γιατί η διεύρυνση έγινε με το ίδιο επίπεδο προπολογισμού. Και αυτή ήταν η δική μου ανησυχία, αυτό ήταν το δικό μου μέλημα με τον επιπλέον αυτό πληθωρισμό στον πρώτο πυλώνα ε, χρηματοδοτήσουμε την σταδιακή εισαγωγή των νέων κρατών μετά το 2014 χωρίς να πειράσουμε το γενικό επίπεδο των άμεσων πληρωμών. Και τελικά αποδεσμεύσαμε από τη δεύτερη κατηγορία κάποιες πληρωμές που εμπίπτουν στο χαρτοφυλάκιο του Επιτρόπου Γεωργίας και συνδέονται με την κοινή γεωργική πολιτική, αλλά θα χρηματοδοτηθούν από άλλες κατηγορίες. Έτσι αποδεσμεύσαμε το απαραίτητο ποσό προκειμένου να συνεχίσουμε τη χρηματοδότηση της σταδιακής εισαγωγής του phasing in χωρίς αυτό να επηρεάσει το ύψος των άμεσων πληρωμών. Έχουμε δηλαδή εδώ κάποιες πληρωμές για την εκρίζωση ή την εξάλληψη ε, φυτικών, ε, ε, νόσων ή επιζωτιών 2,5 ε, εκατομμυρίων ευρώ. Επίσης ε, για 2,8 δις ευρώ σε τρέχοντα ευρώ, 2,5 ευρώ για σταθερά ευρώ για τους ε, πλέον χρήζοντες βοήθεια Βέβαια, εδώ η Γενική Διεύθυνση Άγκρη ε, διαχειρίζεται αυτά τα προγράμματα. Υπήρξε μια διεύρυνση τη νομική βάση και σε ό,τι αφορά τα μέτρα τη αγορά, μια και κάθε χρόνο έχουμε για τις ε, παρεμβάσει αγοράς ε, πολλά κονδύλια που προσπαθούν να μετριάσουν τις επισταστικές κρίσεις όπως συνέβη με τα κυβευτικά πρόσφατα ή με την ιδιωτική αποθήκευση για το χείριο κρέας την Άνοιξη μετά την κρίση της διοξίνης στη Γερμανία. Αυτά τα μέτρα πια δεν επιβαρύνουν τον πρώτο πυλώνα της δεύτερης κατηγορίας, αλλά μπήκαν σε μια εξωτερική ξεχωριστή κατηγορία 3,9 εκατομμύρια τρέχοντα, δις 3,5 δις σταθερά. Επίσης 2,9 δισεκατομμύρια τρέχοντα ευρώ. Θα, με, θα, ε, χρηματοδοτήσουμε το facing in χωρίς να επηρεάσουμε τις άμεσες πληρωμές. Γιατί μέχρι στιγμής ε, αυτό το χρηματοδοτούσαμε από την αύξηση του 1% του, του πληθωρισμού κάθε χρόνο. Και επειδή εξελίχθηκε αυτό το 1% ο πληθωρισμός, προσπαθήσαμε να αποδεσμεύσουμε κονδύλια από τη δεύτερη κατηγορία, χρηματοδοτώντας την ΚΑΠ και από άλλες κατηγορίες. Επιπλέον, ενισχύσαμε κάτι που στο παρελθόν χρηματοδοτούσαμε από το δεύτερο πυλώνα. Πολύ συχνά μιλήσαμε για την ανάγκη ενίσχυσης ε, του δεσμού μεταξύ των γεωργών και της έρευνας και τεχνολογικής ανάπτυξης. Στόχος μου ήταν τα πλαίσια του δεύτερου πυλώνα να χρηματοδοτήσω αυτές τις δράσεις για την καινοτομία, την τεχνολογική ανάπτυξη και το σχετισμό γεωργίας και έρευνας και τεχνολογικής ανάπτυξης. Γι' αυτό και προβλέψαμε 5,1 δις ε, τρέχοντα ευρώ στην πολιτική έρευνας που έχουν προσημαθεί για το πρόγραμμα χρηματοδότησης έρευνας και τεχνολογικής ανάπτυξης για τη γεωργία ειδικά. Για πρώτη φορά η Ευρωπαϊκή Επιτροπή προβλέπει στον προπολογισμό της έρευνας ένα ειδικό κονδύλιο για τη γεωργία, κάτι που θα μας επιτρέψει να χρηματοδοτήσουμε ένα γνήσιο πρόγραμμα εφαρμοσμένης έρευνα για να δούμε αυτή τη σχέση παραγωγής, γεωργίας και έρευνας. Και επίσης αυτό το πρόγραμμα θα χρηματοδοτηθεί πλήρως από την Ευρωπαϊκή Ένωση. Είναι 100% κοινοτικό προπολογισμό από ένα κονδύλιο τη έρευνα. Αρχικά ήθελα να το θέσω στο δεύτερο πυλώνα της ΚΑΠ, αλλά στο δεύτερο πυλώνα θα έπρεπε να με εμπίπτει στην εθνική συγχρηματοδότηση. Μια όμως και έχουμε ειδικό κονδύλιο στην έρευνα για τη γεωργία, θα μπορέσουμε να εξασφαλίσουμε πλήρη κοινοτική χρηματοδότηση, 100% δεν χρειάζεται συγχρηματοδότηση και στα πλαίσια τη χρήση αυτού του προπολογισμού όλο το πλαίσιο θα ε, προσδιοριστεί από την κοινή γεωρική πολιτική και θα εμπίπτει στι δραστηριότητε τη Γενική Διεύθυνσης Άγκρη. Τώρα αυτό το ερευνητικό πρόγραμμα φυσικά θα ευθυγραμμίζεται με τους στόχους που έχουμε προσδιορίσει για την κοινή γεωργική πολιτική. Και μάλιστα θα σας υποβάλλω σχετικά σύντομα ε, μία πρόταση για την Ευρωπαϊκή Εταιρική Σχέση καινοτομία για τη Γεωργία που θα περιλαμβάνει και το τμήμα αυτής της χρηματοδότησης. Σε ό,τι αφορά το Ταμείο Παγκοσμιοποίησης, εκεί 2,8 δις τρέχοντα ευρώ, 2,5 δισεκατομμύρια σταθερά ευρώ προβλέψαμε ένα κονδύλιο για τη γεωργία, για την κοινή γεωργική πολιτική, για να χρηματοδοτήσουμε κάποιες ε, αποζημιώσεις για τους γεωργούς εξαιτία της επίπτωσης ε, της παγκοσμιοποίησης, της ρευστότητας των τιμών, στις ε, διεθνείς αγορές, που φαίνεται ότι πειράζουν όλο και περισσότερο το εισόδημα των γεωργών. Βέβαια, αυτή τη στιγμή δεν έχουμε ούτε δημοσιονομικά, ούτε κανονιστικά, ούτε νομικά εργαλεία και μηχανισμούς στην ΚΑΠ για να παρεβαίνουμε σε τέτοιες καταστάσεις. Αυτή τη στιγμή τώρα έχουμε ε, μια σώρευση μηχανισμών με τις άμεσες πληρωμές αφενός, με τα αμοιβέ μία αφετέρου που θα βάλουμε στο δεύτερο πυλώνα, αλλά και με τη δυνατότητα χρηματοδότησης από το Ταμείο παγκοσμιοποίηση, τέτοιων αποζημιώσεων αντισταθμιστικών μέτρων για τους γεωργούς. Αυτά τα 5,1 δις ε, τρέχοντα ευρώ για την έρευνα, 2,8 δις από το Ταμείο Παγκοσμιοποίησης είναι ε, κονδύλια που δεν υπάρχουν αυτή τη στιγμή ούτε στη νομική βάση ούτε ε, από το, στον προϋπολογισμό. Είναι χρήματα επιπλέον που προστίθενται στις, στους στόχους της ΚΑΠ που χρειάζονται επειδή δεν έχουμε πια τη διόρθωση με τον πληθωρισμό στο δεύτερο πυλώνα. Φτάνουμε λοιπόν σε ένα συνολικό ποσό 435,5 δις σε τρέχοντα ευρώ για την κοινή πολιτική, κάτι που προθέτει 486,9 σταθερά ευρώ, δις εκατομμύρια σταθερά ευρώ. Οπότε με αυτό το δημοσιονομικό κονδύλιο για την ΚΑΠ μπορούμε να χρηματοδοτήσουμε ναι μεν από διαφορετικές κατηγορίες αλλά να υλοποιήσουμε το στόχο της ΚΑΠ. Γιατί πολύ συχνά λέμε ότι η ΚΑΠ είναι τομεακή πολιτική με πολυκλαδική επίπτωση. Τώρα το βλέπουμε αυτό και στον προπολογισμό. Έχουμε την κοινωνική πολιτική αλλά και άλλες πολιτικές που χρηματοδοτούνται από την Ευρωπαϊκή Επιτροπή και μάλιστα η διάρθρωση του προϋπολογισμού αντικατοπτρίζει αυτή την πολυμορφία της ΚΑΠ και όλα αυτά τα κονδύλια, όλα αυτά τα ποσά και η χρηματοδότηση από διαφορετικές ε, ε, δημοσιονομικές γραμμές ε, θα εμπίπτουν στο χαρτοφυλάκιο του Επιτρόπου Γεωργίας και στις αρμόδιες διευθύνσεις Γεωργίας της Ευρωπαϊκής Επιτροπής και θα αντανακλούν το, τις αποφάσεις που θα λάβουμε από κοινού για το μελλοντικό νομοθετικό πακέτο της κοινή γεωργικής πολιτικής. Και τέλος θα ήθελα να σας υπενθυμίσω ότι ε, θα θυμάστε όταν είχα έρθει στα πλαίσια των ακροάσεων πριν διοριστώ Επίτροπος Γεωργίας, μερικοί με είχαν ρωτήσει ποια είναι η θέση μου ως προς κάποιες φημολογίες για τη μείωση της κοινή γεωργικής πολιτικής κατά 25-30% με βάση το πραγματικό κόστος. Για να δούμε με βάση αυτά τα στοιχεία που βρισκόμαστε. Νομίζω ότι αυτό ακριβώς ήταν το αποτέλεσμα όλων των κοινών προσπαθειών για να υποβάλουν μια κοινή γεωργική πολιτική που θα είναι πολύ πιο ανοιχτή προς την ευρωπαϊκή κοινωνία και που θα δικαιολογεί αδρό προπολογισμό. Η Ευρωπαϊκή Επιτροπή θέλησε να διαφυλάξει τις φιλοδοξίες της ως προς την κοινή γεωργική πολιτική, εξασφαλίζοντας ε, κάποια κονδύλια για να χρηματοδοτήσει και τις προτεραιότητες του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου αλλά να κρατήσει την κοινή γεωρική πολιτική και για τη μελλοντική δημοσιονομική περίοδος η βασική δαπάνη του κοινοτικού προϋπολογισμού. Η κοινή γεωρική πολιτική εξακολουθεί να είναι η πρώτη κοινοτική πολιτική με το μεγαλύτερο μερίδιο του κοινοτικού προϋπολογισμού, με βάση και τη νέα πρόταση της Ευρωπαϊκής Επιτροπής. Αυτά και αν έχετε περισσότερες απορίες, πολύ ευχαρίστω να σας δώσω και διευκρινήσεις. Δεν μπορούμε να αρνηθούμε ότι η Επίτροπος μας παρουσίασε πάρα πολύ καλά επιχειρήματα για την πρόταση αυτή ε, του Επιτροπή Λεβαντοφσκή και της Επιτροπής. Έτσι λοιπόν, ας ξεκινήσουμε τους συντονιστές των ομάδων. Καταρχήν, Αλμπερντές. Ευχαριστώ κύριε Πρόεδρε, κύριε Επίτροπε, κύριε Σόλος. Σας ευχαριστούμε που ήρθατε τόσο σύντομα μετά την παρουσίαση της ανακοίνωσης της Ευρωπαϊκής Επιτροπής και παρά τις ε, περικοπές ε, θέλω να σας ευχαριστήσω για την ε, προσπάθεια που κάνατε γιατί ξέρουν πως όλα τα μάτια ήταν στραμμένα στον προϋπολογισμό της Γεωργίας. Παρ' όλα αυτά πρέπει να διαπιστώσουμε πως η Ευρώπη μεγαλώνει. Θα πρέπει να επεκταθούν οι πλήρωμες ε, για τους ε, αγρότες. Ξέρετε πως ε, πάμε από τα 413 στα 360,9 όσον αφορά το ύψος της κοινή γεωργικής πολιτικής και βεβαίως πρέπει να συζητήσουμε την μείωση όταν μιλάμε ειδικά για ε, μια επικέντρωση μόνο στον τομέα της κοινή γεωρικής πολιτικής. Ε, το ΔΕ Κοινοβούλιο υποστήριξε πολύ την κοινή γεωρική πολιτική. Είχαμε και τη σχετική έκθεση η οποία έλεγε πως θα έπρεπε να παραμείνουμε στην ίδια τάξη μεγεθών. Και βεβαίως νομίζω πως ε, για αυτά τα οποία θα έρθουν. Νομίζω πως ε, θα έπρεπε να διατηρηθεί ο υπάρχον προπολογισμό της ε, κοινή γεωργικής πολιτικής χωρίς να κατηγορώ τώρα εδώ πέρα σας. Έχουμε ήδη μία πράσινη βίβλο για τα γεωργικά προϊόντα. αν δείτε τα μέσα τα οποία προβλέπονται εδώ πέρα για την ε, περικοπή όσον αφορά τα μέσα πρόθεση των προϊόντων μας, κάτι δεν ε, πάει καλά. Θα πρέπει λοιπόν να προσέξουμε να μπορέσουμε να στηρίξουμε την ε, κατανάλωση των προϊόντων μας και δεν ξέρω, μπορείτε να με διορθώσετε, αλλά από ό,τι διαβάζω εγώ αυτή τη στιγμή νομίζω πως έχουμε περικοπές. Επίσης κάτι το οποίο μου προξενεί εντύπωση είναι πως η Κομισιόν μπήκε ήδη στις ε, λεπτομέρειες. Μιλάει για ένα 13% για τα μέτρα πρασινίσματος ε, και το πώς θα διαμεριστούν όμως τα κράτη-μέλη. Αυτά αναφέρονται ήδη στην ανακοίνωση. Νομίζω πως ε, αυτό θα πήγαινε στην νομοθετική σας πρόταση και θεωρώ πως η Κομισιόν πήγε κάπως πολύ μακριά ήδη στην ανακοίνωση του προϋπολογισμού με το να μπει σε τόσες ε, λεπτομέρειες. Συνοψίζοντας, θα έλεγα πως η ομάδα μου, η ομάδα του ΕΛΚ, ε, κύριε Επίτροπε, θα σας υποστηρίξει έτσι ώστε η χρηματοδότηση της ε, γεωργικής ε, πολιτικής να έχει μια στέρεη βάση Είχατε πει όταν είχε εγκριθεί και η έκθεσή μου πως ε, θέλετε στήριξη από την Επιτροπή μας για να υπερασπιστούμε τα συμφέροντα Τη ε, κοινή γεωργική Πολιτική. Οπότε η ομάδα του ΕΛΚ θα συνεργαστεί μαζί σα, ε, κύριε Επίτροπε για να επιτύχουμε αυτό τον κοινό στόχο. Ευχαριστώ. Ευχαριστώ Άλμπερτ. Ευχαριστώ. Και εγώ θέλω να σας ευχαριστήσω για την παρουσία σας ε, εδώ σήμερα και για την ε, μόνιμη διαθεσιμότητά σας. Όλοι γνωρίζουμε τα, σε ποιο πλαίσιο ζούμε, πόσο δύσκολες είναι αυτές οι διαπραγματεύσεις ε, και φυσικά δεν αμφισβητώ τις προσπάθειες που καταβάλλατε για να πετύχετε το καλύτερο δυνατό προπολογισμό για τη Γεωργία. Όμως πρέπει να σας ομολογήσω ότι αυτή η πρόταση είναι μικρότερη από όσο περιμέναμε και είμαι μέλος αυτού του κοινοβουλίου που δύο φορές φέτος με συντριπτική πλειοψηφία ενέκρινε μια θέση ξεκάθαρη για το θέμα αυτό, μια θέση που υπερασπίζεται τη διατήρηση του προπολογισμού για τη γεωργία στο επίπεδο του 2013. Και έτσι λοιπόν κάτι τέτοιο θα πρέπει να ερμηνευτεί με ένα δημοσιονομικό επίπεδο σε, με πραγματικούς όρους. Δυστυχώς δεν είναι αυτό το οποίο συμβαίνει. Ήδη ακούσαμε διάφορα σχόλια και αντιδράσεις. Στο δικό μου γραφείο κάνουμε τους δικούς μας υπολογισμούς και θεωρούμε ότι θα έχουμε... Ε, ε πραγματική μείωση μεταξύ 7 και 20% 7 με 10% και θα θέλαμε κύριε Επίτροπε να μας εξηγήσετε ε, γιατί πρέπει να ξέρουμε πώς ε, το αποθεματικό για τις ε, κρίσεις είναι αγοράς πώς θα συμπληρώσει σε σχέση με τα εργαλεία της αγοράς που θα εγκρίνουμε ε, στο εσωτερικό της ε, ΚΑΠ. Ε, έχουμε κάποιες αμφιβολίες για το αν μπορούμε να χρησιμοποιήσουμε το χάρη κονδύλια από το Ταμείο για την παγκοσμιοποίηση, για την αντιμετώπιση της παγκοσμιοποίησης. Έτσι λοιπόν πραγματικά ποια είναι η πραγματική δυνατότητα να χρησιμοποιήσουμε αυτούς τους πόρους. Έχουμε κάποιες αμφιβολίες. Αυτή αποτελεί μια βάση εργασίας, η οποία δεν ανταποκρίνεται στις προσδοκίες μας, όμως είμαι σίγουρο ότι θα συνεχίσει να είναι ε, συνεπές ε, το Κοινοβούλιο και συνεκτικό σε σχέση με τις θέσεις που έλαβε δύο φορές ήδη και δεν πρόκειται μόνο για θέσεις των βουλευτών της Επιτροπής Γεωργίας, αλλά οι θέσεις αυτές αποσύστηκαν από την Ολομέλεια του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου. Έτσι λοιπόν ε, μπορείτε να μας δείτε ως συμμάχους για να βελτιωθεί ουσιαστικά η πρότασή σας και για να σας βοηθήσουμε με την επίτευξη ενός προπολογισμού που απαιτούν οι νέε προκλήσεις που διαφαίνονται ευχαριστώ. Ο George παρακαλώ. Κύριε Πρόεδρε, κύριε Επίτροπε, προσπαθείτε να υπερασπιστείτε τον ε, τομέα σα. Ε, δύσκολα τα πράγματα, Νομίζω πως ε, το Κοινοβούλιο βοήθησε να διατηρηθεί ο προπολογισμό. Μπορεί να μην έγιναν βεβαίως ε, τα όλα, όλα αυτά τα οποία ψήσαμε. Λοιπόν, αν δούμε τους αριθμούς και κάνουμε μία σύγκριση με τα στοιχεία του 2007-2013 σχέση με το προσωρινά τα οποία προτείνονται εδώ πέρα, οι περικοπές ε, στον τίτλο 1 είναι 50 δισεκατομμύρια ή 40 δισεκατομμύρια, να δούμε τα σύνολα των ε, δύο περίοδων. Οπότε θα έχουμε νομίζω ε, αρκετά, αρκετά σοβαρή περικοπή. Καταλαβαίνω πως βεβαίως υπάρχουν 15,2 ε, δισεκατομμύρια ευρώ που έρχονται από άλλες πηγές, αλλά αν δείτε την πολιτική συνοχής, έχουν εντύπωση πως σε πραγματικούς όρους ε, ε, έχουν ε, ελάχιστες περικοπές εκεί πέρα και νομίζω άρα πως οι σοβαρές περικοπές γίνονται στη Γεωργία. Δεν υπάρχει νομίζω εξορρόψη στα δύο μεγαλύτερα ποσά του ευρωπαϊκού προϋπολογισμού. Εάν δείτε τώρα του νούμερα ανά έτος, Μιλάμε για τον ε, τίτλο 2 με 60,3 δισεκατομμύρια και περνάμε σε 51,7 το έτος 2020. Πολύ σημαντική ε, μείωση. Αν δείτε δε τις άμεσες ενισχύσεις πάμε από 47 σε 38 δισεκατομμύρια. Ε, μιλάμε δηλαδή για περικοπές κατά 20%. Οπότε είμαστε σοβαροί όταν λέμε ότι μπορούμε να χρηματοδοτούμε τις άμεσες πληρωμές στο μέλλον χωρίς περικοπές. Πώς θα γίνει αυτό και ταυτόχρονα βεβαίως ε, θα αντιμετωπιστούν οι προσδοκίες των νέων μελών για υψηλότερη χρηματοδότηση στις άμεσες πληρωμές. Και θα έχουμε και άλλα δύο νέα κρατημέλη που θα ενταχθούν. Οπότε, δεδομένη τη ε, κλίμακα τη μείωση σε βάση, δεν βλέπω πώ θα καταφέρουμε να τα κάνουμε όλα αυτά. Εάν δούμε τώρα τα νέα κονδύλια που υπάρχουν στο σύστημα, αλλά δεν ξέρω εάν ε, είναι εκτός του τίτλου 2 και άρα εάν μπορούν να χρησιμοποιηθούν ε, ως αδιάθετα σε άλλους ε, τομείς, δεν ξέρω, θα ήθελα μια διευκρίνηση ως προς αυτό. Όσον αφορά λοιπόν το αποθυματικό για κρίση των 3,5 δισεκατομμυρίων, τι θα γίνει με αυτό, θα έχετε πρόσβαση σε αυτό, πώς θα μπορέσετε να χρησιμοποιήσετε αυτά τα λεφτά εάν υπάρχει μεγάλη πτώση των τιμών και χρειάζεται παρέμβαση. Και πάλι το ερώτημα είναι αν ε, δεν χρησιμοποιηθεί σε αιτήσια βάση τι γίνεται με αυτά τα λεφτά. Θα πάνε αλλού ή θα μπορεί να διατεθεί άλλο το χρονικά. Καλωσορίζω την αύξηση της επένδυσης σε έρευνα και ανάπτυξη. Πάρα πολύ θετικό. Αυτό το οποίο ενδιαφέρει ιδιαίτερα τη Σκωτία και το Ηνωμένο Βασίλειο και την Γαλλία είναι τα 2,5 δισεκατομμύρια του Ταμείου Παγκοσμιοποίησης για να αντισταθμίσουν τη συμφωνία με το Μερκοσούρ όσον αφορά ιδιαίτερα τα βοηδή. Οπότε καταλαβαίνω πρόκειται για μια εφάπαξ ε, πληρωμή για να προσαρμοστεί η κοινότητα. Τι σημαίνει αυτό. Ε, πληρώνουμε τους εκτροφείς ε, βοηδών για να αλλάξουν κατεύθυνση στην επιχείρησή τους ή τους πληρώνουμε για να κλείσουν την επιχείρηση. Θα ήθελα κάποιες απαντήσεις. Grazie George. Ο κύριος Νίκολσον, παρακαλώ. Ευχαριστώ. Ευχαριστώ πάρα πολύ κύριε Πρόεδρε. Να πω και εγώ πως άκουσα με μεγάλο ενδιαφέρον αυτά τα οποία είπατε και αναγνωρίζω πως ε, όταν ε, πρώτο ήρθατε εδώ πέρα το 2009 γίνονταν λόγος για περικοπές ε, στον προϋπολογισμό και νομίζω πως όλοι λέγαμε πως ε, και εγώ θα έλεγα τότε πως ε, είναι τρελές περικοπές που ακούγονταν για 25-30%. Το πρόβλημα με όλους τους ε, προϋπολογισμούς είναι πως όπως ξέρετε υπάρχουν ψέματα, μεγάλα ψέματα και στατιστικές. Οπότε πρέπει να δείτε πώς θα διασφαλίσετε το μέλλον. Αλλά νομίζω πως ξέρετε κύριε Επίτροπε και με παρεξηγήσετε Νομίζω πως ε, πρέπει να σας ευγενήσουμε τουλάχιστον για αυτά τα οποία ε, επιτύχατε. Η σκληρή αλήθεια είναι, αν δούμε την ιστορία της κοινή ε, γεωργικής πολιτικής, πως αποτελεί εύκολο στόχο για όλους εντός της Ευρώπης και όποιος θέλει να πάρει λεφτά από την κοινή γεωργική πολιτική θα τα προσπαθήσει να τα αποσπάσει και αυτή είναι η θέση που βρισκόμαστε εδώ και πολλά χρόνια. Οπότε Πώς θεωρείτε εσείς πως ο προϋπολογισμός σας ε, θα ενταχθεί ε, σε σχέση με αυτό το οποίο μας λένε αυτοί οι οποίοι μιλάνε για την ε, ασφάλεια των τροφίμων δηλαδή ως πρόβλημα. Μπορεί αυτός ο προϋπολογισμός να εξασφαλίσει κάτι τέτοιο και αυτή είναι νομίζω μια πρόκληση στην οποία θα πρέπει να ανταποκριθεί ο προϋπολογισμός αυτός είναι νομίζω ένα κριτήριο που θα πρέπει να εκπληρώσει. Μπορεί να ανταποκριθεί σε αυτές τις απαιτήσει και να πω πως ε, και εγώ καλωσορίζω τα κονδύλια για την έρευνα και ανάπτυξη. Στο παρελθόν το είχαμε παραμελήσει και οπωσδήποτε είναι κάτι θετικό. Το Ταμείο Παγκοσμιοποίησης είναι κάτι που με ενδιαφέρει όπως ε, και τους προλαλήσαντες. θα είναι το αντιστάθμισμα που θα δοθεί στους εκτροφείς βοηδών για συμφωνία με τη Μερκοσούρ για να έρθει από το παραθυράκι η συμφωνία αυτή και αν όχι με το Μερκοσούρ με κάποιον άλλο τομέα. Γιατί αν συμβαίνει αυτό κύριε Επιτροπέ, σας το λέω από τώρα, πως ε, θα σας ε, θα αντισταθούμε. Δεν φτάνει αυτό, δεν θα έρθετε εδώ πέρα γιατί ξέρετε πως οι Ευρωπαίοι αγρότες παλεύουν με το ένα χέρι δεμένο στην πλάτη, εισάγουμε τρόφιμα από άλλες περιοχές οι οποίες δεν παράγουν ούτε κατά διάνοια με τις ίδιες παρτιαγραφές που παράγουμε εμείς. δεν θα δεχτούμε εδώ πέρα να μας χρυσώσετε το χάπι, εάν αυτός είναι ο σκοπός σας. Το άλλο που παρατήρησα, η ευελιξία μεταξύ πυλώνα 1 και 2. Μιλάμε για τις μειονεκτικές περιοχές, μιλάμε για την ε, συγχρηματοδότηση από τις εθνικές κυβερνήσεις για να χρησιμοποιήσουν καλύτερα τα κονδύλια του πυλώνα 2 χωρίς να συγχρηματοδοτούν. Και ε, το άλλο θέμα στο οποίο θα ήθελα να κάνω μια ερώτηση και νομίζω πως ε, σχετίζεται με ένα σχόλιο που, ανέφερε ο κύριος, που έκανε ο κύριος Ντες πως ε, ίσως μπήκατε σε πολύ μεγάλο βαθμό λεπτομέρειες πάρα πολύ γρήγορα. Ε, γιατί αναφέρατε πως το 13% θα είναι για πρασίνισμα του πυλώνα 1. Γιατί εφόσον δεν υπάρχει ανάγκη αυτή τη στιγμή να, να ξεκινήσετε κάτι τέτοιο. Μπορούμε να το δούμε αυτό το ζήτημα του επόμενου 18 μήνε όταν θα φέρετε το... την ομοθετική πρόταση. Αλλά το να λέτε τώρα εδώ πέρα 30% για πρασίνισμα στον πυλώνα 1 δεν είναι αποδεκτό και θα είναι πάρα πολύ δύσκολο να κάνουμε κάτι. Γιατί ε, αυτή στιγμή ε, αρχίσουμε να μιλάμε για αυτά τα ζητήματα, δημιουργούμε περισσότερη γραφειοκρατία, και τα λεφτά δεν πάνε στον αγρότη που παράγει το φαΐ για την ασφάλεια των τροφίμων για να ταΐσουμε τους λαούς της Ευρώπης. Ευχαριστώ. Ευχαριστούμε. Μάρτιν Χόισλινγκ. Ναι κύριε Επίτροπε. Πρέπει εγώ να σας συγχαρώ για την πρόταση αυτή γιατί αν είμαστε ειλικρινείς πριν από ένα έτος δεν ήταν τόσο σίγουρο πως ε, θα έχουμε το ύψος ε, αυτό και θα μπορέσουμε να το διατηρήσουμε όσον αφορά τις πληρωμές της ε, κοινή γεωρικής πολιτικής. Θυμόμαστε non-papers που κυκλοφορούσαν και μιλούσαν για 30-40% περικοπές. Οπότε νομίζω πως μπορούμε να είμαστε ικανοποιημένοι με την πρόταση που έχουμε τώρα. Βεβαίως, αυτό δεν λέει τίποτα ακόμα για την κατανομή των, ε, των δαπανών. Αυτό είναι το συναρπαστικό θέμα βεβαίως. Πού θα πάνε τα λεφτά, πώς ε, θα έχουμε και άμεσες ε, αναδιανομές στο εσωτερικό της γεωργίας και της δικαιοσύνης μεταξύ των κρατών μελών. Αυτή η ιστορία δεν έχει τελειώσει ακόμα. Σε αντίθεση τώρα με τους προλαλήσαντες από το ΕΛΚ και τον κύριο που μόλις μίλησε, που είπε πως δεν είναι σωστό να πάμε σε ένα 30% πρασινίσματος, είναι καλό εγώ θεωρώ να το συζητάμε και αυτό το 30% είναι εγγύηση για το ότι θα διατηρηθεί σε αυτό το ύψος ο προπολογισμό. Θα φύγουμε δηλαδή από τη λογική της ε, αντιστάθμισης ότι πληρώνονται για κάποια παραγωγή και πληρώνονται θα λέμε για κάποια περιβαλλοντική ε, επίδοση και υπηρεσία οι αγρότες και άρα έτσι θα ε, μπορέσει να διατηρηθεί ο προπολογισμός στο ίδιο ύψος. Τώρα ένα ερώτημα για τους πυλώνες και την αρχιτεκτονική αν θέλετε. Πράγματι ο δεύτερο πυλώνα ε, ευτυχώ έμεινε στο ύψο που ήταν, αν και εγώ θα ήθελα να ισχυθεί ακόμη περισσότερο. Αλλά εντό ε, του δεύτερου πυλώνα, και αυτό πρέπει να είναι σαφές, δεν μπορεί να έχουμε ε, κονδύλια από το δεύτερο πυλώνα να πηγαίνουν η ενίσχυση του πρώτου. Πρέπει να υπάρχει μια σαφή δομή και αναμένω στη μεταρρύθμιση που θα γίνει όλες οι χώρες ε, να έχουν ένα δεύτερο ισχυρό πυλώνα με περιβαλλοντικά προγράμματα, αηφορία. Είναι πυρήνα κοινή γεωργικής πολιτικής και δεν μπορούμε να πάρουμε αυτά λεφτά και να τα δώσουμε στον πρώτο πυλώνα. Επίσης το πρόγραμμα Leader βασικό πρέπει να διατηρηθεί και να επεκταθεί. Θεωρώ Ναι, εντάξει, καλά τα κονδύλια για την έρευνα στον τομέα της γεωργίας, αλλά τίθεται εδώ πέρα το ερώτημα πού πάνε τελικά. Δεν ε, νομίζω να είναι, κύριε Νίκολσον, ε, κάποιο αντίτιμο για τις ε, διαπραγματεύσεις Μερκοσούρ. Νομίζω πως ερευνούμε για την γεωργία του μέλλοντος γιατί η γεωργία θα είναι βασικό για, θέμα για τα επόμενα χρόνια. Ερωτήσεις, ε, πράγματι έχω και εγώ όπως και οι πόσο σίγουρα είναι τα κονδύλια για την παγκοσμιοποίηση, πού πηγαίνουν και πώς μπορούν να διατεθούν. Είναι κάπως ανοιχτό το θέμα. Και με ποια μορφή τώρα για τις, ε, την κινητοποίηση την ε, διακύμανση των ε, τιμών δεν ξέρω αν μπορούμε να τα χρησιμοποιήσουμε. Εγώ πάντως είμαι πεπισμένος πως είμαστε σε καλό δρόμο με κονδύλια τα οποία δεν αυξάνονται αλλά εν πάση περιπτώσει αν διατηρηθούν νομίζω μπορούμε να είμαστε ικανοποιημένοι και ούτως ή άλλως συνολικά ε, το ερώτημα για τη διατήρηση αφορά ολόκληρο τον προπολογισμό γιατί είναι και απόφαση των κρατών μελών, είναι συναρπαστικό, ακόμα και δεν έχει απαντηθεί και όπως είπαμε οριστικό δεν είναι τίποτα. Ευχαριστούμε, Λορέντσο Φοντάνα. Ευχαριστώ, Πρόεδρε και ευχαριστώ και τον Επίτροπο για την παρουσία του. Εγώ, κύριε Επίτροπο, είμαι πραγματικά επεπισμένο ότι εσεί βάλατε τα δυνατά σα για να υπερασπίσετε τον προπολογισμό τη κοινή αγροτική πολιτική, ακόμη και αν είναι προφανέ ότι από τη δική μα σκοπιά Έχουμε πραγματικές περικοπές, όπως είπατε και εσείς. Τώρα το μπαλάκι είναι και στο δικό μας γήπεδο και εμείς ως Επιτροπή και ως Κοινοβούλιο ε, θα προσπαθήσουμε να δώσουμε όθηση και στις δικές μας θέσεις στο ιστορικό του Κοινοβουλίου. Χαίρομαι που υπάρχει αυτό το Ταμείο ε, της Παγκοσμιοποίησης, αλλά και εγώ θα ήθελα να μάθω κάποιες περισσότερες λεπτομέρειες για το θέμα αυτό, γιατί νομίζω ότι ε, το μέλλον της Ευρώπης και της Ευρωπαϊκής Γεωργίας θα βασιστεί ιδιαίτερα σε αυτό, δηλαδή αν η γεωργία μας θα μπορέσει να αντιμετωπίσει ε, τον αντίκτυπο του παγκοσμίου εμπορίου λόγω της παγκοσμιοποίησης γιατί βλέπουμε ότι πολλά προβλήματα τέτοιου χαρακτήρα αντιμετωπίζουν ήδη οι γεωργοί μας. Ε, και μια ερώτηση. Εσείς κάνετε πολύ καλή δουλειά αλλά συνεχίζουμε να ακούμε ότι θα πρέπει να υπάρχουν περικοπές στην ΚΑΠ, ότι δεν έχει τόσο η γεωργία σήμερα όπως παλιά. Εγώ θέλω να σα ρωτήσω, στην Ευρώπη δηλαδή, ε, να, κάποιοι να πούν ε, ότι θα περικόψουμε τη γεωργία για να προωθήσουμε έναν άλλο τομέα, γιατί οι φίλοι μου οι αγρότε που δεν μπορούν να πουλήσουν τα προϊόντα τους γιατί έχουν πολύ ψηλό κόστο παραγωγή που ξεπερνά τι δαπάνε. ε, αναρωτιέμαι μήπως υπάρχει βούληση από την πλευρά κάποιου, όχι δική σας η δική μας φυσικά, αλλά κάποιος έχει αυτή τη βούληψη να καταστρέψει την Ευρωπαϊκή Γεωργία, αν υπάρχει κάτι τέτοιο. Εγώ εύχομαι φυσικά να μην ισχύει, αλλά αν ναι, ισχύει κάτι τέτοιο, θα ήθελα εμείς να κάνουμε κοινό μέτωπο για να αντιμετωπίσουμε αυτό το θέμα και να υπερασπίσουμε την Ευρωπαϊκή Γεωργία. Ο κύριος Ρούμπιξ. Ευχαριστώ. Θα ήθελα και εγώ να συμφωνήσω με τους ε, συναδέλφους που αναφέρουν το ότι ε, πράγματι χαιρόμαστε που συνομιλούμε με τον κύριο Επίτροπο. Έρχεστε πάρα πολύ συχνά εδώ πέρα, μιλάμε ανοιχτά μεταξύ μας, αλλά ταυτόχρονα κατέληξα στο συμπέρασμα πως ε, όσο το συντομότερο φτάσουμε στη στιγμή όπου θα πρέπει να ανταποκριθούμε στις ε, υποσχέσεις μας και να βασιστούμε σε πραγματικούς ε, και κονδύλια. Όσο πιο κοντά φτάνουμε σε αυτή τη στιγμή, τόσο πιο πολύ αδειάζει το πορτοφόλι μας. Σας έχω ρωτήσει επανειλημμένα πώς μπορώ να εξηγήσω στους ψηφοφόρους μου στην Λετωνία το ότι εμείς λαμβάνουμε τις χαμηλότερες άμεσες πληρωμές ε, σε ολόκληρη την Ευρωπαϊκή Ένωση. Είμαστε 27 27. Έχουμε πει πολλές φορές πως πρέπει να εξισωθούν οι πληρωμές. Έχουμε βοηθήσει όσους ε, είχαν μείνει πίσω και εξακολουθώ να διαβάζω και να βλέπω πως μέχρι το 2020 οι Λετωνοί αγρότες ε, θα λαμβάνουν 52% του μέσου ευρωπαϊκού επίπεδου σε άμεσες ε, πληρωμές. Δεν μπορώ να το εξηγήσω αυτό τους ψηφοφόρους μου και βεβαίως ο τύπος είναι επιθετικός στη Λετωνία. Δεν ξέρω, ίσως και εμείς να πρέπει να ανταποκριθούμε κατά 52% στις υποχρεώσεις μας, αν είναι έτσι. Δηλαδή ε, ο κόσμος ε, δεν ξέρει τι να κάνει πλέον. Ε, αντιμετωπίζει πρόβλημα επιβίωσης. Υπάρχουν πολλά σημεία εντός του προϋπολογισμού και μπορούμε βεβαίως να μετατοπίζουμε από τον ένα τύλο στον άλλον τα κονδύλια. Είναι δυνατόν αυτό εντός του προϋπολογισμού, το αντιλαμβάνουμε, αλλά τι πρέπει να κάνουμε εμείς για να λυθεί αυτό το πρόβλημα και να υπάρχει επαρκής ε, χρηματοδότηση. Πρέπει να θυμόμαστε πως ε, η κοινή γεωργική πολιτική και ο Γεωργία γενικός είναι μία από τις σημαντικότερες κοινέ πολιτικές που κρατάει την Ευρωπαϊκή Ένωση Ενωμένη. Και δεν μπορούμε με υποσχέσεις ε, ανεκπλήρωτες να ε, υπονομεύουμε την εμπιστοσύνη στην Ευρωπαϊκή Ένωση. Και ελπίζω λοιπόν μαζί να μπορέσουμε να έχουμε κάποια θετικά αποτελέσματα. Πολύ ωραία. Σας ευχαριστούμε για αυτό το πρώτο γύρο ε, σκέψεων και τοποθετήσεων από τους συντονιστές. Εγώ θα δώσω τώρα το λόγο στον Επίτροπο για να μπορέσει να δώσει κάποιες απαντήσεις και κατόπιν θα συνεχίσουμε δίνοντας το λόγο στους υπόλοιπους συναδέλφους. Παρακαλώ κύριε Επίτροπε. Ευχαριστώ. Λοιπόν, θα αναφερθώ στις ερωτήσεις ε, μία προς μία. Ο κύριος Ντες ε, είπε ότι ΚΑΠ είναι η μόνη πολιτική η οποία δέχτηκε περικοπές. Εφαρμόσαμε τους ίδιους τρόπους υπολογισμούς ε, και για την ε, ΚΑΠ και για τη συνοχή, δηλαδή ονομαστικά ο πάγωμα χωρίς υπολογισμό του πληθωρισμού και σας υπενθυμίζω ότι εγώ με προσοχή διάβασα την έκθεση του Κοινοβουλίου που προτίθηκε από την Επιτροπή ΣΟΥΡΕ και εκεί είπαμε, υπόθηκε διατήρηση του προπολογισμού της ΚΑΠ χωρίς να δίνονται λεπτομέρειες για τον πληθωρισμό και τον υπολογισμό του. Και ξέρω ότι υπήρχαν κάποιες τροπολογίες προς την κατεύθυνση αυτή, όμως δεν εγκρίθηκαν οι τροπολογίες αυτές. Έτσι λοιπόν η Επιτροπή έλαβε αυτό το αίτημα του Κοινοβουλίου και το εφάρμοσε και για την ε, πολιτική συνοχή και για την ΚΑΠ. Και αν για την πολιτική συνοχή ε, δείτε τα 50 δις ευρώ σε τρέχουσα αξία ε, που εκταμιεύονται για τα μέσα υποδομής Connecting Europe συνδέοντας στην Ευρώπη θα δείτε ότι και η πολιτική συνοχή βρίσκεται στην ίδια κατάσταση μόνο που στη συνέχεια δημιουργήσαμε ένα σύνδεσμο μεταξύ αυτού του δημοσιονομικού φακέλου για την πολιτική συνοχή, γιατί ένα τμήμα αυτού του δημοσιονομικού φακέλου που αφορά το Interconnecting Europe ε, θα έρθει από την πολιτική συνοχή. Δεν θέλω να πω τώρα σε λεπτομέρειε, αλλά αν δούμε το καθαρό ποσό για την πολιτική συνοχή και το καθαρό ποσό για την ΚΑΠ, έχουμε εφαρμόσει την ίδια μέθοδο. Και για το λόγο αυτό, όπως σας είπα, με την δημοσιονομική, τη συνολική δημοσιονομική κατανομή. Η ΚΑΠ μένει στην πρώτη θέση. Είναι η πολιτική που χρηματοδοτείται περισσότερο από τον κοινοτικό προπολογισμό. Αν ε, θέλετε λοιπόν, είναι η ίδια η ταξινόμηση τελικά. Τώρα για την πράσινη βίβλο, για την προώθηση. Θα παρουσιάσουμε αυτή την πράσινη βίβλο και φυσικά σκοπεύω να χρηματοδοτήσω την ε, προώθηση Νομίζω ότι με την εκταμείευση που θα έχουμε στη διάθεσή μα θα μπορέσουμε να χρηματοδοτήσουμε και μια πολιτική πρόθεση. Η πρόθεσή μα τουλάχιστον παραμένει ίδια. Στην ανακοινώση αναφέραμε ορισμένε λεπτομέρειε ακριβώ για να δείξουμε το ότι ΚΑΠ είναι μια πολιτική η οποία ανοίγεται και σε άλλου τομεί ε, και συμπεριλαμβάνει και τι προσδοκίε που μπορούμε να έχουμε για άλλου ε, τομεί, περιβάλλον, ε, παραδείγματο χάρη, κλιματική αλλαγή. Και αντί να επιτίθετε στην Κομισιόν για να λέτε δεν λάβατε υπόψη αυτές τις φιλοδοξίες που βάζετε στη Στρατηγική Ευρώπη 2020, δείξαμε, και το έχουμε πει επανειλημμένω και στι δύο εδώ, ότι η ΚΑΠ ε, είναι μια τομεακή πολιτική με ε, πολυτομεικέ συνέπειε και έχουμε συμπεριλάβει κάποια στοιχεία για να δείξουμε ακριβώ ότι η ΚΑΠ ε, έχει τη φιλοδοξία να πετύχει ορισμένου στόχου ε, που συμπεριλαμβάνονται στη στρατηγική Ευρώπη 2020 με πολύ συγκεκριμένο τρόπο. Και εσεί επαναλημμένα είπατε ότι ο στόχο τη ΚΑΠ πρέπει να διασφαλίζει, να είναι διασφάλιση με συγχωρείτε τη επιστημιστική ασφάλεια και να ευθυγραμμιστεί καλύτερα με του στόχου ε, Ευρώπη 2020 με ορισμένα στοιχεία που έχουμε δώσει στην νομοθετική πρόταση, αυτό υπογραμμίσαμε, χωρίς να μπαίνουμε υπερβολικά σε λεπτομέρειε. Γι' αυτό βάλαμε αυτό το ποσοστό του περσινίσματος ε, και το περιεχόμενο αυτού του περσινίσματος ε, θα το συζητήσουμε μαζί σας. Ε, θα παρουσιαστεί και στις νομοθετικές προτάσεις. Θα έχουμε τον τρόπο εφαρμογής. Πάντοτε εγώ επιθυμώ να έχουμε μία απλή εφαρμογή, χωρίς ιδιαίτερη γραφειοκρατία, αλλά δείξαμε ότι η ΚΑΠ μπορεί να απαντήσει και να καλύψει στόχου στόχους αυτούς. Ε, κύριε Ντέ, ε, δεν παρουσιάσαμε κατανομή μεταξύ των κρατών μελών. Στι δημοσιονομικέ προοπτικέ ε, δεν υπάρχουν τέτοια στοιχεία. Αυτό θα γίνει με τη μεταρρύθμιση τη ΚΑΠ. Απλώς έχουμε βάλει το συνολικό ποσό, τα ποσά για τον πρώτο και το δεύτερο πυλώνα και είχαμε πει μαζί με τη δυνατότητα σε ορισμένες ε, περιπτώσεις να έχουμε μεταφορές από τον ένα στον άλλο τομέα για να ε, μην ε, παγώσουμε τη συζήτηση γύρω από την χρηματοδότηση της ΚΑΠ. Γιατί αυτό το fine tuning, ο συντονισμός θα πρέπει να γίνει στο τέλος. Μπορεί να γίνουν κάποιες προσαρμογές για το τάδε κράτος μέλος ή το άλλο κράτος μέλος για να φτάσουμε στη συμφωνία. Ξέρετε υπάρχουν ιδιαιτερότητες μεταξύ των κρατών μελών. Δεν θέλαμε ε, να δέσουμε τα χέρια της Κομισιόν, ε, καταρχήν και στη συνέχεια του Συμβουλίου και του Κοινοβουλίου στις διαπραγματεύσεις. Αλλά το διευκρινίσαμε και σας το λέω εδώ. Δεν ε, πρόκειται για ευελιξία που θα δώσουμε στα κράτη-μέλη αιώνια, δηλαδή να μεταφέρουν όπω θέλουν τα κονδύλια από τον πρώτο στο δεύτερο πυλώνα. Τα ποσά για τους δύο πυλώνες αυτούς θα καθορίζονται με σαφήνεια για το κάθε κράτος μέλος στο νομοθετικό πακέτο, στο νομοθετικέ δέσμη μέτρων που θα προτείνουμε για τη μεταρρύθμιση τη ΚΑΠ αλλά αφήσαμε εδώ αυτή τη δυνατότητα να μπορέσουμε ε, να το διαπραγματευτούμε όταν θα εκπονούμε το ίδιο νομοθέτημα. Αυτή την δυνατότητα την έχει ο Επίτροπος Γεωργίας, τις προτάσεις που θα σας υποβάλει, ε, να έχει αυτή την ευελιξία και μπορεί να κινηθούμε προς την πίδη ή την τάδε κατεύθυνση. Είπαμε, αυτή είναι η ιδέα δική μου δηλαδή, ότι τα κονδύλια που μπορούμε να λάβουμε με την εφαρμογή του ανώτατου ορίου να τα μεταφέρουμε το χάρη από τον πρώτο στο δεύτερο πυλώνα για τη χρηματοδότηση ορισμένων μέτρων. Και εδώ χρειαζόμαστε αυτή την ευελιξία στις συζητήσεις. Γι' αυτό βάλαμε αυτή τη φράση. Αλλά δεν μιλάμε για αιώνια ευελιξία για τα κράτη-μέλη πρόκειται για ευελιξία για όσου λαμβάνουν τι αποφάσει σε ευρωπαϊκό επίπεδο όταν θα ληφθεί η απόφαση για τη μεταρρύθμιση τη ΚΑΠ. Λοιπόν, τώρα πώς ε, θα ενεργοποιηθούν ε, τα μέτρα για την εξκρίση της αγοράς. Αν διαβάσετε για το αποθεματικό. Ε, αν διαβάσετε το κείμενο, θα είδατε ότι αυτός ο φάκελο θα χρησιμοποιηθεί με τον ίδιο βαθμό ευελιξίας που έχουμε σήμερα για τις παρεμβάσεις της Κομισιόν σε περιπτώσεις κρίσης. Δηλαδή, ενεργοποίηση των πόρων πολύ γρήγορη, όπως γίνεται και σήμερα, στα πλαίσια της ΚΑΠ, όταν χρειάζεται. Η διαδικασία είναι γρήγορη και δεν χρειάζεται να ληφθούν γραφειοκρατικές αποφάσεις. Αλλά θα θυμάστε και γιατί είναι σημαντικό να έχουμε αυτό το επαθηματικό για την αντιμετώπιση της ε, κρίσης στην αγορά που είναι εκτός ε, του συνολικού προεπλογισμού που περιλαμβάνονται και άμεσες ενισχύσεις και άλλα είδη μέτρων αγοράς. Θα θυμάστε ότι συχνά, σχεδόν κάθε χρόνο, έχουμε ποσά στον πρώτο πυλώνα που δεν είχαν χρησιμοποιηθεί γιατί δεν ε, είχαμε τέτοιες καταστάσεις, κρίση στην αγορά δηλαδή, και είχαμε τις μειώσεις ε, στον πρώτο πυλώνα, μεταφορά για άλλες δαπάνες και δίναμε και την εντύπωση προς τα έξω ότι η ΚΑΠ έχει πάρα πολλά χρήματα ε, και δεν μπορεί να τα δαπανίσει. Ξέρετε πολύ καλά ότι αυτά τα ποσά που είχαν εκτεμιευτεί για τη διαχείριση των αγορών ε, όταν δεν είχαμε περιπτώσεις κρίσης δεν τα χρησιμοποιούσαμε. Τώρα το ότι τα βάζουμε αυτά ξεχωριστά από τις άμεσες ενισχύσεις ε, μας οδηγεί στο να έχουμε ξεκάθαρα τις δαπάνες που θα είναι πάνω κάτω σταθερές και στις ε, άμεσες ενισχύσεις ξέρετε ότι για τον πολιτικό τομέα έχουμε δαπάνες που είναι σταθερές πάνω κάτω και έχουμε και ένα τμήμα κειμενόμενο που το χρησιμοποιούμε όταν το χρειαζόμαστε. Έτσι λοιπόν ένα μεγάλο τμήμα τώρα αυτού του δημοσιονομικού φακέλου που δεν είναι σταθερός θα διαχωριστεί τώρα από τη γραμμή του υπολογισμού που αφορά τις άβασες ενισχύσεις αλλά θα φυλάσσεται για τη γεωργία. Και ξέρετε ότι έχουμε όλο και περισσότερες κρίσεις στην αγορά ε, λόγω ε, κρίσεως στον τομέα των υγειονομικών. Και ξέρετε ότι κάτι τέτοιο λοιπόν θα μας διευκολύνει να διαχειριζόμαστε την κατάσταση. Και όπως σας είπα, αυτό το ποσό θα χρησιμοποιείται με ευέλικτο και γρήγορο τρόπο. Θα είναι πολύ γρήγορη η ενεργοποίησή του. Τώρα για το αποθεματικό λοιπόν αυτό και για το Ταμείο για την Παγκοσμιοποίηση. Με ρωτήσατε πώς θα χρησιμοποιηθεί αυτό το Ταμείο για την παγκοσμιοποίηση. Πράγματι χρειάζεται να έχουμε συγκεκριμένε νομοθετικέ προτάσει για να διευκρινίσουμε σε ποιες περιπτώσεις και με ποιο τρόπο χρησιμοποιούμε αυτά τα κονδύλια. Έτσι λοιπόν θα παρουσιάσουν δυο συγκεκριμένε προτάσει, γιατί καθώ είναι πρώτη φορά που έχουμε αυτή τη δημοσιονομική γραμμή, αυτή τη γραμμή του προπολογισμού, θα πρέπει να έχουμε και εκπόνηση νομοθεσία. Αλλά αυτό το ταμείο για την αντιμετώπιση τη παγκοσμιοποίηση, κύριε Νίκολσον, σα διαβεβαιώνω ότι η δική μου θέση για τι ε, διεθνεί ε, συμφωνίε δεν έχει αλλάξει. Εγώ παρακολουθώ πολύ προσεκτικά αυτέ τι ε, διαπραγματεύσει. Δεν βάλαμε αυτό το ταμείο για την παγκοσμιοποίηση, ε, για να είμαστε πιο ευέλικτοι τώρα στις διαπραγματεύσεις. Εγώ θεωρώ ότι οι απώλειες που οφείλονται σε κακές διαπραγματεύσεις των εμπορικών συμφωνιών δεν μπορούν να αντισταθμιστούν με ένα ταμείο για την παγκοσμιοποίηση, ένα άλλο είδους ταμείο αλλά εμπορικές συμφωνίες που μπορεί να τύχουν καλής διαπραγμάτευσης και να έχουν πραγματικά αντίκτυπο μας οδηγούν σε μια άλλη κατάσταση πέρα από τις ε, διαπραγματεύσεις. Κάποια στιγμή, κάποιο έτος, βλέπουμε ότι ε, υπάρχει επίπτωση στο εισόδημα των γεωργών επειδή μπορεί να υπάρχει κερδοσκοπία αστάθεια στις τιμές σε παγκόσμιο επίπεδο και μέχρι τώρα στο δικό μας προπολογισμό στην ΚΑΠ δεν έχουμε ούτε δημοσιονομική γραμμή ούτε νομική βάση για να μπορούμε να αποζημιώσουμε τους γεωργούς για τέτοιες απώλειες εισοδήματος που οφείλονται σε διακυμάνσεις ε, των τιμών στην παγκόσμια αγορά και όχι στην ευρωπαϊκή αγορά. Έτσι λοιπόν, αυτό το ταμείο όταν ε, θα έχουμε και το νομικό πλαίσιο για να το χρησιμοποιήσουμε θα μπορεί να ενεργοποιηθεί σε ένα πολύ ευρύτερο πλαίσιο. Ε, όχι μόνο στα πλαίσια των διεθνών εμπορικών συμφωνιών. Γι' αυτό στην ανακοίνωση έχουμε αυτόν τον ευρύτερο ορισμό και δεν το περιορίσαμε στις εμπορικές συμφωνίες. Εξήγησα όμως ότι κατά την άποψή μα και βάσει των υπολογισμών που κάναμε, αν δείτε την πολιτική συνοχή ε, και την ΚΑΠ, Δίχω ε, το Connecting Europe, η μέθοδο υπολογισμού είναι ίδια. επειδή οι ορισμένε ε, δαπάνε εξήχθησαν τον πρώτο πυλώνα και πήγαν σε άλλε γραμμέ προπολογισμού. Σα είπα ότι έχουμε το απαραίτητο ποσό, λίγο παραπάνω από 9 δι σε τρέχουσα αξία, για να μπορούμε να χρηματοδοτήσουμε το phasing in για τα νέα κρατημέλη, χωρί αυτό να θίξει τι άμεσε ενισχύσει για τα άλλα κρατημέλη. Τώρα χρηματοδοτούμε αυτή τη σταδιακή εισαγωγή, το phasing in, με την εφαρμογή του 1% πληθωρισμού για τον πρώτο πυλώνα. Δεν έχουμε αυτό το 1% για τον πρώτο πυλώνα, αλλά αφαιρέσαμε τα απαραίτητα ποσά βάζοντάς τα σε άλλες γραμμές του προπολογισμού. Έτσι λοιπόν, χωρίς να θίγονται οι καθολικές πληρωμές για τους υπόλοιπους, μπορέσαμε να διασφαλίσουμε αυτή τη χρηματοδότηση για το phasing in. Τώρα για το Ταμείο για την Κρίση και για το Ταμείο Παγκοσμιοποίησης, σας είπα ότι θα χρειαστούν περαιτέρω νομικέ διευκρινήσεις για τη χρήση τους αλλά κατόπιν ε, τα κονδύλια που δεν θα χρησιμοποιηθούν ε, ε, θα έχουμε κάποια ευελιξία για να μπορέσουμε να χρησιμοποιήσουμε τα κονδύλια για άλλες προτεραιότητες. Όμως παρόλα αυτά στα πλαίσια της ΚΑΠ. Ο κ. Νίκολσον ρώτησε πώς διασφαλίζεται η επιστημιστική ασφάλεια βάσει του προπολογισμού. Υπάρχουν ε, πολλέ τέτοιε ερωτήσει ε, και θα απαντήσουμε ε, με τον τρόπο που θα προσδιορίσουμε την κάπη στο νομοθετικό πακέτο που θα προτείνουμε. Τώρα, αν θέλετε, έχουμε το καύσιμο. Νομίζω ότι είναι σημαντικό να μπορέσουμε να διασφαλίσουμε ότι έχουμε τα απαραίτητα καύσιμα, το ελάχιστο καύσιμο. Τώρα, όταν θα σχεδιάσουμε τη μηχανή, αν θέλετε, αυτή η νομοθετική δέσμη μέτρων της ΚΑΠ ε, είναι η μηχανή. Έτσι λοιπόν εκεί θα δούμε πώς αυτό το καύσιμο θα το χρησιμοποιήσουμε με τον πιο αποτελεσματικό τρόπο για να πετύχουμε τους στόχους που έχουμε θέσει. Αλλά Νομίζω ότι διατηρήσαμε, διφλάξαμε χρήματα για τις άμεσες ενισχύσεις και για το ότι προσθέσαμε και δημοσιονομικές ε, γραμμές καινούριε για να αντιμετωπίσουμε και συγκεκριμένε καταστάσει κρίση και τα αποτελέσματα τη παγκοσμιοποίηση και ότι έχουμε ε, προπολογισμό για το δεύτερο πυλώνα, νομίζω ότι ε, όλα αυτά στοχεύουν στην επιτεύξη των στόχων που έχουμε θέσει στην ανακοίνωση της ΚΑΠ και τις φιλοδοξίες που έχουμε στα πλαίσια της νομοθετικής μέτρων. Δεν ε, θέλαμε να παρουσιάσουμε πολλές λεπτομέρειες για τη μεταρρύθμιση στο δημοσιονομικό πακέτο, αλλά παρουσιάσαμε απλώ τα στοιχεία που μας δείχνουν με ποιο τρόπο ε, η ΚΑΠ ε, μπορεί να απαντήσει και σε άλλους στόχους που προβλέπονται στη στρατηγική για το 2020. Γι' αυτό έχουμε όλα αυτά τα διευκρινιστικά στοιχεία, όχι για κανέναν λόγο, αλλά φυσικά αφήνεται έτσι ένα περιθώριο ε, ευελιξίας ε, όταν θα διαπραγματευτούμε το νομοθέτημα, την νομοθετική πρόταση. Κύριε Ρέσλινγκ, ε, δεύτερο πυλώνα. Γι' αυτό βάλαμε με σαφήνεια τα ποσά για το δεύτερο πυλώνα, για να διασφαλίσουμε ότι διατηρούμε τη σημερινή αναλογία μεταξύ πρώτου και δεύτερου πυλώνα. Και σας επαναλαμβάνω, η μεταφορά μεταξύ πρώτου και δεύτερου πυλώνα και αντιστρόφω είναι απλώς ένα περιθώριο λιγμών που θα έχει ο νομοθέτης όταν θα ε, εκπονήσει την νομική βάση για τη μεταρρύθμιση της ΚΑΠ. Ε, δεν θα γίνει αυτό ε, δίνοντας αιώνια ευκαιρία στα κράτη-μέλη. Θα προσδιορίσουμε την κατανομή για το διάφορα κράτη-μέλη, για τον πρώτο και για το δεύτερο πυλώνα. Έτσι πρέπει να ερμηνεύσετε αυτή τη φράση με την ευελιξία της μεταφοράς μεταξύ των κρατών μελών. Λοιπόν, προπολογισμό για έρευνα και ανάπτυξη πώς θα γίνει η κατανομή. Και γι' αυτό θα προσδιορίσουμε την νομική βάση, θα παρουσιάσουμε μια ανακοίνωση για τις ε, ευρωπαϊκές εταιρικές σχέσεις καινοτομία, θα προσδιορίσουμε εκεί τις αρχές και κατόπιν ε, θα υπάρχουν οδηγοί εφαρμογής. Εκεί θα παρουσιάζονται οι λεπτομέρειες, όπως και να έχει όμως ε, η διαχείριση του προγράμματος αυτού θα είναι σε ευρωπαϊκό επίπεδο. Όμως το περιεχόμενο θα το προσδιορίσουμε στις μελλοντικές νομοθετικέ προτάσει. Κύριε Φοντάνα, Νομίζω ότι ο τρόπος με τον οποίο παρουσίασε η Κομισιόν τη θέση της ΚΑΠ ε, στον Ευρωπαϊκό Πολιτισμό Μα δείχνει ακριβώ το αντίθετο, ότι σε καμία περίπτωση δεν θέλουμε να εξελίψουμε τη γεωργία στην Ευρωπαϊκή Ένωση. Βλέπουμε με σαφήνεια ότι για την Ευρωπαϊκή Επιτροπή η ΚΑΠ παραμένει προτεραιότητα και για τι μελλοντικέ δημοσιονομικέ προοπτικέ. Έχουμε ε, την πρώτη δημοσιονομική θέση και έχουμε και συνεπή προπολογισμό παρά την δύσκολη οικονομική συγκυρία. Έχουμε μια κοινοτική πολιτική και ένα κοινοτικό προπολογισμό. Νομίζω ότι αυτό είναι ένα σαφέ πολιτικό μήνυμα προ την κατεύθυνση γιατί για τις έμεσες ενισχύσεις για ορισμένε χώρες. Δεν ε, προσδιορίσαμε εδώ την κατανομή των κονδυλίων για τη Λετωνία, τη και κάποια άλλη χώρα. Αυτό θα το πράξουμε στο νομοθετικό πακέτο. Δεν ε, ήταν ο στόχος ε, εδώ να προσδιοριστούν το επίπεδο των πληρωμών για κάθε χώρα ξεχωριστά. Θα γίνει αυτό στο νομοθετικό πακέτο. Αυτά είναι θα σα είχα να απαντήσω. Ευχαριστώ πολύ αγαπητέ επίτροπε. Πιστεύω ότι με αυτό το πρώτο γύρο ερωτήσεων και απαντήσεων ε, ήδη παρουσιάστηκαν πάρα πολλά στοιχεία. Τώρα θα ξαναδώσουμε το λόγο στους βουλευτές. 21 άτομα έχουν ζητήσει το λόγο. Έτσι λοιπόν σας παρακαλώ είστε σύντομοι. Ας ξεκινήσουμε με την ε, κυρία Ελίζα Πετιέκη. Ευχαριστώ. Θα προσπαθήσω λοιπόν να είμαι σύντομη κύριε Πρόεδρε. Κύριε Επίτροπε, στις απαντήσεις σας απαντήσατε σε πολλά ερωτήματα. Εγώ θα ήθελα να αναφέρω δύο σημεία που θα ήθελα να τονίσω. Το ένα είναι η σχέση πρώτου και δεύτερου πυλώνα, το πρασίνισμα, το οποίο επί της αρχής όπως ξέρετε υποστηρίζω και υποστηρίζω τα πολλά αγροπεριβαλλοντικά μέτρα που έχουν γίνει ήδη σε πολλά κράτη-μέλη. Για μένα αυτό είναι πάρα πολύ σημαντικό να μην υπάρχει εδώ πέρα διακριτική μεταχείριση των κρατών μελών εκείνων που σε τελική ανάλυση κάτι κάνουν και πως ε, συμφωνούμε νομίζω όλοι πως χρειαζόμαστε περισσότερο πρασίνισμα. Τώρα πως θα έχουμε έναν ε, ισχυρό δεύτερο πυλώνα και στο μέλλον. Πρώτα απ' όλα για τις περιοχές εκείνες ειδικά που δεν λαμβάνουν ε, κονδύλια από τα διαρθρωτικά ταμεία. Για αυτές τις περιοχές αυτά ο δεύτερος πυλώνας είναι κάποιες ε, δυνατότητες που έχουμε για να διαμορφώσουμε την κατάσταση, να έχουμε τον κόσμο με το μέρος μας. Και... Γιατί αλλιώ ξέρετε, είναι κάτι το επίμαχο η η γεωργική πολιτική. Επίσης αναφέρατε κάποια πράγματα ήδη για τις ε, διμερείς σχέσεις, αλλά το ότι ε, συζητιέται τόσο πολύ αυτό το θέμα στην Επιτροπή μας ε, σας δείχνει το ότι έχουμε ένα πρόβλημα και χαίρομαι για το ότι το παρατηρείτε και λέτε πως θα κάνετε κάτι, αλλά ξέρετε πως δεν είναι άτοποι οι φόβοι μας όταν λέμε πως ε, μία-μία η συμφωνία ίσως να μην είναι τόσο άσχημες, αλλά συνολικά πόσα ευρωπαϊκά γεωργικά προϊόντα θυσιάζονται εδώ πέρα και ε, αγρότες στο βωμό των ε, εμπορικών συμφωνιών και δεν ξέρω αν αρκεί το χρήμα για να το αντισταθμίσει και για το δημοσιονομικό πλαίσιο βίως διαπραγματευτήκατε όσο το δυνατόν καλύτερα μπορούσατε. Δεν επιτύχατε αυτά τα οποία θα θέλαμε όλα αλλά περισσότερα από αυτά τα οποία ήθελα να δώσουν κάποια κράτη-μέλη οπότε είναι πολύ καλό το, το αποτέλεσμα. Οπότε εγώ και πολλοί άλλοι οπωσδήποτε θα παλέψουμε μαζί σας για αυτό τον προϋπολογισμό. Χρειαζόμαστε κάποια κοινά λοιπόν επιχειρήματα. Σας ευχαριστώ. Ευχαριστώ. Στεφάν Λεφόλ. Μετά ο Αντιπρόεδρος Βοητσεχόφσκι. Ευχαριστώ κύριε Πρόεδρε και ευχαριστώ τον Επίτροπο που ήρθε τόσο γρήγορα να μας παρουσιάσει τις θέσεις του για τον προϋπολογισμό. Θα ήθελα να πω ότι όλοι συμφωνούμε ότι αποφύγαμε τον όλεθρο. Αν μη τι άλλο, αυτό είναι θετικό. Πάντως, ως Ευρωβουλευτής και το Κοινοβούλιο γενικώ, το είπε και η Επιτροπή ΣΟΥΡ, δεν έχει τελειώσει ο αγώνας, η μάχη για τον προϋπολογισμό. Αυτό που μας περιμένει είναι η συνέχεια της μείωσης του προϋπολογισμού. Δεν χρειάζεται να μιλάμε μόνο για την γεωργική πολιτική. Η δημοσιονομική μάχη είναι γενική. Και σίγουρα η πιο μαχητική ε, θα πρέπει εδώ να είναι η Ευρωπαϊκή Επιτροπή, άσχετα από τον Επίτροπο Γεωργίας. Αυτή είναι η συζήτηση. Ας δούμε την πραγματικότητα κατά πρόσωπο. Και αν ε, καταφέρουμε να κρατήσουμε ένα πάγωμα στη γεωργική χρηματοδότηση, θα μειωθεί ο προπολογισμό των διαρθρωτικών ταμείων. Είπαμε πριν ότι ε, κάποιες χώρες που δεν ε, Εποφελούνται από το Ταμείο Συνοχή, ούτε στο μέλλον θα το, το φυσικά. Υπάρχει μια ευρεία συζήτηση για τον προπολογισμό και φυσικά αγγίζει και τη Γεωργία. Μέχρι στιγμή αποφύγαμε την καταστροφή και χαίρομαι γιατί χάρη σε εσά αποφύγαμε αυτή την καταστροφή, κύριε Επίτροπε. Τώρα, έχουμε λίγα καύσιμα, έχουμε λίγη βενζίνη, πρέπει να, να σχεδιάσουμε τον κινητήρα. Πολύ ωραία εικόνα που μα δώσατε. Υπάρχει όμω ένα πρόβλημα με το Ταμείο Παγκοσμιοποίηση, το θέλουμε όχι, είναι Ταμείο προσαρμογή μα επιβάλλει την παγκοσμιοποίηση, θα πρέπει να προσαρμοστούμε. Μιλήσετε για 2,7 δισεκατομμύρια. Ούτε καν 3 τρισεκατομμύρια δυναμικό δεν έχει αυτό το ταμείο. Πώ λοιπόν η γεωργία από μόνη τη θα απορροφήσει περίπου 70%. Δεν είμαστε ήσυχοι ότι θα τηρηθεί αυτό. Σε ό,τι αφορά το επιστηστικό σχέδιο για τους απόρους ή για τους πλέον έχοντας ανάγκη μπορούμε να ε, δεσμευτούμε ότι θα έχουμε μια πολιτική ελάχιστον αποθεμάτων ε, για την επιστημιστική ασφάλεια στην Ευρώπη. Νομίζω ότι είναι πολύ επίκαιρο αυτό το θέμα και πολύ σημαντικό. Σε ό,τι αφορά την κρίση της κρίσης, είπαμε να είμαστε ελαστικοί και ευέλικτοι και να διαφυλάξουμε τους μηχανισμούς ε, ε ρύθμισης όσο μπορούμε για να επιλύσουμε τα προβλήματα πρέπει να είμαστε λίγο πιο διορατικοί και να προλαμβάνουμε περισσότερο. Τώρα για το κινητήρα που είπατε, άκουσα τα επιχειρήματά για το πρασίνισμα. Θέλω κάποιες διευκρινήσεις ε, σε ό,τι αφορά την αυθύνουσα ε, ε, αποχώρηση ή την, το ανάτοτα όρια ή μια νέα διαδικασία της διαφοροποίησης ε, που ίσως ε, θα τροφοδοτήσει στο δεύτερο πυλώνα και γι' αυτό θα ήθελα ε, κάποιες ευκαιρίες και για τη σταδιακή μείωση. Ευχαριστώ Στέφαν. Τώρα ο Αντιπρόεδρος Βοητσεχόφσκι και μετά η κυρία Πατράου Νέβες. Ευχαριστώ. Δεν κρύβω ότι η πρόταση της Ευρωπαϊκής Επιτροπής με στεναχώρησε. Πριν από 7 χρόνια, το 2004, το 2005, προετοιμάσαμε, καταρτήσαμε τις ε, δημοσιονομικές προοπτικές για την περίοδο 2007-2013, είχαμε για τη Γεωργία μια σύγκριτα καλύτερη κατάσταση. Και είχαμε στην παραγωγή πλεονάσματα, ζάχαρη για παράδειγμα, είχαμε πλεονάσματα βουτύρου, γάλακτος. Τότε ήταν πλεονάσματα όλα. Κανείς ε, δεν μίλησε τότε για επιστηστική ασφάλεια. Λίγα χρόνια μετά, το 2007-2008, εμφανίστηκε η κρίση και άρχισαν, άρχισαμε με την ακρίβεια των τιμών να αντιμετωπίζουμε προβλήματα και τώρα έχουμε μια άλλη τελείως διαφορετική κατάσταση να μιλούμε για την επιστηστική ασφάλεια. Και δεδομένης αυτή τη κατάσταση. αντί να ενισχύουμε του γεωργού, αφαιρούμε ενισχύσει. Αυτό πραγματικά είναι αδιανόητο. Πιστεύω ότι είναι τελείω ακατάλληλη αντίδραση στι προκλήσει που αντιμετωπίζουμε. Μία τέτοια χρηματοδότηση για τη γεωργία δεν αρκεί. Δεν μπορεί να ανταπεξέλθει στι προκλήσει που έχει η γεωργία. Πραγματικά δεν καταλαβαίνω γιατί υιοθετούμε αυτή την στάση. Ένα άλλο ζήτημα αφορά την ταξινόμηση, την κατανομή των ε, πληρωμών μεταξύ των παλιών και νέων. Έχουμε τεράστιες ε, διαφορές στο επίπεδο πληρωμών. Αυτό που προτείνει η Ευρωπαϊκή Επιτροπή ε, δεν είναι κάποια εξισορρόπηση, είναι κάποια μείωση των διαφορών περισσότερο. Δεν είναι μια εξίσωση. Με ποια νομική βάση όμως ενεργούμε εδώ. Έχουμε τη συνθήκη της Λισαβόνας που εξασφαλίζει την ισότητα των κρατών μελών της Ευρωπαϊκής Ένωσης. Ε, γιατί έχουμε το 90% το 1 τρίτο, έχουμε διάφορους μαθηματικούς ε, χειρισμούς, αλλά ποια είναι η πραγματική νομική βάση για όλα αυτά και γιατί ε, αντιστρέφουμε εδώ την πολιτική μας. Γιατί στην Γεωργία ειδικά ισχύει ε, αυτή η παράλογη αρχή ότι βοηθούμε τους πλούσιους περισσότερο και λιγότερο τους φτωχούς. Μα είναι αντίθετο το θεμέλιο της Ένωσης. Η Ένωση σε, άλλα, σε άλλες βάσεις στηρίζεται. Είμαι κατά αυτής της προσέγγισης. Με τέτοιο εγχείρημα, αυτοί που έχουν πολλά θα έχουν λίγο λιγότερα, αλλά θα εξακολουθούν να έχουν πολλά, ε, ενώ αυτοί που έχουν λίγα θα εξακολουθούν να έχουν λίγο περισσότερα, αλλά πάλι θα είναι πολύ λίγα αυτά που έχουν. Νομίζω ότι είναι απαράδεκτη αυτή η προσέγγιση. Ευχαριστώ. Η κυρία Πατράου Νέβε και μετά ο κύριο Σλαβία. Ευχαριστώ κύριε Πρόεδρε και ευχαριστώ και τον Επίτροπο που ήρθε για να συνεχίσουμε το διάλογο, ευρύ διαφανή διάλογο για τον οποίο είστε διαθέσιμο απέναντι στο Ευρωπαϊκό Κοινοβούλιο. Οι πρώτε εξαγγελίε για την ΚΑΠ μιλούσαν για μία μείωση του προϋπολογισμού γύρω στο 10%. Σήμερα είπατε ότι θα καταφέρουμε να κρατήσουμε αμύωτο τον προπολογισμό χάρη σε μια ανακατονομή διαφόρων ποσών από άλλες δημοσιονομικές γραμμές. Θα ήθελα να εκφράσω κάποιες ανησυχίες και επιφυλάξεις ως προς την αισιοδοξία σας, κύριε Επίτροπε, και να σας θέσω και ορισμένες ερωτήσεις. Πρώτον, τι επιχειρήματα ή τι συγκεκριμένες δράσεις πρόκειται να αναλάβει η Ευρωπαϊκή Επιτροπή για να αποφύγει τις αρνητικές προβλέψεις πέραν της ανακατανομής των κονδυλίων. Έχετε και άλλες προτάσεις, άλλα μέτρα. Δεύτερον, πώς θα προ... μια πραγματικά πιο δίκαιη ΚΑΠ, διορθώνοντας τις ανισορροπίες που υπάρχουν σήμερα και μάλιστα σε μια γενικώ αρνητική συγκυρία. Το καθεστώς των άμεσων πληρωμών δεν θα επηρεαστεί, μας είπατε τι θα γίνει, θα γίνει πιο δίκαιο αυτό το σύστημα των άμεσων πληρωμών. Αυτό προσδοκούμε και στην Επιτροπή Γεωργίας. Τρίτον, τι επίπτωση θα έχουν συγκεκριμένα προγράμματα θα έχουν αυτές οι αρνητικές αμφιβολίες. Το ΠΟΖΕΙ, το πρόγραμμα ΠΟΖΕΙ, υποστηρίζει τις ε, γεωργικές δραστηριότητες ιδιαίτερα στις εξόχως απόκεντρες ε, ε, περιοχές που πλήττονται πολύ περισσότερο από την, λόγω της απομόνωσής τους και εξαιτίας της παγκοσμιοποίησης. Καλό θα ήταν να ενισχυθούν αυτά τα κονδύλια για να αντισταθμιστούν τα αρνητικά αποτελέσματα του, της εξάλληψης των ποσοστώσεων και της πιθανής σύναψης συμφωνίας Ευρωπαϊκής Ένωσης Μερκοσούρ. Ευχαριστώ κύριε Επίτροπε και περιμένω απαντήσεις στις τρεις συγκεκριμένες ερωτήσεις που υπέβαλα. Ευχαριστώ. Κύριε Λαβία, συγγνώμη, προηγείται ε, ο κύριο, η κυρία Καλνιέτε. Ευχαριστώ πάρα πολύ. Κύριε Πρόεδρε, κύριε Επίτροπε, πρώτα απ' όλα να σας ε, συγχαρώ και εγώ για το αποτέλεσμα που επιτύχατε με τη συνεργασία του Κοινοβουλίου σχεδόν καταφέραμε να διατηρήσουμε άθικτα τα κονδύλια της κοινή γεωργικής πολιτικής ε, λαμβάνοντας υπόψη βεβαίως και τα προγράμματα που περιλαμβάνονται σε άλλους τίτλους στον ε, κοινοτικό προϋπολογισμό. Πρέπει να σας πω όμως πως σοκαρισμένη είναι η γεωργοί στη Λετωνία με βάση τις αρχές για τον υπολογισμό των άμεσων πληρωμών όπω ορίζονται στις δημοσιονομικέ προοπτικέ και οι φωνέ που είχαμε από τη Λιθουανία και την Εσθονία επίση ε, μαρτυρούν πω και εκεί πέρα επικρατεί το ίδιο σοκ. Ναι, πράγματι έχετε δίκιο. Δεν ε, ορίζεται ξεκάθαρα τι ποσά θα δοθούν σε κάθε χώρα, αλλά οι γεωργοί μας ε, διαβάζουν και μπορούν να υπολογίσουν ποια θα είναι η άμεση πληρωμή που θα λάβουν με βάση αυτά τα στοιχεία και προτείνουν προτείνεται μάλλον να φτάσουν στο 1 τρίτο εντός 7 ετών. Ε, είναι απαράδεκτο αυτό και παραβιάζει αρχές και της αλληλεγγύης και της ίσης μεταχείρισης. Ε, ειδικά αν δούμε τους ε, στόχους που διακήρυξε 18 Νοεμβρίου η Κομισιόν, οι οποίοι διαβάζω αναφέρουν. Να διασφαλίσουμε πως οι ενισχύσεις της κοινής γεωρικής πολιτικής ε, μοιράζονται δίκαια μεταξύ όλων των ακροτών των κρατών μελών. Και εκεί πέρα προτείνουν σαφώς οι ευρωβουλευτές κάθε κράτος μέλος να λαμβάνει ένα υποχρεωτικό ποσοστό του μέσου δίκτυ των άμεσων πληρωμών και να οριστεί ένα ανώτατο όριο γι' αυτό. Εάν δούμε αυτή την πρόταση λοιπόν, τότε οι Λετωνοί αγρότες ακόμα και το 2020, δηλαδή 30 χρόνια μετά την πτώση του παραπετάσματος θα λαμβάνουν μόνο το 1 τρίτο της στρεμματικής ενίσχυσης ενός Ολλανδού ή Βέλγου αγρότη. Αυτό δεν είναι σωστό. Κανένα κράτος μέλος δεν θα πρέπει να λαμβάνει λιγότερο από 80% και περισσότερο από 120% της μέσης στρεμματικής ενίσχυσης. Και οι χώρες εκείνες οι οποίες λαμβάνουν σήμερα μόλις το 30% θα πρέπει να ξεκινήσουν ε, ήδη από το 2014 μια μεταβατική περίοδο. Οπότε θα ήθελα να σας ε, παροτρύνω να συνεισφέρετε σε αυτό τον στόχο και να αποτελέσετε μέλη του ίσου ανταγωνισμού η κοινή γεωργική πολιτική και εμείς θα σας υποστηρίξουμε. Μάλιστα, θα δώσουμε το λόγο αργότερα στον Επίτροπο για να απαντήσει. Παρακαλώ να συνεχίσουμε με τους ομιλητές, που λέει και μετά Παστάμκος. Ευχαριστώ, Πρόεδρε. Κύριε Επίτροπε. Τα δεδομένα που προκύπτουν από την παρουσίαση του πολιτού δημοσιονομικού πλαισίου η πρώτη εβδομάδα δέχτηκε ιδιαίτερα διάφορες ερμηνείες γιατί ε, η δυσκολία του υπολογισμού με αυτή τη μεταφορά των ποσών μεταξύ όσων σας ε, ζήτησε το Κοινοβούλιο σε ό,τι αφορά το πάγωμα των δαπανών ε, σε επίπεδα 2013 και σε σύγκριση με αυτό που είδαμε κατόπιν τα επίπεδα του 2011 για τους πόρους μας μπέρδευσαν κάπως και ίσως πρέπει να ξανακάνουμε τον υπολογισμό στο Κοινοβούλιο γιατί συνεχίζουμε να βλέπουμε πολύ μεγάλες διαφορές όπως ε, είπαν και πολλοί συνάδελφοι, δεν υπάρχει ιδιαίτερη ικανοποίηση και πιθανότατα περιμέναμε κάτι παραπάνω. Γνωρίζουμε βέβαια ότι σημειώθηκε μεγάλη πρόοδος Διανύθηκε πολλή δρόμο από τις ε, πρώτες ε, πληροφορίες που είχαμε από τον επίσημο έγγραφο. Όμως ε, παρόλα αυτά το αποτέλεσμα δεσμεύει όλο το Κοινοβουλίο σε συνεχή δράση υποστήριξη τη δική σας ε, δράση ε, για να ενισχυθούν οι πόροι για την ΚΑΠ. Και υπάρχει βεβαιότητα ότι θα έχει συμμάχους το Κοινοβούλιο. Τώρα σε δύο, για δύο πιο συγκεκριμένες πτυχές για να είμαι σύντομος. Ανησυχώ κάπως από μια πτυχή που αναφέραν πολλοί συνάδελφοι και που μάλλον θα μπορούσατε να εξηγήσετε εύκολα το θέμα του Ταμείου Παγκοσμιοποίηση. Γιατί εμεί έχουμε ήδη ένα Ευρωπαϊκό Ταμείο για την Προσαρμογή στην Παγκοσμιοποίηση που εφαρμόζεται σήμερα για το βιομηχανικό τομέα, αλλά αντίθετα με δυσκολία θα δούμε να εφαρμοστεί για τον αγροτικό τομέα. Αν ε, ε σήμερα χρησιμοποιείται, παραδείγματο χάρη, αν θα χρησιμοποιηθεί για να δοθεί ενίσχυση στου ανθρώπου που βγαίνουν από τη Γεωργία για να απασχοληθούν σε άλλου τομεί. Τώρα, σε ό,τι αφορά τη βοήθεια στου απόρου το άκουσα, αλλά νομίζω ότι μήπως ήταν ε, λάθος. Ε, ε, αναφερθήκατε σε 8 δισεκατομμύρια ευρώ, ενώ στις δημοσιονομικές προοπτικές βλέπω κάτι διαφορετικό. Ποια είναι τα πραγματικά νούμερα, 8 ή 2,5 δις, όπως βλέπουμε στις δημοσιονομικές προοπτικές. Και γιατί θα πρέπει να βρούμε και μια νέα νομική βάση και νομίζω ότι το Κοινοβούλιο βεβαίως θα βοηθήσει στην Κομισιόν να αντιμετωπίσει όλη αυτή την κατάσταση. Ο κύριος Παπαστάμκος, παρακαλώ, ένα λεπτό. Ε, ε, Ο κύριος Ολένιτσακ πρώτα. σε σχέση με την αφετηριακή απεσιοδοξία, αξιολογώ την πρόταση της Επιτροπής ε, ως μια εύλογη βάση διαπραγματεύσεων. Και πρέπει να γνωρίσουμε όλοι το ρόλο του Επιτρόπου, του κυρίου Τσόλος, σε αυτήν, στη διαμόρφωση αυτής της πρότασης. Και επίτροπε το ερώτημα είναι ανοιχτό, σαφές. Εάν προτίθεστε πράγματι να κινηθείτε με όρους ανωδικούς, ανωδικής κλιμάκωσης της πρότασης, αντιλαμβάνεστε ότι η Επιτροπή Γεωργίας στο Ευρωπαϊκό Κοινοβούλιο θα σας στηρίξει. Ε, αυτό πρέπει να γίνει απολύτως ε, κατανοητό. Αν όχι, θα δημιουργηθεί χάσμα στη μέχρι τώρα πάρα πολύ καλή διαθεσμική μας συνεργασία. Θεωρώ ότι η πρόταση για το, την επέκταση του εδαφικού πεδίου εφαρμογής του Ευρωπαϊκού Ταμείου Παγκοσμιοποίησης ότι αποτελεί ένα αντίδοτο, μια αντιστάθμιση, μια αντισταθμιστική στήριξη και έναντι των παραχωρήσεων στις οποίες προβαίνει ή προτίθεται να προβεί η Επιτροπή, η Κομισιόν στις εμπορικές διαπραγματεύσεις με τρίτες χώρες ή ομάδες χωρών. Και θα κάνω και εγώ μια ερώτηση ε, εισηγήσετε τη μεταφορά του προγράμματος σύντησης απόρων από την ε, ΚΑΠ στο Heading 1, ε, δηλαδή στο κοινωνικό ταμείο. Αυτό θα σημάνει και συγχρηματοδότηση εκ μέρους των κρατών μελών. Ευχαριστώ κύριε Πρόεδρε. Ολενίτσκα. Κύριος Ολενίτσακ. Ευχαριστώ. Ε, κατάλαβα από τις απαντήσεις σας κύριε Επίτροπε ότι είστε ικανοποιημένο με την πρόταση που προβάλλεται μετά από διαπραγματεύσεις ε, ως πρόταση Ευρωπαϊκής Επιτροπής. Και αν αυτό είναι ο στόχος, αν αυτό είναι το τέλος, θα μπορούσαμε να είμαστε συγκρατημένα ικανοποιημένοι. Αλλά μόνο συγκρατημένα, γιατί ξέρουμε ότι μόνο στην αρχή των διαπραγματεύσεων βρισκόμαστε ακόμη, στην αφετηρία τους τι θα κάνουμε αν όπως φημολογείται είτε στο Συμβούλιο είτε και εδώ ο προϋπολογισμός ε, για, τις, για την κοινή πολιτική συρρυκνωθεί μετά τις τελευταίες διαπραγματεύσεις ε, στο Συμβούλιο. Τότε υπάρχουν κάποιες, εκεί σε τέτοια περίπτωση θα υπήρχαν κάποιες δυνατότητες ε, ευελιξίας, ελαστικότητας. Άλλο θέμα τώρα. Η πρόταση που καταθέσατε για την ε, ευελιξία μεταξύ πρώτου και δεύτερου πυλώνα φαίνεται εκ πρώτης όψεως ενδιαφέρουσα. Καλή, καλή ιδέα, αλλά μας ενδιαφέρουν περισσότερο οι λεπτομέρειες και μέχρι ποιο βαθμό μπορούν τα κράτη-μέλη στο σχεδιασμό ε, των, ε, των επόμενων δημοσιονομικών προοπτικών να χρησιμοποιήσουν αυτή την ευελιξία. Και η πρόταση που υποβάλλεται για το Ταμείο για την ε, καινοτομία και την ανάπτυξη της έρευνας ε, σε σχέση με τη γεωργία. Πολύ καλή αυτή η πρόταση και καλό θα είναι αυτό το σχέδιο να έχει ευρωπαϊκό χαρακτήρα και φυσικά περιμένουμε και γι' αυτό περισσότερες λεπτομέρειες. Τι μορφή θα έχει αυτό το πρόγραμμα, το σχέδιο στήριξης ε, της καινοτομίας και της έρευνας στη γεωργία. Και μια άλλη ερώτηση. Η Ευρωπαϊκή Επιτροπή κάνει κάποιες προσωμιώσει με βάση την πρόταση του προπολογισμού που κατέθεσε. Το 2013 κλείνει η επταετία ε, ε, των προοπτικών αυτών και οι γεωργοί θα λάβουν κάποια ποσά. Και με βάση τις ε, εκμεταλλεύσεις ξέρουν ότι περιμένουν μια συγκεκριμένη ενίσχυση από την Ευρωπαϊκή Ένωση. Τώρα, η πρόταση που υποβάλλατε σήμερα, τι μορφή θα έχει μετά το 2013. Θα είναι συγκρίσιμα τα ποσά αυτά μεταξύ των γεωργών, για αυτές οι ποσοστώσεις. Γιατί ε, θα είναι συγκρίσιμα με τα σημερινά επίπεδα αυτά τα κονδύλια ή από ό,τι ακούσαμε θα είναι αισθητά πιο μικρά. Ο κύριος Σεκέρσκι Κύριε Επίτροπε, δεν νομίζω ότι το πάγωμα του γεωργικού προϋπολογισμού είναι καμία επιτυχία. Δεν είναι επιτυχία. Αποτυχία είναι. ήττα είναι το πάγωμα του γεωργικού προϋπολογισμού. Γιατί έχουμε νέες προκλήσεις ε, και νέα, νέες υποχρεώσεις απέναντι στις νέες χώρες που πρέπει να τις χρηματοδοτήσουμε. Έχουμε συγκεκριμένες υποχρεώσεις και δεσμεύσεις που έχουμε αναλάβει και έχουμε και νέους στόχους για την κοινή γεωργική πολιτική. Από τη στιγμή που έχουμε νέες προκλήσεις, νέους στόχους, νέες δεσμεύσεις, πώς είναι δυνατόν να τις χρηματοδοτήσουμε από έναν παγωμένο προϋπολογισμό. Και σε πραγματικούς όρους έχουμε και μείωση. Είπαμε και προσπαθήσαμε να συζητήσουμε την Ευρωπαϊκή Επιτροπή, πώς θα γίνουν οι κατανομές, τι θα δώσουμε σε ποιον και ο κύριος Ντες και άλλοι το επισήμαναν, αλλά έχουμε και τη σχετική έκθεση. Προσπαθήσαμε να δούμε πώς θα ταξινομήσουμε τα ποσά ώστε να κρατήσει κανένας αυτό που είχε, αλλά και να μην έχουμε και γενικότερη αύξηση. Αυτό όμως δεν γίνεται. Επίσης έχουμε κάποιους κοινούς στόχους για την κοινή πολιτική σε ό,τι αφορά τη διατήρηση του επίπεδου του γεωργικού εισοδήματο. Ποια είναι τα εισοδήματα των γεωργών, γνωρίζουμε πόσο πενιχρά είναι αυτά τα εισοδήματα. Τώρα, το Ταμείο Συνοχής. Η συνοχή και τα κονδύλια συνοχή. ε, πώς θα δρομολογηθούν προς την Ήπεθρο ή προς τα αστικά κέντρα γιατί θέλουμε να αξιοποιηθούν όσο γίνεται τα κονδύλια της συνοχής. Γι' αυτό και θα, θα θέλαμε να ετοιμάσετε κάποιες ε, συγκριτικές μελέτες για το πώς αξιοποιούν τα κονδύλια μας συνοχής οι πόλεις και πώς η ύπεθρος. Σε ό,τι αφορά τους μηχανισμούς παρέμβασης. Νομίζω ότι είναι απαραίτητοι μηχανισμοί παρέμβασης για τα διάφορα προϊόντα. Και αυτό που περιμένουμε είναι να μην ε, ε, δημιουργηθεί μια δυσμενής κατάσταση για τους εκτινοτρόφους. Επίσης, ε, η συγκυρία είναι αρνητική, αυξάνεται η φτώχεια, δημιουργείται μια γενική κρίση και θα πρέπει να υποστηρίξουμε και να χρηματοδοτήσουμε κονδύλια για την επιστημιστική ασφάλεια των, λιγότερο, των περισσότερων αδύναμων. Και η τελευταία ερώτηση. Δεν θα μπορούσαμε να έχουμε μια νομοθετική πρόταση που δεν θα μιλάει απλώς για γεωργική πολιτική. Αλλά ε, εδώ έχουμε μια πρόταση που μιλάει ουσιαστικά για μια γεωργοπεριβαλλοντική πολιτική. Δεν έχουμε μια γεωργική αμυγός πολιτική. Πολλά και διάφορα μπερδεύουμε εδώ. Επίσης ε, έχουμε το πρόβλημα του Μερκοσούρ. Προσπαθούμε να λύσουμε το πρόβλημα που έχουμε με τη Μερκοσούρ στο Παγκόσμιο Οργάνωση Γεωργίου ε, εις βάρος της γεωργίας. Στις πολιτικές ομάδες και στις εθνικές αντιπροσωπείες ε, συζητούμε όλα αυτά τα θέματα. Ε, και νομίζω ότι θα πρέπει να έχουμε πιο σοβαρή συζήτηση από ότι ε, σε ποιον θα δώσουμε και από ποιον θα αφαιρέσουμε για να δώσουμε σε άλλον. Δεν νομίζω ότι εκεί θα πρέπει να περιοριστεί η συζήτηση. Όστιγκερ. Ευχαριστώ κύριε Πρόεδρε, κύριε Επίτροπε. Νομίζω πως μπορούμε να πούμε πως παλέψατε πάρα πολύ καλά και επιτύχατε το καλύτερο δυνατό αποτέλεσμα αυτή την χρονική στιγμή. Και εμείς βεβαίως ε, δεν μπορέσαμε να περάσουμε όλα όσα θέλαμε στην έκθεση Σούρε και έπρεπε να αποδεχτούμε τις ε, πραγματικότητες και, τις, και την πλειοψηφία. Βεβαίω για μένα είναι σημαντικό αυτό το οποίο είπε ο πρόεδρος της Κομισιόν και ο κύριος Λεβαντόφσκι, ο αρμόδιος για τον προπολογισμό, μας έδωσε άλλα νούμερα από αυτά τα οποία ε, μας ε, δώσατε εμείς και νομίζω πως οι συζητήσεις οι οποίες εν μέρει έγιναν και μέσω των ε, ΜΜΕ έδειξαν πόσο δύσκολο είναι αυτό το θέμα. Παρ' όλα αυτά, εμείς εκπροσωπούμε την ε, γεωργία και τους αγρότες όπως ε, και εσείς. Γι' αυτό για εμάς είναι πάρα πολύ σημαντικό να έχουμε επαρκή προϋπολογισμό για το μέλλον. Προβληματικό θεωρώ το να καθορίσουμε αυτό το 30% του πρασινίσματος ε, σε αυτή την πρόταση ήδη, γιατί Ήδη αρκετά προγράμματα έχουν επενδύσει πάρα πολύ σε προγράμματα, αρκετά κρατημέλη έχουν επενδύσει πάρα πολύ σε προγράμματα του δεύτερου ε, πυλώνα και θα είναι προβληματικό αυτό για το μέλλον. Και αναφέρθηκε νομίζω ο κ. Χωσλίνγκ το πόσο σημαντικό είναι το πρασίνισμα στον πρώτο πυλώνα. Ας δούμε μόνο πόσο επιτυχή ήταν τα προγράμματα του δεύτερου πυλώνα τις προηγούμενες ε, δεκαετίες ε, στην εφαρμογή τους από τα κράτη-μέλη. Δεύτερη παρατήρηση αφορά τις μειονεκτικές περιοχές που δεν αναφέρθηκαν ρητός όπου πάντα ακούμε πως χρειάζεται να πάνε οι περιοχές αυτές στον πρώτο πυλώνα οι μειονεκτικές. Θα ήθελα κάποιο κάτι πιο συγκεκριμένο από εσάς ε, για αυτό το θέμα. Όπως σας είπα, σας ευχαριστώ για την ε, προσέγγισή σας. Όσον αφορά την ε, κριτική, δεν νομίζω πως θα πρέπει να απευθυνόμαστε σε εσά, μάλλον αυτά αφορούν τον Επίτροπο του Υπερπολογισμού. Σας ευχαριστώ, Γκαρσία Μπερέζ. Ευχαριστώ. Εγώ δεν θέλω να αμφισβητήσω εδώ τη φιλοδοξία και το έργο του κυρίου Επιτρόπου ε, όταν μας παρουσίασε την πρόταση αυτή και θα του συνιστούσα να μην ε, τις ε, παρεμβάσει των βουλευτών αυτής της Επιτροπής ως επίθεση αλλά ως επικοδομητική κριτική. Το αντικείμενο αυτής της κριτικής και των παρεμβάσεων ε, είναι να εγγυηθούμε το μέλλον της ΚΑΠ και όχι να επιτεθούμε στην ε, Κομισιόν. Έτσι λοιπόν πρέπει αυτές τις παρεμβάσει να τις δείτε με καλό μάτι και θέλω να αξιολογήσω αυτή την πρόταση με πρόταση με καλά αλλά και με μελανά σημεία γιατί γιατί σίγουρα περιλαμβάνονται νέα μέσα από εμεί από αυτό το κοινοβούλιο. Ε, τα είχαμε ζητήσει σε προηγούμενες συζητήσεις ε, και νομίζω ότι αυτό ανταποκρίνεται στην αμφιβολία που είχαμε και στην, ε, στο ότι αναρωτιόμαστε αν μπορούν αυτά τα μέσα να απαντήσουν στην κρίση ή στις συνέπειες της παγκοσμιοποίησης. Εσείς είπατε ότι θα υπάρξουν νομοθετήματα, θα αρμιστεί η νομική βάση. Εγώ έχω την αμφιβολία για το αν το Ταμείο Ταμείο για την Αντιμετώπιση των Κρίσεων ή την Αντιμετώπιση τη Παγκοσμιοποίηση θα ενεργοποιηθούν με μοφωνία από το Συμβούλιο, θα υπάρξουν ε, άλλα μέσα. Γιατί αυτό που επί τη αρχή μπορεί να είναι ένα καλό μέσο μπορεί να μετατραπεί ανάλογα με την ε, μετέπειτα νομοθετική δράση σε ένα μέσο που δεν ανταποκρίνεται στι προσδοκίε και στι αναγκαιότητε του τομέα. Και μπορώ να πω ότι, και λέω ότι έχει θετικά στοιχεία καθώ συμπεριλαμβάνονται θετικά ε, νέα μέσα, αλλά υπάρχει περικοπή στον πρώτο πυλώνα των άμεσων ενισχύσεων και εκεί θα έπρεπε να το ξαναδούμε το θέμα αυτό με ανησυχούν οι διαπραγματεύσει γιατί ξέρουμε όταν ε, ανοίγουν όλα τα χαρτιά θα πρέπει να προσπαθήσουμε να κερδίσουμε και αν στην πρόταση την αρχική της Κομισιόν υπάρχει ήδη περικοπή εγώ θέλω να επιμείνω στην μετέπειτα συζήτηση να μην υπάρχει μεγαλύτερη μείωση ε, σε σχέση με όσα έχει θέσει η Κομισιόν αυτή τη στιγμή και φυσικά αυτή τη θέση θα έχει αυτό το Κοινοβούλιο τοποθετήθηκε και η Επιτροπή Γεωργίας όπως και η του Κοινοβουλίου στις εκθέσεις ε, και, και για τις δημοσιονομικές προοπτικές και νομίζω ότι θα συνεχίσουμε να διεκδικούμε αυτή τη θέση για να εγγυηθούμε βιώσιμο μέλλον για την ΚΑΠ που να μπορεί να απαντά στις υφιστάμενες προκλήσεις. Μαρία και κατόπιν ε, Χέρας Γκαρσία. Ευχαριστώ. Κύριε Επίτροπε, θα ήθελα να σας ευχαριστήσω και εγώ, όπως ε, έκαναν και άλλοι, και για την παρουσίασή σας και για τις ε, προσπάθειές σας για να διατηρηθεί ε, στο τωρινό του ύψος ο προπολογισμός γεωργίας. Έχω τέσσερις ερωτήσεις. Σχετίζεται με την νέα κοινή γεωργική πολιτική, η οποία θα είναι πιο δική. Θα είμαστε σε θέση να μειώσουμε την ε, διαφορά στις άμεσες πληρωμές ε, μεταξύ των κρατών μελών, ειδικά όσον αφορά τα νέα κράτη-μέλη και αυτό θα συμβεί ήδη το 2014 αντί για το 2016 όπως θέλουν κάποιοι δεύτερον. Ε, θα ήθελα να σας ρωτήσω εάν ο προπολογισμός κοινής γεωργικής πολιτικής ευθυγραμμίζεται με ε, Προπολογισμού όπως αυτός για την περιφερειακή πολιτική και την ε, στρατηγική του Δούναβη που αφορά κυρίως ε, την ανάπτυξη πέθρου και τη βιοποικιλότητα κατόπιν. Όσον αφορά τον τομέα της μελισσοκομείας σκοπεύετε να την στηρίξετε και τι σκοπεύετε να κάνετε για πληρωμές ανά κυψέλη μετά το 2014. Ξέρουμε πως δεν είναι δυνατόν αυτή τη στιγμή, αλλά η μελισσοκόμη είναι πραγματικά σε απολυπιστική κατάσταση. Και τέταρτον, το Ταμείο Παγκοσμιοποίησης υπάρχει, αλλά ξέρουμε πως σε κάποια κράτη-μέλη, δεδομένων των διοικητικών διαδικασιών, είναι πρακτικά δυνατόν να ε, ενταχθεί κανείς σε αυτό το ταμείο, το οποίο ακούγεται θα, θαυμάσιο, αλλά θα πρέπει να έχει και νόημα για όλα τα κράτη-μέλη. Ευχαριστώ. Κύριε Πίτροπε εσείς γνωρίζετε πολύ καλά την κοινοτική γεωργία και στα παλιά και στα νέα κράτη-μέλη. Ε, γι' αυτό ξέρω ότι δεν είναι αυτός ο προϋπολογισμός που εσείς θα θέλετε να μας ανακοινώσετε σήμερα, αλλά επί αυτού πρέπει να εργαστούμε και εγώ θα έλεγα ότι όλο αυτό μου φαίνεται ανησυχητικά γιατί αυτό που εξευγενισμένα αποκαλεί η Κομισιόν ε, πάγωμα έχουμε μείον 11% ε, στον ε, πρώτο πυλώνα και μείον 5% στο δεύτερο πυλώνα της ανάπτυξης της υπέτρου. Έτσι λοιπόν για αυτή την ανησυχία εγώ σας προτείνω και στην πρότασή σας που θέλουμε να μας πείτε ποια θα είναι, ποιο θα είναι το ποσό τον Οκτώβριο και επίσης ε, για αυτό το πρασίνισμα 30%. Αυτό το 30% δεν συνάδει με το πέσμα που μας παρουσιάζει η Επιτροπή και σας ε, είπα ότι εδώ κρούω και τον κοδόνα του κινδύνου γιατί όταν ε, μιλάμε για μεταφορές μεταξύ πρώτου και δεύτερου πυλώνα εγώ εδώ θεωρώ ότι μπορεί να ανοίξουμε την πόρτα για την επαναθηνικοποίηση της ΚΑΠ. Μου φαίνεται ε, ότι αυτό είναι ένα πολύ επικίνδυνο προηγούμενο και ξέρουμε ποια μπορεί να είναι η κατάληξη. Και όταν ε, μιλάτε για το Ταμείο Προσαρμογή στην Πικοσμιοποίηση, εγώ αυτό που βλέπω είναι ένα κίνδυνο γιατί εδώ προτρέχουν και, και μάλλον έχουμε μία πληγή και βάζουμε έναν επίδεσμο απλά. Και σας ε, αναφερθήκατε σε αυτά τα 2,5 δισεκατομμύρια για τις, ε, ε, στις, στα πλαίσια των διεθνών συμφωνίων, όμως ξέρετε πότε θα μπορέσουν να ενεργοποιηθούν αυτά τα κονδύλια. Μισελ Νταντέν και κατόπιν Καλινόσκι. Ευχαριστώ. Θέλω και εγώ να ευχαριστήσω τον Πρόεδρο για το έργο του. Ευχαριστώ λοιπόν τον Επίτροπο για τη δουλειά που έκανε. Όλοι γνωρίζουμε ότι έχουμε διανύσει πολύ μεγάλο δρόμο και ακόμη και αν δεν είμαστε απόλυτα ικανοποιημένοι είμαστε κοντά τώρα. Θέλω να αναφερθώ στη διάρθρωση με το Ταμείο Συνοχής με άλλους επιτρόπους, ε, όπως και με τον Πρόεδρο της Κομισιόν, να λάβατε την πρωτοβουλία ε, για το ε, πώς θα γίνει η προετοιμασία και του προϋπολογισμού σε σχέση και με το Ταμείο Συνοχής και στους ίδιους πόρους. Υπήρχαν κάποιοι πόροι για την καλλιέργεια ζαχαρότευθλου ε, και έτσι λοιπόν θα ήθελα να ρωτήσω αν θα συνεχίσει να υπάρχει αυτή η συνεισφορά για τη συγκεκριμένη καλλιέργεια. Ευχαριστώ. Κύριος Καλινόφσκι και μετά ο κύριος Γιάρ. Ευχαριστώ κύριε Πρόεδρε. Κύριε Επίτροπε, το ύψος ε, των κονδυλίων προβλέπονται για την κοινή γεωρική πολιτική. Αυτό είναι ένα πράγμα και ο τρόπος ταξινόμηση κατανομή των κονδυλίων αυτών στα διάφορα επιμέρου κεφάλαια τη γεωργική πολιτική, αλλά και η κατανομή μεταξύ των κρατών είναι κάτι διαφορετικό. Άλλο το ένα, άλλο το άλλο και νομίζω ότι περισσότερο μας ενδιαφέρει το δεύτερο θέμα της κατανομής, δηλαδή παρά το συνολικό ύψος των κονδυλίων της α, γεωργικής πολιτικής. Και επανέρχομαι εδώ στην ανακοίνωση της Ευρωπαϊκής Επιτροπής του περασμένου Νοεμβρίου. Εκεί αναφερόταν μια πολύ σημαντική δήλωση σε ό,τι αφορά την, ε, ε, τις ιστορικές, ε, τα ιστορικά επίπεδα αναφοράς και η αντικατάσταση αυτών των ιστορικών επίπεδων αναφοράς από αντικειμενικά κριτήρια. Πού είναι λοιπόν αυτά τα αντικειμενικά κριτήρια, αγαπητέ κύριε Επίτροπε. Δεν μπορούμε τους μηχανισμούς το 33 προς 90% του μέσου όρου να τα θεωρούμε ως αντικειμενικά κριτήρια. Πού είναι τα αντικειμενικά κριτήρια που υποσχεθήκατε, που όντως θα πρέπει να καθορίζουν το ύψος ε, της ε, ενίσχυσης για τους μεμονωμένους γεωργούς, παρόλο που έχουν την ίδια γεωργική δραστηριότητα. Επίσης, η διαφορά μεταξύ του σχεδίου της Ευρωπαϊκής Επιτροπής ε, είναι από 140 από 440 σε 450 δεν έχει και μεγάλη, σε 500 δεν έχει και μεγάλη διαφορά. Τι γίνεται όμως με τους γεωργούς στην Πολωνία, στην Πορτογαλία, στην Αυστρία, στην, στην, στην Σουηδία, στην ε, Μεγάλη Βρετανία που θα λάβουν 200-250 εκτάρια. Το εκτάριο θα, έχουν την, θα πρέπει να έχουν ανταγωνισμό με άλλους γεωργούς που θα λαμβάνουν 400-450 ευρώ ανά Η ενιαία αγορά έχει νόημα και η εσωτερική αγορά έχει νόημα όταν πραγματικά εξασφαλίζουμε συνθήκε ισότιμου ανταγωνισμού. Αλλά δυστυχώς δεν φαίνεται να έχουμε ισότητα στην Ευρωπαϊκή Ένωση γιατί η μερική είναι ισότερη από του υπόλοιπου. Ευχαριστώ κύριε Καλινόφης και κύριο Γιάρ και μετά όσο Ζεμποβέ. Κύριε Σιγιάρα, ευχαριστώ κύριε Πρόεδρε, ευχαριστώ κύριε Επίτροπε για την παρουσία σα. και θα ήθελα να σας ευχαριστήσω για τον αγώνα που δώσατε για τον προϋπολογισμό της Γεωργίας. Έχω τέσσερα σύντομα ερωτήματα. Το πρώτο ε, σχετίζεται με τα πολιτικά επιχειρήματα και την πραγματικότητα επιτόπου. Γιατί είπατε πώς καταφέρατε να ενισχύσετε τον προϋπολογισμό της Γεωργίας. Βεβαίως οι Γεωργοί μας θα το δουν αλλιώς και θα δουν τι θα λάβουν το 2013 και το 2014 και το 2013 στον πρώτο πυλώνα έχουμε 46,6 δις και 2014 μιλάμε για 40,3 οπότε μιλάμε για μείωση 40 ευρώ ανά εκτάριο οπότε θα δουν τι θα λάβουν οι γεωργοί οπότε πρέπει να τα πούμε ανοιχτά τα πράγματα. Έχω κάνει εγώ λάθος υπολογισμούς ή ε, υπάρχει διαφορά μεταξύ ε, πραγματικής, ε, μεταξύ πραγματικότητας και πολιτικών επιχειρημάτων. Δεύτερον, έχουμε ένα ε, πρόβλημα. Τα κράτη-μέλη δεν αποδέχονται ακόμα τον ευρωπαϊκό προπολογισμό. Θέλουν να μας δώσουν λιγότερα από όσα χρειαζόμαστε. Πώς εκτιμάτε την ε, κατάσταση. Θα υποχωρήσουν τα κράτη-μέλη, θα υπάρχουν περικοπές. Εάν υπάρξουν περικοπές, πού θα γίνουν κατά την άποψή σας. Τρίτον, η ένταξη νέων κρατών μελών. Θα έχουμε περισσότερα λεφτά ή θα πρέπει να τα βρούμε από τον υπάρχοντα προπολογισμό. Και τέταρτο και τελευταίο πότε θα καταθέσετε συγκεκριμένες ε, προτάσεις ε, για την σταδιακή μείωση των ε, άμεσων πληρωμών, της αποσύνδεσης δηλαδή. Ζωζέ Θα προσπαθήσω να είμαι σύντομος γιατί περνάει και η ώρα. Ένα σχόλιο Καταρχήν, νομίζω ότι έδωσε μάχη ο Επίτροπος ε, για τον προπολογισμό και έκανε περισσότερο από ό,τι μπορούσε στο πλαίσιο που γνωρίζουμε. Το θέμα είναι ότι έχουμε ενώπιον μας και το Συμβούλιο και το Συμβούλιο δεν είναι ε, απαραίτητο ο καλύτερος σύμμαχος του ΣΠΑΚ γιατί έχουμε διάφορες αποκλήσεις και εγωσμούς από τα κράτη. Το δεύτερο πρόβλημα που έχουμε είναι ότι ζητάμε σήμερα να έχουμε ένα προπολογισμό σε ένα περιορισμένο πλαίσιο του 1% του ΕΕΠ των κρατών ε, και σήμερα θέλουμε και περισσότερες πολιτικές. Εγώ πιστεύω ότι θα πρέπει να σκεφτούμε προοδευτικά τους ίδιους πόρους. Πώς μπορούμε λοιπόν να επανατροφοδοτήσουμε ε, μέσω των ίδιων πόρων την ΚΑΠ όπω στο παρελθόν ε, πριν ε, από το 1991 φτάναμε μέχρι το 60% του προπολογισμού της ΚΑΠ που χρηματοδοτούνταν από τους ίδιους πόρους και μάλιστα από τους φόρους στα σύνορα. Ε, έτσι λοιπόν νομίζω ότι πρέπει να το σκεφτούμε αυτό γιατί θα βλέπουμε όλο και περισσότερο να περιορίζεται ο προπολογισμό μας αν δεν έχουμε χρηματοδότηση και από ίδιου φόρους. Ε, τώρα η πολιτική για την έρευνα, ναι νομίζω είναι ενδιαφέρον, αγροτική έρευνα είναι πρώτη φορά που θα το έχουμε αυτό αλλά νομίζω ότι πρέπει να σχετίζεται με τις προτεραιότητες της ΚΑ δηλαδή να μπορούμε να έχουμε μία συνέπεια, μία συνάφεια έτσι ώστε αυτός ο προπολογισμό να μπορέσει να ενισχύσει, ε, παραδείγματο χάρη, την καταπολέμηση τη κλιματική αλλαγή, να υπάρχει παρασύνισμα. Ενίσχυση λοιπόν σε αυτό. Και δεύτερο στοιχείο, δεν θέλω να επαναλαβώ σε είπαν για το Ταμείο για την Παγκοσμιοποίηση, αλλά αν προσθέσουμε το Ταμείο τη Παγκοσμιοποίηση και τα έκτακτα μέτρα, έχουμε 6 δι, 6,3 δι που σχετίζονται με τι οικονομικέ κρίσει, με τα οικονομικά προβλήματα σχετικά με την ΚΑΠ. Εγώ νομίζω ότι κάτι που πρέπει να είναι στο επίκεντρο αυτών των αριθμών είναι το θέμα του κόστους ε, της παραγωγής. Ψηφίσαμε την έκθεση που παρουσίασα ε, και είπαμε ότι δεν πρέπει να πληρώνω τη γεωργία κάτω από το κόστος παραγωγής τους, αλλά νομίζω ότι εδώ έχουμε ένα πολύ σαφές σημείο, δηλαδή για να βρούμε τους τρόπους υποστήριξης, ενίσχυσης και αύριο θα χρειαζόμαστε λιγότερο τις άμεσες ενισχύσεις, αν μπορούν οι γεωργοί να ζουν πολλούντας, τη δική τους παραγωγή για, ε, με έναν τρόπο ώστε να καλύπτουν το κόστος παραγωγής. Μάτο και κατόπιν Ευχαριστώ. Συμφωνούμε όλοι ότι ο Επίτροπος ε, έκανε τεράστιες προσπάθειες υπέρ ενός αξιοπρεπούς προϋπολογισμού της γεωργικής πολιτικής. Αλλά δεν θα πρέπει μετά την ε, προσπάθεια αυτή να παρετηθείτε. γιατί σήμερα σας είδα όχι μόνο παρετημένο, αλλά να σκέφτεστε για παρηγοριά ότι θα μπορούσαν να είναι και χειρότερα τα πράγματα. Θα σας θέλω παρακαλούσα να μην σταυρώσετε τα χέρια, να μην παρετηθείτε και θα έχετε όλοι μας την υποστήριξη για να συνεχίσετε την προσπάθεια. Και παρά την δύσκολη κατάσταση που αντιμετωπίζουν οι γεωργοί, με όλο και πιο αυστηρέ απαιτήσει και για περιβαλλοντικές προδιαγραφές και για την, για την ποιότητα της διατροφής, προτείνεται παρόλα αυτά σημαντική συρρήκνωση των κονδυλίων της ΚΑΠ. Και αυτό είναι απαράδεκτο. Δεν μπορούμε να ζητούμε από τους γεωργούς να αναλαμβάνουν νέες υποχρεώσεις και ταυτόχρονα να τους κόβουμε τα κονδύλια. Επίσης έχουμε απευδίσει να πληρώνει όλα τα σπασμένα ο Γεωργός και την κρίση και τις εμπορικές συμφωνίες και τα σπασμένα των δημοσιονομικών περικοπών φτάνει πια. Και αναφερθήκατε και στις εμπορικές συμφωνίες. Είπατε ότι το Ταμείο Παγκοσμιοποίησης θα περιορίζεται στις συνέπειες των εμπορικών συμφωνιών. Ε, θα καλύψει δηλαδή όλες τις εμπορικές συμφωνίες. Για παράδειγμα με την Κολομβία, τη συμφωνία με το Περού, γιατί και αυτές οι συμφωνίες ε, αποβαίνουν εις βάρος σημαντικών καλλιεργιών, όπως ε, τις καλλιέργειες μπανάνας. Ποια θα είναι, ποιο θα είναι το πεδίο εφαρμογής του Ταμείου Παγκοσμιοποίησης και για τις εξόχως απόκειτες περιοχές. Αν η οι μειώσει αυτέ πλήξουν ε, τον απλό γεωργό, φανταστείτε τι θα γίνει με του γεωργού των απόμακρων περιοχών. Δεν θα πρέπει να του δώσουμε μία ακόμη λυπητερή να πληρώσουν, γιατί έχουν, έχουν πληρώσει διπολά. Θέλουμε την επαρκή χρηματοδότηση του ΠΟΣΕΙ. Δεν θα πρέπει να το μειώσουμε, αντίθετα να το αυξήσουμε. Και παρακαλώ να μην μα απογοητεύσετε και να μην διαψεύσετε τι προσδοκίε μα, κύριε Επίτροπε. Σα ευχαριστούμε, κύριε Μάτο, ο κύριο Άλντε και τελευταίο ο κύριο Ρέμερ. Ευχαριστώ, κύριε Πρόεδρε. Κύριε Επίτροπε, για να χρησιμοποιήσω τη δική σας εικόνα των καυσίμων και του κινητήρα, θα ήθελα να πω ότι σε πολλούς τομείς χρειαζόμαστε βενζίνη και καύσιμα στην Ευρώπη. Και κάνατε ό,τι μπορούσατε φυσικά για να μην μειώσετε περαιτέρω τα ποσά. Αλλά εμείς στο Ευρωπαϊκό Κοινοβούλιο θέλουμε να έχουμε έναν ισχυρό κινητήρα που θα καταφέρει να ανταποκριθεί στις προκλήσεις και να καλύψει και την απόσταση που έχει για να υλοποιήσει τους στόχους που έχει θέσει. Και ελπίζω να μείνει στο δρόμο το μηχάνημα λόγω έλλειψης καυσίμων. Χρειαζόμαστε περισσότερα καύσιμα για τον κινητήρα, τον ισχυρό κινητήρα που κατασκευάζουμε. Γιατί έχουμε και μεγάλες αποστάσεις να διανύσουμε. Έχουμε τις προκλήσεις που ήδη αναφέραμε και που ήδη έχουμε συμφωνήσει. Θέλουμε να βελτιώσουμε την ε, ισότητα κατανομής ε, των κονδυλίων μεταξύ των γεωργών. Και αυτή είναι η σημαντική πρόκληση, να αποκαταστήσουμε μια ισορροπία. Και επίση έχουμε και την πρόκληση των ε, λιγότερων ανεπτυγμένων περιοχών, ώστε να διασφαλίσουμε τη γεωργία σε ολόκληρη την Ευρωπαϊκή Ένωση. Γιατί έχουμε τι εξόχω απόκεντρε περιοχέ που υφίστανται πολύ ε, μεγαλύτερες ε, συνέπειες από τις συμφωνίες ε, του Μερκοσούρ για παράδειγμα και από τις ποσοστώσεις χρειαζόμαστε και οι περιφέρειες χρειάζονται μια φιλόδοξη γεωρική πολιτική για να αντιμετωπίσουν τις πιο δύσκολες προκλήσεις που έχουν. Ευχαριστώ. Ναι, θα ήθελα πρώτα απ' όλα να σας ευχαριστήσω για τη μεγάλη σας υπομονή που μας ακούτε τόση ώρα και σύντομα να αναφερθώ στο ότι αυτό το οποίο συζητάμε είναι ακόμα σχέδιο, μια πρώτη τοποθέτηση της Κομισιόν. Και θα έχουμε ακόμα πολύ έντονες συζητήσεις στο προσεχές μέλλον, ειδικά αν σκεφτούμε το ότι δεν έχουμε ξεπεράσει ακόμα την οικονομική κρίση. Δεν υπάρχει μόνο η γεωργία στον ευρωπαϊκό προϋπολογισμό. Νομίζω λοιπόν πως η Κομισιόν θα πρέπει και θα γίνουν οπωσδήποτε έντονες συζητήσεις μεταξύ Συμβουλίου, Κοινοβουλίου και Κομισιόν και βεβαίως είναι πιθανόν να αυξηθούν ή και να μειωθούν τα κονδύλια. Και αν μειωθούν, πρέπει να σας ρωτήσω ξεκάθαρα πόσο χαμηλά μπορούμε να πάμε και αν είναι δυνατόν να εφαρμοστεί μετά ένα πρασίνισμα. Πόσο χαμηλά μπορούμε να πάμε και πρέπει να μετά αναλυφθεί μια απόφαση προστασία του περιβάλλοντος ή ασφάλεια των τροφίμων. Πότε φτάνουμε στο όριο του πόνου των ε, περικοπών για να εργαστούμε επιλεκτικά και να πούμε πρέπει να αποφασίσουμε πού θα κόψουμε, γιατί αν κόψουμε γενικώ δεν θα έχουμε πλέον ε, ευρωπαϊκή γεωργική πολιτική. Molto bene, abbiamo finito questo lungo. Πολύ ωραία, ολοκληρώσαμε λοιπόν και αυτό το μακρύ κατάλογο των ομιλητών. Ευχαριστώ τον Επίτροπο που όχι μόνο άκουσε τα πάντα, αλλά σημείωσε και με πολύ μεγάλη ακρίβεια όλες τις παρεμβάσεις όλων των βουλευτών. Λοιπόν, αγαπητέ Επίτροπε, όπως ε, είπε ο κύριος ε, Λεφόλ, είμαστε στην αρχή αυτού του αγώνα και εμείς η Επιτροπή Γεωργίας και το Ευρωπαϊκό Κοινοβούλιο ε, ξέρουμε ε, ότι μας περιμένει και το Συμβούλιο και ότι δεν θα θέλει να δώσει πολλά στη Γεωργία, γι' αυτό δεν είμαστε και ιδιαίτερα ικανοποιημένοι. Έτσι λοιπόν, εμείς είμαστε συμμαχοί σας για να συνεχίσετε αυτόν τον αγώνα και να ε, κατορθώσουμε να δώσουμε περισσότερο περισσότερα και να έχουμε την κοινή αγροτική πολιτική που όλοι επιθυμούμε για τη Γεωργία. Έχετε το λόγο. Ευχαριστώ, Πρόεδρε. Είπε κάποιος εδώ, ο κύριος Μάτο, νομίζω ότι δεν θα πρέπει να τα παρατήσει ο Επίτροπος. Εγώ καθόλου παρατημένος δεν είμαι. Σας είπα απλώς ε, ότι από την αρχή της αιτίας μου μέχρι τώρα σας ε, έλεγα πάντοτε ότι ο στόχος μου είναι να προσπαθήσω να διατηρήσω τον προπολογισμό της ΚΑΠ. Τώρα μπορώ να έρθω και να σας πω εδώ ότι αυτή είναι η πρόταση της Κομισιόν. Λέω λοιπόν απλώ ότι αυτό είναι ένα στάδιο, ένα βήμα το οποίο κάναμε. Ξέρω ότι δεν έχει ολοκληρωθεί η διαδικασία και εσείς το γνωρίζετε, αλλά λέω επίσης ότι τώρα βάσει των προτάσεων της Κομισιόν, που είναι μια επίσημη πρόταση, ε, η οποία μας δείχνει και το επαναλαμβάνω ότι η Κομισιόν διατηρεί την ΚΑΠ, την Κοινή Αγροτική Πολιτική, ως ε, την κύρια δημοσιονομική δαπάνη στην πρότασή της. Έτσι λοιπόν αναγνωρίζεται τώρα η ΚΑΠ από το σύνολο των επιτρόπων ως ένας ε, πρωταρχικός στόχος ε, του κοινωτικού προπολογισμού. Αλλά αυτή είναι μια πρόταση που υποβάλλει η Κομισιόν. Ένας ε, προϋπολογισμός ο οποίο είναι φιλόδοξο αλλά και ρεαλιστικό όπω είπε και ο πρόεδρο τη Κομισιόν. Γιατί υποβάλαμε αυτέ τι προτάσει, τώρα τι καταθέσαμε ενώπιον Συμβουλίου και Κοινοβουλίου σε δύσκολους δημοσιονομικούς ε, καιρούς για την Ευρωπαϊκή Ένωση, αλλά και σε μια κατάσταση όπου τα κράτη-μέλη ζητούν από την Κομισιόν να είναι πιο φιλόδοξη, όχι μόνο να διατηρήσει δηλαδή τις παραδοσιαστές της πολιτικές, αλλά να κάνει και πολλά περισσότερα και σε άλλους τομείς. Νομίζω ότι μπορείτε να συμφωνήσετε με το ότι δεν είναι εύκολη η επιλογή και δεν ήταν ε, εύκολη συζήτηση που είχαμε στο Σώμα των Επιτρόπων ε, για να βρούμε μια ισορροπία αφενός να διατηρήσουμε ισχυρές πολιτικές όπως ε, η ΚΑΠ αλλά και από την άλλη να έρθουμε και να καταθέσουμε σε εσά και στο Συμβούλιο προτάσει με φιλόδοξους στόχους που δεν είχαμε στο παρελθόν. Έτσι λοιπόν, σε αυτή το δύσκολο πλαίσιο, στη δύσκολη συγκυρία, το μόνο που λέω εγώ είναι ότι εγώ, ως Επίτροπος ε, Γεωργίας, μπορώ να μιλήσω εξ ε, του Σώματος των Επιτρόπων και να σα πω, ορίστε ένας φιλόδοξος προπολογισμό για την ΚΑΠ σε αυτή τη δύσκολη συγκυρία. Δεν πρόκειται λοιπόν καθόλου για παρέτηση. Επίση, συμφωνώ μαζί σας και γι' αυτό τώρα θα μπω σε λεπτομέρειες, ορισμένε ερωτήσει, πώ θα κάνουμε το τάδε ή το δίνα θα ξεκινήσουμε από τον Οκτώβριο να συζητούμε λεπτομερώς πώς θα τα χρησιμοποιήσουμε όλα αυτά. Νομίζω ότι κατανοείτε ότι δεν μπορώ να έρθω τώρα και να σας δώσω περισσότερες λεπτομέρειες. Ορισμένοι εξημών είπατε ότι μπαίναμε σε υπερβολικές λεπτομέρειες για τις δημοσιονομικές προοπτικές για τις ΚΑΠ, ενώ άλλοι ε, είπατε ότι θέλετε περισσότερες λεπτομέρειες. Αλλά όλα αυτά θα τα βρείτε στην νομοθετική πρόταση. Και ξέρω ότι οι δυσκολίες μόλις ξεκινούν στη δουλειά που έχουμε μπροστά μας. Γιατί με όσα έχουμε ως καύσιμο θα πρέπει να δούμε πώς θα το χρησιμοποιήσουμε, πώς θα το μοιραστούμε για να μπορέσουμε να πετύχουμε καλύτερα τους στόχους μας. Λοιπόν, κύριε Γιαγγέλ, για το πρώτο δεύτερο πυλώνα, το πρασίνισμα και τα αγιοπεριβαλλοντικά μέτρα. Θα σας ασφαλίσω για το εξής επειδή βάζουμε το πρασίνισμα στον πρώτο πυλώνα, δεν σημαίνει αυτό ότι θα αποδυναμώσουμε τον ένα πυλώνα για να τα μεταφέρουμε στον άλλο. Αυτό το είπα και στην Ολομέλεια, όταν συζητήσαμε την έκθεση Και το είδατε κι εσείς. Προσπαθήσαμε να το καθορίσουμε στις δημοσιονομικές προοπτικές. Δεν θα χρεώσουμε το πρασίνισμα του πρώτου πυλώνα στο δεύτερο πυλώνα. Στο δεύτερο πυλώνα μένουμε με υγειοπεριβαλλοντικά μέτρα που θα δώσουν δυνατότητα στα κράτη-μέλη και στις περιφέρειες να συνεχίσουν να χρηματοδοτούν ε, τα μέτρα αυτά συν τα μέτρα περί πρασινίσματος. Δεν θα θυσιάσουμε τον υπέρ του άλλου. Για τις εμπορικές συμφωνίες. Λέτε ότι είναι φόβος για το Κοινοβούλιο και για την Επιτροπή Γεωργίας. Ε, πρέπει να δούμε τι σκεφτό και τα κράτη. είπα και επαναλαμβάνω, δεν σημαίνει ότι επειδή βάλαμε αυτή τη ε, δημοσιονομική γραμμή για το Ταμείο Παγκοσμιοποίηση, αυτό σημαίνει ότι τώρα πιο εύκολα θα συναπτούμε εμπορικέ συμφωνίε. Πρέπει να είμαστε εξίσου προσεκτικοί και πάντοτε θα πρέπει να αξιολογούμε τον αντίκτυπο. Γιατί μπορεί να υπάρχει κάποιο σοβαρό αντίκτυπο ε, από ορισμένες ε, εμπορικέ συμφωνίε που δεν έχουμε διαπραγματευτεί σωστά, που δεν μπορούμε να αντισταθμίσουμε με αυτά τα 2,8 δισεκατομμύρια. Δεν τα βάλαμε λοιπόν γι' αυτό, αλλά όταν υπάρχει ένα συγκεκριμένο αντίκτυπο, θα πρέπει να έχουμε και τα μέσα για να μπορούμε να κάνουμε αυτή την αντιστάθμιση και να μην χρησιμοποιήσουμε τι άμεσε πληρωμέ ε, ή το δεύτερο για αυτές τις συγκεκριμένε αποζημιώσεις. Και αυτό το Ταμείο Παγκοσμιοποίησης εγώ το βλέπω ευρύτερα, πέρα από τις εμπορικές συμφωνίες. Αλλά και πάλι με ρωτάτε επί περισσότερων λεπτομεριών. Θα πρέπει να παρουσιάσουμε περισσότερε λεπτομέρειε, θα πρέπει να παρουσιάσουμε νομική βάση. Τώρα δεν μπορώ να σα δώσω περισσότερα στοιχεία, γιατί ε, επί πολλών στοιχείων ζήτησα από τι υπηρεσίε μου ήδη να προβούν σε μια νομική ανάλυση για το πώ θα χρησιμοποιήσουμε όλα αυτά τα μέσα. Μόλις ολοκληρώσαμε τη διαδικασία διαπραγματεύσεων για τα αριθμητικά στοιχεία τώρα, τους επόμενου μήνες, θα έχουμε την ευκαιρία να σκεφτούμε επί των νομοθετικών προτάσεων. Κύριε Λεφόλ, είπε ο κύριο Λεφόλ ότι δεν έχει ολοκληρωθεί η δημοσιονομική μάχη, το είπε και στην αρχή, συνειδητοποιώ ότι για πρώτη φορά εδώ και πολύ καιρό συζητούμε τη μεταρρυθμίση της ΚΑΠ και τον προπολογισμό. Υπάρχουν κάποιοι σύνδεσμοι που πρέπει να γίνουν και προσαρμογές και υπάρχει και ένα σύνδεσμο μεταξύ της πολιτικής συνοχής, δηλαδή τον προπολογισμό για την πολιτική συνοχή και τον προπολογισμό για την ΚΑΠ, για να μπορέσουμε να διατηρήσουμε μια ισορροπία στη δημοσιονομική κατανομή μεταξύ των διαφόρων κρατών μελών. Υπάρχουν ορισμένα όρια που πρέπει να βάλουμε και από τη μία και από την άλλη πλευρά σε ό,τι αφορά την κατανομή των κονδυλίων μεταξύ των κρατών μελών. Έτσι λοιπόν είναι σαφέ ότι ανάλογα με το πώ θα εξελιχθούν οι διαπραγματεύσει μεταξύ Συμβουλίου και Κοινοβουλίου βάσει των προτάσεων τη Κομισιόν για τον προπολογισμό, ίσως ε, θα έχουμε και κάποιες οριακές επιπτώσεις ό,τι αφορά την κατανομή των κονδυλίων μεταξύ των κρατών μελών στα πλαίσια της ΚΑΠ. Γι' αυτό πολλοί από τους ομιλητές ε, αναφέρθηκαν σε αυτό το όριο επανεξισορρόπησης με το 1 τρίτο. Θα είμαι σαφής, σαφής, με συγχωρείτε. Δεν είναι το 1 τρίτο του μέσου όρου. Αυτό που λέει η πρόταση Βάσει αιτήματο ε, του Αρμόδιου Επιτρόπου για τον Προπολογισμό και μπορώ να σα πω ότι όλο το Σώμα των Επιτρόπων, όλοι οι Επίτροποι συμφωνούσαν με αυτή την πρόταση. Όλοι συμφώνησαν να αυξηθεί ακόμη κατά ένα τρίτο το σημερινό επίπεδο για να φτάσουμε στο, στο επίπεδο το 90% με την ε, επανισορρόπηση που θα κάνουμε το περιορίσαμε αυτό σε μία αύξηση ενός τρίτου και όχι παραπάνω. Για την συνολική κατανομή του δημοσιονομικού φακέλου μεταξύ των κρατών μελών, έτσι ώστε να μην δημιουργηθεί ανισορροπία σε σχέση με το τι μπορεί να λάβουν κρατημέλη με αυτή την αύξηση για την ΚΑΠ και σε σχέση με το τι μπορεί να λάβουν βάση πολιτική συνοχή ή άλλων πολιτικών, αλλά κυρίω για την πολιτική συνοχή. Από εκεί προέρχεται ο περιορισμό. Πρόκειται για μια πρόταση που έγινε από τον αρμόδιο Επίτροπο για τον Προπολογισμό. Είδε αυτό το θέμα τη ισορροπία και αυτή η πρόταση έγινε αποδεκτή από όλου του επιτρόπους. Υπάρχει λοιπόν συνδυσμός μεταξύ των διαπραγματεύσεων του συνολικού πακέτου και του τρόπου της κατανομής ε, των κονδυλίων μεταξύ των κρατών μελών. Τώρα για τους ε, απόρους. Επαναλαμβάνω το ότι μεταφέραμε αυτό το δημοσιονομικό άκθο στο κοινωνικό ταμείο δεν σημαίνει ότι το πρόγραμμα για τους απόρους αποσυνδέεται από την κοινή αγροτική πολιτική. Το πρόγραμμα για τους απόρους ξεκολουθεί να παραμένει συνδεδεμένο με την ΚΑΠ, γιατί τώρα διασφαλίζεται αυτός ο φάκελος ε, αυτός. Ε, έχουμε 0,8 δισεκατομμύρια για αυτό το τομέα. Τώρα δεν έχει σημασία αν θα υπάρχει ε, αποδηματικό παρέμβασης καθώς ε, η μόνη πηγή χρηματοδότησης ήταν και είναι πολιτική νομικά, συνόμασταν με την ε, τιμή ε, του αποθέματος τη παρέμβασης. Τώρα δεν μπορούμε να χρηματοδοτήσουμε περισσότερο σε σχέση με το απόθεμα που έχουμε στη διάθεσή μας τώρα με αυτό το ποσό 2,8, με συγχωρείτε, δισεκατομμύρια, έχουμε διασφαλίσει για το πρόγραμμα των απόλων 400 εκατομμύρια ευρώ ετησίων. Αν υπάρχουν αποθέματα παρέμβασης, αυτό το επίπεδο της κατανομής θα μπορούσε να ανέβει. Γιατί μπορούμε να το συμπληρώσουμε με το απόθεμα παρέμβαση, αλλά τουλάχιστον αυτό το διασφαλίσαμε. Αλλά η νομική βάση παραμένει αυτή που είχαμε προτείνει. Θα την προσαρμόσουμε τώρα μετά το 2013, αλλά και πάλι ευχαριστώ την προσοχή σας στο ότι αν δεν καταλήξουμε σε συμφωνία στο ιστορικό του Συμβουλίου με τα κράτη-μέλη, με την πλειοψηφία των κρατών μελών για την νομική βάση και η Κομισιόν ήδη πρότεινε το 2008 επαναπροσαρμογή, το 2010 δεν κινδυνεύουμε το 2012 και ξέρετε ότι έχουμε πολύ μειωμένη κατανομή το 2013 και κινδυνεύουν να έχουμε 0 ευρώ για το πρόγραμμα για του οπόρου. Έτσι λοιπόν, η νομική βάση που προτείνει η Κομισιόν εξακολουθεί να ισχύει και θα πρέπει να βρούμε τη λύση για να μπορέσουμε να την αφήσουμε και να μπορέσουμε να συνεχίσουμε το πρόγραμμα αυτό και το 2013. Σε ό,τι αφορά τώρα το νότατο όριο και τη σταδιακή μείωση, περισσότερε λεπτομέρειε με την ε, νομοθετική πρόταση τον Οκτώβριο. Αυτό που κάναμε στις δημοσιονομικέ προοπτικέ ήταν να υπογραμμίσουμε ότι τα στοιχεία που συνδέονται με το πρασίνισμα και με το νότο όριο είναι στοιχεία κλειδιά και για την αξιοπιστία της ΚΑΠ. Και πρόκειται για στοιχεία που θα πρέπει να βρίσκονται και πάλι να ξαναβρεθούν στη μεταρρύθμιση. Τώρα, λεπτομέρειες για το πώς θα το εφαρμόσουμε αυτά θα, θα παρουσιάσουμε στην πρόταση. Σημειώσαμε την πρόταση του Κοινοβουλίου και βέβαια θα επανέλθουμε με μια νομοθετική πρόταση που θα συζητήσουμε. Euh, Ο κύριος Βοητσεχόφσκι είπε ότι απογοητεύτηκε γιατί το 2004-2005 είχαμε αποθέματα, είχαμε πλεονάσματα ενώ τώρα τα κράτη-μέλη ζητούν ε, περικοπές στον προϋπολογισμό, μειωμένο γεωργικό προϋπολογισμό. Όντως, τα κράτη-μέλη ε, θα διαδραματίσουν σημαντικό ρόλο στις μελλοντικέ συζητήσει. Και η τελική συμφωνία θα περιλαμβάνει και τη θέση των κρατών μελών, αλλά όπως σας είπα και η Ευρωπαϊκή Επιτροπή σχεδίασε έναν προπολογισμό που είναι με φιλόδοξος αλλά ταυτόχρονα είναι και ρεαλιστικός, λαμβάνοντα υπόψη την ε, παρούσα οικονομική κατάσταση που δεν είναι ίδια με αυτή που είχαμε το 2004-2003 ή νωρίτερα. Χρειάστηκε και από αυτή την άποψη να προσαρμόσουμε τι ε, δημοσιονομικέ μα προτάσει στη σημερινή συγκύρια και πραγματικότητα. Και από αυτή την άποψη η ΚΑΠ εξακολουθεί να είναι η πρωταρχική προτεραιότητα του κοινοτικού προϋπολογισμού με βάση την πρόταση Ευρωπαϊκή Επιτροπή. Αυτό με το ξεχνάτε. Και αν τα κράτη-μέλη και το Κοινοβούλιο θεωρήσουν ότι θα πρέπει να αυξηθούν τα κονδύλια της ΚΑΠ, ότι θα πρέπει να αυξηθεί ο κοινοτικό προϋπολογισμός, εδώ είμαστε και θα το ξανασυζητήσουμε. Για τις άμεσες πληρωμές και την εξισορρόπηση, εξίσωση σας ε, εξήγησα ότι προσπαθήσαμε να βρούμε μια ισορροπία μεταξύ των συνολικών ποσών των διαφόρων κρατών μελών και με αυτή τη βάση να καταθέσουμε στη συνέχεια μέθοδο υπολογισμού για την κατανομή. Αλλά αυτό θα ακολουθήσει με τις νομοθετικές προτάσεις. Κυρία Πατραονέρες, ρωτήσατε πώς θα γίνει πιο δίκαιη η ΚΑΠ και για το πρόγραμμα ΠΟΖΕΙ με την πρόταση που έχουμε δεν νομίζω ότι θα υπάρξει αρνητικός αντίκτυπος στο πρόγραμμα ΠΟΖΕΙ. Δεν προβλέπεται ιδιαίτερη μείωση για το πρόγραμμα ΠΟΖΕΙ. Το ΠΟΖΕΙ διαφυλάσσει τη θέση που έχει σήμερα στην κυνηγιορική πολιτική. Τώρα πώς θα γίνει πιο δίκαιη η ΚΑΠ με το συνολικό ποσό και με τη μέθοδο υπολογισμού που θα προτείνουμε και που θα συζητήσουμε όλοι μαζί, ελπίζω ότι θα αποκαταστήσουμε μια μεγαλύτερη ισότητα και δικαιοσύνη στην ΚΑΠ. Σε ό,τι αφορά τις απόκεντρες περιοχές, όπως σας είπα, δεν έχει προβλεφθεί ή δεν προβλέπεται από τις προτάσεις μας αρνητική επίπτωση στις ε, απόκεντρες περιοχές, το προτείνεται μείωση των κονδύλιων. Κύριε Καλνιέτε, σας εξήγησα το πρότυπο και με βάση αυτό το πρότυπο θα υποβάλουμε τον Οκτώβριο διεξοδικότερες προτάσεις. Κύριε Λαβία, δεν είναι 8 δις, είναι 2,8 ε, δισεκατομμύρια για το Ταμείο Παγκοσμιοποίησης. Δεν είναι 8 δισεκατομμύρια. 9 είναι τα δισεκατομμύρια που ε, αφορούν το, τη σταδιακή εισαγωγή των κρατών μελών. Αλλά αυτό που αφαιρέσαμε από τη δημοσιονομική γραμμή 2, από το κεφάλαιο 2, το κατανείμαμε σε άλλες δημοσιονομικές γραμμές για να χρηματοδοτήσουμε αυτή τη σταδιακή εισαγωγή. Για τους απόρους. Έφυγε ο κύριος Παπαστάνκος, αλλά για τους απόρους η νομική βάση δεν έχει αλλάξει. Είναι αυτή που είχε προτείνει η Ευρωπαϊκή Επιτροπή. Τώρα, αν θα υπάρξει χρηματοδότηση από τα κράτη-μέλη, θα εξαρτηθεί αυτό από, τα, την έκβαση των συζητήσεων για την έγκριση των νομοθετικών προτάσεων της Ευρωπαϊκής Επιτροπής. Σε ό,τι αφορά τι λεπτομέρειε ευελιξία μεταξύ πρώτου και δεύτερου πυλώνα. Η ευελιξία αυτή, η ελαστικότητα αυτή ισχύει μόνο για την υιοθέτηση του νομοθετικού πακέτου. Δεν πρόκειται να παραμείνει ξέφραγο απέλη ή ε, απόλυτη διακριτική ευχαίρεια για τα κράτη-μέλη που θα κάνουν ό,τι θέλουν. Ε, έχει συγκεκριμένη διάρκεια το νομοθετικό πακέτο και μετά θα γίνουν κάποιες προσαρμογές από το Συμβούλιο και το Κοινοβούλιο, αλλά εξασφαλίζοντας η ισορροπημένη σχέση μεταξύ πρώτου και δεύτερου πυλώνα. Αυτό το θέμα με ενδιαφέρει ιδιαίτερα το πρόγραμμα έρευνας και ανάπτυξης. Όντως θα είναι πανευρωπαϊκό με πλήρως κοινοτική χρηματοδότηση, 100% από τον κοινοτικό προϋπολογισμό και στην ανακοίνωση που θα σας υποβάλουμε και στην ομοθετική πρόταση που θα καταθέσουμε με τις λεπτομέρειες πριν το 2013 θα συμπληρώσουμε το πλαίσιο για τη χρήση αυτού του προγράμματος. Επαναλαμβάνω θα είναι ευρωπαϊκό το πρόγραμμα και σα διαβεβαίω κύριε Μποβέ ότι θα εξασφαλίζει την υλοποίηση των προτεραιοτήτων τη ΚΑΠ. Τα 5,1 δις δηλαδή θα χρηματοδοτήσουν τις προτεραιότητες που έχουμε για την έρευνα, καινοτομία, ανάπτυξη και τη σχέση ε, γεωργίας ε, και έρευνα στην πράξη. Αυτές οι προτεραιότητες ε, καθορίζονται για την κοινή γεωργική πολιτική και αυτές θα εξυπηρετηθούν από το πρόγραμμα. Σε ό,τι αφορά τα ποσά του 2014 σε σχέση με το 2013 νομίζω ότι είναι πρόωρο να κάνουμε τέτοιε προβλέψει, θα εξαρτηθεί από τι διαπραγματεύσει για το νομοθετικό πακέτο και τη μεταρρύθμιση τη ΚΑΠ. Και είναι λογικό, γιατί δεν έχουμε τις, το πολιτέ δημοσιονομικό πλαίσιο που καθορίζει το επίπεδο πληρωμών για τον, για τον Α θα εξαρτηθεί από το μοντέλο κατανομής των άμεσων πληρωμών από τα κράτη-μέλη στα πλαίσια του πρώτου πυλώνα και θα εξαρτηθεί και από την τελική συμφωνία για τη μεταρρύθμιση της ΚΑΠ. Ο κύριος Σεκέρσκι είπε ότι το πάγωμα του γεωρικού προϋπολογισμού είναι αποτυχία ήττα γιατί περιμέναμε αύξηση του προϋπολογισμού. Το Κοινοβούλιο ζήτησε πάγωμα, διατήρηση του προϋπολογισμού και τώρα έχουμε επιτάπητος τις προτάσεις Ευρωπαϊκής Επιτροπής που ακριβώς ε, δέχονται, στερνίζονται την πρόταση του Κοινοβουλίου για πάγωμα. Τώρα για τις αγροτικές ζώνες, για την Ήπεθρο, ε, περιμένετε τις νομοθετικές προτάσεις και για τα μέτρα αγορά, τις μικρές εκμεταλλεύσεις, τις μικρές γεωργικές εκμεταλλεύσεις. Όλα αυτά τα σημεία θα περιληφθούν στις νομοθετικέ προτάσεις. Κυρία Κέστιγκερ, για τι λιγότερο ανεπτυγμένε περιοχές δεν μετατοπίζονται στον πρώτο πυλώνα. Το είπα, παραμένουν στο δεύτερο πυλώνα. Ένα συμπλήρωμα ε, παρέχει ο πρώτος πυλώνας, αλλά αυτό το είπα προηγουμένως για το Ταμείο Παγκοσμιοποίησης και το Ταμείο για την Κρίση. Σε ό,τι αφορά το Ταμείο για την Κρίση ε, θα ενεργοποιηθεί ε, άμεσα με τον ίδιο ρυθμό, ταχύ ρυθμό που κινητοποιούμε και τα μέτρα της αγοράς. Ίδια κατεπήγουσα διαδικασία. Όταν υπάρχει ένα πρόβλημα στις αγορές εξαιτία μιας υγειονομικής ή άλλης κρίσης, κινητοποιούμε το κονδύλιο αυτό αμέσω με πολύ συνεπτικέ διαδικασίε, όπω γίνεται και με τα μέτρα αγορά. Το ίδιο θα για το Ταμείο Κρίση. Σε ό,τι αφορά το Ταμείο Συνοχή, και γι' αυτό θα καταθέσουμε πιο λεπτομεριακέ προτάσει στη συνέχεια. Και ο κύριος Νταντά, από ό,τι κατάλαβα, έφυγε μίλησε για το Ταμείο Συνοχής και τη διάρθρωση με το Ταμείο Συνοχής. Θα το δούμε παράλληλα με τις δημοσιονομικές προοπτικέ και τη μεταρρύθμιση των δύο πολιτικών, της ΚΑΠ και τη πολιτικής συνοχής. Σε δημοσιονομικό επίπεδο θα υπάρξει μια συνάρτηση και να, για να εξασφαλιστεί και μια ισορροπία μεταξύ της κατανομή των κονδυλίων. Κύριε Καρινόφσκι, εγώ είμαι υπέρ μια πιο ισορροπημένη και δίκαιη κατανομή. Αυτό φυσικά μέσα στα όρια, τα δημοσιονομικά όρια που ξεπερνούν και την ΚΑΠ, γιατί για να έχουμε ένα, ένα κοινοτικό προπολογισμό θα πρέπει να εξασφαλίσουμε την ισορροπία μεταξύ των κρατών μελών και δεσμευόμαστε από κάποια όρια. Και επειδή η μεταρρύθμιση της ΚΑΠ συμπίπτει με τη συζήτηση για τη μεταρρύθμιση του προπολογισμού, θα πρέπει να συντονιστούμε και στην πορεία να βρίσκουμε την εξισορρόπηση. Τώρα, αν θα εγκρίνουν τα κράτη-μέλη τον προπολογισμό. Κύριε Γιάννη, μιλήσατε για σύγκριση 2013-2014. Ας περιμένουμε όμως την έγκριση του νομοθετικού πακέτου και μετά θα κάνουμε προβλέψεις. Τώρα, αν τα κράτη-μέλη εγκρίνουν το προπολογισμό ή όχι. Και η κυρία Ρέινερς είπε από πού θα γίνουν οι περικοπές. Κατά τη γνώμη αυτό είναι το ελάχιστο απολύτως απαραίτητο για την ΚΑΠ η πρόταση που κάναμε για την ΚΑΠ δεν έγινε με την ιδέα ότι στη συνέχεια θα περικοπεί ο προπολογισμό. Αν τώρα τα κράτη-μέλη, του Κοινοβούλιο ε, αποφασίσουν περικοπές θα πρέπει να αναλάβουν και την πολιτική ευθύνη για την Ευρωπαϊκή Επιτροπή. Αυτό είναι ο απολύτω απαραίτητο προπολογισμό για την ΚΑΠ, για να γίνουν επενδύσει, για να εξασφαλιστεί ο στόχο τη επισητιστική ασφάλεια. Εγώ δεν βλέπω άλλα περιθώρια για περαιτέρω μείωση του προπολογισμού Τη ΚΑΠ σε σχέση με τον υπόλοιπο προπολογισμό. Δεν έγινε η πρόταση αυτή έχοντα κατά νου ένα περιθώριο μείωση. Νομίζω ότι είναι το απολύτω απαραίτητο, το ελάχιστο όριο για την ΚΑΠ. Τώρα, ποια θα είναι η θέση των κρατών μελών, αυτό δεν μπορώ να το ξέρω εγώ από τώρα, θα δούμε. Sí, euh, je le fais. Chiediamo scusa <laughs> Grazie. Grazie commissario. Ευχαριστώ κύριε Επίτροπε. Νομίζω ότι ήταν εξαντλητικές ε, οι απαντήσεις ε, σε όλους τους παρεμβαίνοντες. Ε, λοιπόν, θα κλείσουμε εδώ τη συνεδρίασή μας. Θα υπενθυμίσω στους συντονιστές αύριο στην αρχή της συνεδρίασης θα κάνουμε τη συνεδρίαση, συγγνώμη, στο τέλος της συνεδρίας θα κάνουμε τη συνεδρία των συντονιστών. Ευχαριστώ. Λήξη της συνεδρίασης.